Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση για διήμερη συνεδρίαση που πιθανότατα είναι η τελευταία της θητείας εκτός από κάποια έκτακτη σύνοδο της ε, Επιτροπής για κάποιο κατεπήγον θέμα θα μπορούσε να υπάρξει και αυτό εξηγεί και το, τη βαριφορτωμένη μερίσια διάταξη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τις εργασίες, αν και αρκετοί, μάλλον πολλοί συνάδελφοι απουσιάζουν και αν έχετε την καλοσύνη θέλω να ρωτήσω αν έχετε αντιρρήσεις όσον αφορά τα πρακτικά. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις πρώτα απ' όλα όσον αφορά την ημερήσια διάταξη. Ο κύριος Στέρξ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταφέραμε να πετύχουμε ένα συμβιβασμό για το πακέτο Gross Take επιτρέψτε μου να το αποκαλέσω έτσι, Ωραία, ναι. Πετύχαμε λοιπόν συμβιβασμό για το πακέτο Gross Tikau. Και θα ήθελα να πούμε δύο λόγια στην ημερήσια διάταξη για το θέμα αυτό. Έχω και μία ερώτηση, έχω και μία παρατήρηση σχετικά με αυτό. Καταρχάς να ρωτήσω, ο προσωρινός κατάλογος ψηφοφορίας που είδα αναφέρει ότι αν εγκριθεί το πακέτο δεν θα ε, ψηφιστούν οι μεμονωμένες τροπολογίες. Εγώ θα ήθελα να ψηφιστούν οι μεμονωμένες τροπολογίες και από ό,τι ξέρω είναι δυνατόν και θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσετε αυτό. Δεύτερο σημείο που ήθελα να αναφέρω είναι παρατήρηση. Δεν συμφωνούμε με την ε, συμβαστική πρόταση γιατί θεωρούμε ότι στοιχεία ουσίας απουσιάζουν από το συμβαστικό αυτό σχέδιο. Αυτά λοιπόν, Πρόεδρε. Θα ήθελα λοιπόν να σα ρωτήσω αν ισχύουν και όσα σας ε, ρώτησα για την αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν άλλα θέματα που αφορούν την ημερήσια διάταξη. Έχετε κάποιε αντιρρήσεις. Έχετε κάποια, κάποιο ιδιαίτερο έτοιμο σε αυτή τη ημερήσια διάταξη. Ο κ. Σίμψον. Έχω πρόβλημα να σχολιάσω την ημερήσια διάταξη όταν δεν την έχω μπροστά μου. Ε, ε. Λοιπόν, εκ δεν έχει διανεμηθεί ούτε εκθέσει ούτε... Όχι, όχι, Λίκο Σίμψον. Περιμένουμε λοιπόν. Περιμένουμε 30 δευτερόλεπτα να μοιραστούν τα έγγραφα. Τι γίνεται με του κλητήρε, όλα πάνε καλά, τι γίνεται με τη διανομή των εγγράφων. Θα ζητήσουμε από του κλητήρε να διανύμουν επιτραπέζι τα έγγραφα. Λείπουν εκθέσει. λείπουν έγγραφα. On attend 30... Περιμένουμε 30 δευτερόλεπτα. 10 λεπτά, πολλά είναι. Καλώς. Να ζητήσω από τους βοηθούς να πάνε να βρουν τα έγγραφα για τους βουλευτές. Για να ελαφρύνουμε κάπως τους ε, κλητήρες. Μόλις κατέθεσαν τα εγγράφα και γι' αυτό υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Κύριε Σίμψον, υποθέτω ότι η μερίσια διάταξη δεν έχει, δεν κρύβει μυστικά για σας, παρόλο, που δεν είναι μπροστά σας στο τραπέζι. Λοιπόν, πάμε στο θέμα του κυρίου Στέρξ. Απλά περιμένουμε να καθίσει ξανά ο κύριος Στέρξ. Et puis il Για Στέρξ. Κύριε Στέρξ, ήρθατε. Γκροστικάο, έκθεση Γκροστικάο. Θέλετε λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, να πείτε ότι έχετε δίλημα. Η ομάδα σας δεν είναι υπέρ της συμβαστικής λύσεως. Περί αυτού πρόκειται. Όχι. Α. Εξηγήστε μου, ποιο είναι το ερώτημά σας. Πρόεδρε, στον προσωρινό κατάλογο ψηφοφορίας που έλαβα αναφέρεται ότι η δεύτερη ομάδα τροπολογιών δεν είναι συμβατές με τη συμφωνία της δεύτερης ανάγνωσης. Στα αγγλικά το γράφει. Μπορώ να έχω ένα κείμενο μη μετάφραση παρακαλώ. Το ερώτημα που έχω εγώ να θέσω είναι το εξής. Αυτό τι σημαίνει το not comparable, δεν είναι συμβατό ότι δεν θα το ψηφίσουμε ή ότι αφότου θα συμφωνήσουμε και θα έχουμε ψηφίσει το συμβιβασμό, θα ψηφίσουμε και τις μεμονωμένες τροπολογίες. Αυτό θέλω να μου πείτε, γιατί καλώς και ο συμβιβασμός, αλλά κάποια στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στον συμβιβασμό θέλουμε να τα ψηφίσουμε, γιατί μεταξύ άλλων είναι και κάποιες τροπολογίες που έχω καταβάλει κι εγώ. Κοιτάξτε, μπορούμε να ψηφίσουμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε και επί των δύο την ίδια ισορροπία ψήφων, γιατί δεν συμφιλειώνονται. Δεν υπάρχει όμως αντίθεση πάνω στον κανονισμό. Μπορούμε να ψηφίσουμε τις ε, τροπολογίες σας. Υπάρχουν παρατηρήσεις από αυτού. Καλώς, αν δεν υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις, θα συνεχίσουμε την πορεία. Ακολουθώντας τη μερίσια διάταξή μας στο δεύτερο σημείο, είναι η έγκριση των πρακτικών Υπάρχουν παρατηρήσεις όσον αφορά τα πρακτικά των προηγουμένων συνεδριάσεων. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρούνται εγκεκριμένα τα πρακτικά. Δίνουμε το λόγο στον κύριο Αλμπερτίνη για τα δικαίωμα των επιβατών όσον αφορά τις οδικές μεταφορές. Ο κύριος Αλμπερτίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε μια σύντομη εισαγωγή να κάνω, γενική εισαγωγή όσον αφορά τους στόχους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν για την σύνταξη αυτού του κανονισμού και κάποιες σύντομες παρατηρήσεις όσον αφορά τις υποβληθήσεις τροπολογίες και τις συμβαστικές τροπολογίες που ετοιμάσαμε. Όπως με θύμισε όταν αντιμετωπίσαμε το όλο ζήτημα σφαιρικά και γενικά, αντιμετωπίσαμε τον ορισμό, τον καθορισμό των δικαιωμάτων των επιβατών όσον αφορά τις ε, μεταφορές, ελεοφορία και πούλμαν. Θέλουμε να πετύχουμε ισότιμες συνθήκες όσον αφορά αυτόν το τομέα, δηλαδή ίσα δικαιώματα για όλους, level playing field, ούτω ώστε οι διάφοροι τρόποι μεταφορών να μπορούν υπό τις ίδιες συνθήκες να ανταγωνίζονται οι μεν τους δε και να έχουν τι ίδιε δυνατότητε να πετύχουν. Ταυτόχρονα θα πρέπει οι επιβάτες να έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο που επέλεξαν και όπως επανειλημμένα επενθυμίστηκε, αν υπάρχει και πρόβλημα, αν κάποιος επιβάτης έχει πρόβλημα, έχει μειωμένη κινητικότητα. Έπρεπε να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τα χαρακτηριστικά κάθε τρόπου μεταφοράς, που προφανώς έχει διαφορές ο ένας τρόπος μεταφοράς από τον άλλο. Ένα παράδειγμα όσον αφορά την διαχείριση των καθυστερήσεων. Είναι διαφορετικό να εξεταστούν αν το μέσο κινείται επί ανοιχτού τρόπου και ελαστικών, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν κυκλοφοριακές συμφορήσεις ή κάτι άλλο, διαφορετικά αν υπάρχει, επί, ε, κινείται επί τροχιών, οπότε η διαχείριση του δικτύου και η οργάνωση των μεταφορών ε, ρυθμίζεται από έναν ενιαίο φορέα. Πρέπει να βρεθεί ισορροπία μεταξύ ενοποίησεως των δικαιωμάτων των επιβατών και να λάβουμε υπόψη και τις ιδιαιτερότητες των μεταφορικών συστημάτων επί τροχών των οδικών μεταφορικών μέσων. Να λάβουμε υπόψη τα μικρά και μεσαία οχήματα σε μέγεθος που είναι πιο εύκολο να οργανηθούν αλλά μπορεί να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες δυσκολίες σε σχέση με άλλους τρόπους μεταφορών. Άρα χρειάζεται κάλυψη των ιδιαιτεροτήτων των μεταφορικών μέσων. Χρειάζεται ανάλυση της νομοθεσίας. Και έπρεπε ε, να δούμε τι γίνεται και στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης που περνάμε. Επ' αυτής της βάσης κινηθήκαμε να μπω στην ουσία της επιχειρηματολογίας. Σχετικά με τις προτάσεις που έγιναν από του συναδέλφους επί υπέβαλαν τροπολογίες. Και με τους κοιόδης εισηγητές είχαμε εντατικό διάλογο αυτές τις μέρες για να συνεννοηθούμε και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες. Οι περισσότερες ήταν λογικές και θεωρώ ότι λήφθησαν σοβαρά υπόψη στην πρόταση, στον κατάλογο ψηφοφορίας που προτείνουμε και ευχαριστώ ιδιαίτερα στους κοιόδης εισηγητές που συμμερίστηκαν τις προσπάθειες που καταβάλαμε όλοι μαζί για να λάβουμε υπόψη τις αντιφατικές καμιά φορά πτυχές που έπρεπε όμως να συγκεραστούν ε, για τους λόγους που προανέφερα. Πιο αναλυτικά. Στις τροπολογίες. Θα αναφερθώ σε κάποιες τροπολογίες μόνο. Το περισσότερο χρόνο θα τον αφιερώσω στα σχόλια τα δικά σας να ακουστούν. Και προς το τέλος θα δώσω κάποιες εξηγήσεις όσον αφορά τις προτάσεις μου για την ψηφοφορία και θα εκφράσω και κάποιες σκέψεις μου αφού ακούσω τη δική σας επιχειρηματολογία. Για την τροπολογία 54, συναδέλφου Evans. Εκεί αναφέρεται ο ορισμός της προσβάσιμης μορφής μεταφοράς. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συμφωνώ με τον κύριο Evans καταλήξαμε σε λιγότερο περιοριστικό ορισμό όσον αφορά της προσβάσιμης μορφής μεταφοράς. Διότι αυτός είναι ένας όρος που περιλαμβάνεται σε διάφορα νομοθετήματα. Πιο γενική διατύπωση κάνει πιο εύκολο τον, εύκολη την ανάγνωση του κανονισμού και καλύτερη την εφαρμογή του. Λοιπόν, η τροπολογία 54 είναι προφορική τροπολογία. Όσον αφορά τη συμβαστική τροπολογία που αφορά το άρθρο 8 παράγραφος 6 για την μη δυνατότητα επιστροφής των παρακαταβολών, λάβαμε υπόψη τις διάφορες παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ευρωπαίων Ασφαλιστών και τις απόψεις διαφόρων συναδέλφων. και εξετάσαμε την περίπτωση κατά την οποία το τελικό ποσό το οφειλόμενο από, την, από τη στιγμή που ο φορέας αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του είναι χαμηλότερο από την προκαταβολή. Η προκαταβολή θεωρείται ότι το ανώτατο όριο είναι 21.000 ευρώ. Θα πρέπει να επιστραφεί η διαφορά λοιπόν στο φορέα. Για το άρθρο 19 έχουμε προφορική τροπολογία Απλώς γλωσσική διευκρίνηση είναι αυτή. Και στην προφορική τροπολογία για το 130 και εκεί έχουμε γλωσσική τροπολογία για τις διεκδικήσεις, για τις αμφισβητήσεις, για διάφορα αιτήματα θα πρέπει να ασχολείται με αυτά ένας οργανισμός που θα συνδέεται με τους μεταφορικούς φορείς. Δεν θα είναι ανεξάρτητος φορέας. Αυτή είναι η πρόταση του συναδέλφου Evans. Για την προφορική τροπολογία 139, πάντα του συναδέλφου Evans, ίσως εδώ είναι το μόνο κείμενο επί το οποίου ήθελα να εκφράσω αρνητική άποψη. Όχι τόσο διότι διαφωνώ επί της ουσίας των όσων προτείνονται, αλλά θεώρησα ότι η διατύπωση του κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αρκετά σαφής όταν λέει τεχνικές για, να, για την μεταφορά των ζώων που είναι αναγνωρισμένα που παρέχουν βοήθεια στον ιδιοκτήτη τους. Θεωρώ ότι η πρόταση του κυρίου Evans είναι πλεονασμός. Οπότε γι' αυτό συζητητής είμαι αρνητικό όσον αφορά την τροπολογία. Όπως είπα, προτιμώ να μην υπησέλθω σε ανάλυση τώρα στην εισαγωγή μου. Θέλω να ακούσω τι παρατηρήσει σα. Και στην ολοκλήρωση της συζητήσεως ε, θα αναφερθώ εκτενέστερα και θα δώσω κάποιες εξηγήσεις αφού ακούσω τις προτάσεις των συναδέλφων. Σας ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Ο κύριος Σίμψον ζήτησε το λόγο εκ μέρους των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Έχω ένα μικρό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν το αντιμετωπίζουν και άλλοι συνάδελφοι. Έχουμε τις τροπολογίες 1.36 αλλά άλλες τροπολογίες δεν βλέπω για την έκθεση Αλμπερτίνη. Είναι σαν να πυροβολεί κανεί τα τυφλά. Πού είναι οι άλλες τροπολογίες, τι συνέβη. Εκτός α, κι αν είναι παράληψη από την... αγγλική, από, το αγγλικό, από τον αγγλικό φάκελο. Λυπούμε κύριε Αλμπερτίνη, αλλά εγώ στο χαρτοφυλάκιο όμως έχω μόνο τις τροπολογίες 1 με 36. Τι να πω για τις άλλες. Άλλωστε αντικαθιστώ τον κύριο, τον κύριο Evans που προεδρεύει στην αντιπροσωπεία του αυτή τη στιγμή. Και αναφερθήκατε στο θέμα των σκυλιών που είναι οδηγοί για τυφλούς. Και σίγουρα εκεί θέλουμε να είμαστε συνεπείς σε σχέση με αυτά που συμφωνήσαμε στην αεροπορία για σκυλιά οδηγούς. Σίγουρα φυσικά μας ενδιαφέρει το θέμα της υγείας, αλλά από τη δική μου πείρα ε, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα με τα σκυλιά, γιατί μερικές φορές είναι πιο, ε, έχουν καλύτερο αίμα από ότι ορισμένοι άνθρωποι. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες 45 και 47 αποκλείουν τις περιφερειακές μεταφορές από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Το πρόβλημα με τη διάταξη αυτή είναι ότι οι περιφέρειες μπορεί να είναι μεγάλων διαστάσεων. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από την πατρίδα μου που γνωρίζω καλύτερα. Ένα ε, ταξίδι από το Κάρντεφ στη νότια Ουαλία προς τη βόρεια Ουαλία διαρκεί 8 ώρες με πούλμαν. Ενώ αντίθετα για να πάμε από τις Βρυξέλλες στο Λουξεμβούργο χρειαζόμαστε 2 ώρες. Τι λέτε τώρα, να κρατήσουμε το 2 ώρο ταξίδι Βρυξέλλες-Λουξεμβούργο αλλά να αποκλείσουμε το εσωτερικό ουαλικό ταξίδι που διαρκεί 8 ώρες μόνο και μόνο επειδή 8 ώρες ε, είναι η διαδρομή στην ίδια περιφέρεια. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Καλύτερα να υιοθετήσουμε έναν ε, διαφορετικό ορισμό και όχι στενό γεωγραφικό ορισμό. Δεν νομίζω. με τις 45 και 47 να μην έχουμε προβλήματα. Σε ό,τι αφορά ε, τις ε, εξαιρέσεις άλλων συναδέλφων ε, που αντιπαραγωγικά φαίνεται να αποκλείουν, να ξερούν ολόκληρους λαούς αλλά δεν σχόλιο για αυτές. Ένα άλλο πρόβλημα με την τροπολογία 32, την τροπολογία Σόμερ. Ο κύριος ε, ε, παρέβλεψε το γεγονός ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διευκρίνηση γιατί το barrier free είναι κάπως αμφίσιμο στα αγγλικά. Τι είδου ε, barrier free εννοείται, γιατί υπάρχουν και άλλοι φραγμοί. Όταν λέμε χωρίς φραγμούς, τι φραγμούς καλύπτουμε εδώ. Υπάρχουν και νομικοί φραγμοί. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Είναι οι πύλες, είναι ένας ε, απτός υλικός φραγμός ή μιλούμε για μεταφορικούς φραγμούς, νομικούς για παράδειγμα ή άλλους. Το παρέβλεψε αυτό ο κύριος Evans. Ευχαριστώ πάντως ε, τον εισηγητή εκ μέρους του κυρίου Evans για τη συνεργασία του, αλλά στους τρεις τομείς ε, που ανέφερα θέλουμε κάποιες διευκρινήσεις. Μόλις τώρα έλαβα για τις υπόλοιπες τροπολογίες, θα τις μελετήσω διεξοδικά. Καλώς. Λυπούμε, λυπούμε για αυτά τα μικροπροβλήματα σε ό,τι αφορά τη διανομή των εγγράφων. Στην ε, γαλλική ημερήσια διάταξη έκθεση Αλμπερτίνη φέρνει τον αριθμό 4. Ελπίζω να ισχύει και για τους άλλους συναδέλφους. Ίσως αυτό δημιούργησε κάποιες ε, περιπλοκές. Το λόγο έχει ο κύριος Στέρξ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και κατανοώ φυσικά απόλυτα όλους όσοι βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση και πρέπει να φροντίσουν να πάρουμε τα απαραίτητα έγγραφα και όταν τελευταία στιγμή τους τα φέρνουν τα έγγραφα Προφανώς και είναι δύσκολο να φροντίσουν εγκαίρως να έχουμε τα έγγραφα μπροστά μας. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή εξ ονόματος του συναδέλφου Φεράρη. Ένα στοιχείο το οποίο έθιξε ο Μπράιαν Σίμψον θα ήθελα να αναφέρω και εγώ, οι τροπολογίες για το άρθρο 2, παράγραφος 2. Θα υποστηρίξουμε την ε, τροπολογία MSTK, γιατί νομίζουμε ότι το χρειαζόμαστε αυτό ως θέση διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο προκειμένου οι περιφερειακές ε, μεταφορές να μην εξαιρεθούν εκ των προτέρων και νομίζω ότι θα πρέπει άλλωστε και στο θέμα των σιδηροδρόμων ε, το διαπραγματευτήκαμε αυτό έντονα με το Συμβούλιο άρα ούτε εδώ δεν πρέπει να το αφήσουμε βρισκόμαστε στην πρώτη ανάγνωση Νομίζω ότι, ότι για τις αστικές μεταφορές το Κοινοβούλιο μπορεί να πει ότι ωραία αυτή είναι ιδιαίτερη περίπτωση, αλλά για τις περιφερειακές ε, μεταφορές θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό αναπεριφέρεια, ανακράτος μέλος, να ρωτήσουμε τα κράτη-μέλη το τι θεωρείται εξαίρεση και τι όχι και γιατί. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ πέρα θέλει λίγο χτένισμα η τροπολογία. Γι' αυτό λοιπόν θα υπερψηφίζαμε την 46 και θα καταψηφίσουμε την 45 ε, και την 47. Νομίζω ότι έτσι ως Κοινοβούλιο θα έχουμε περιθώριο ελιγμού για τα θέματα αυτά και κατά τα άλλα θα ακολουθήσουμε τη γραμμή την οποία σύστησε ο εισηγητής. Σε αδρές γραμμές, ε, σε κάποιες λεπτομέρειες έχουμε λίγο κάποιες διαφορετικές απόψεις, αλλά φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε να τα επιλύσουμε τα θέματα αυτά και πριν την ψηφοφορία στην Ολομέλη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στέρξ. Η κυρία Λίχτεμπέργκερ για τους πράσινους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή. Θα συμφωνήσω ότι οι εξαιρέσει για τις περιφέρειες είναι κάπως υπερβολικά ευρείες, γιατί μετά θα παραμείνουν μόνο οι μεταφορές ε, μεγάλων αποστάσεων με τα πούλμαν και τίποτα άλλο. Έχουμε μεγάλες αποστάσεις. Δεν είναι δυνατόν να τα αφήσουμε αυτό έτσι. Αν πρόκειται για τοπικές συνδέσεις, για αστικές συνδέσεις, αν θέλετε μεταφορές, εντάξει, να το συζητήσουμε. Γιατί εδώ δεν ισχύουν και οι σχετικές ρυθμίσεις για τις καθυστερήσεις. Αλλά το να κάνουμε τώρα γενικές εξαιρέσεις για το σύνολο των περιφερειακών μεταφορών, αυτό πραγματικά παραπάει, θεωρώ. Και για παράδειγμα να δούμε τι γίνεται με την γειτονική μας περιφέρεια, την Βαβαρία. Είναι τεράστιες έκτασεις. Αν εξαιρέσουμε όλες τις περιφερειακές μεταφορές, έτσι ε, θα απομείνει μόνο τα Eurolines, τα Pullman αυτά, ξέρετε, τα αντιευρωπαϊκά. Και αν συγκρίνουμε αυτό με τη σύνδεση μεταξύ Ρήγας και Βιλνίους, με μια μεταφορά στην Βαβαρία, που είναι πολύ πιο μεγάλη, αλλά δεν είναι διεθνή μεταφορά. Αυτή είναι η δυσκολία. Τι θα κάνουν δηλαδή οι χώρες που δεν έχουν ορίσει τόσο τις περιφέρειες αυτές. Τι είναι η περιφέρεια. Η Γαλλία, για παράδειγμα, έχει πολύ μικρές περιφέρειες. Και σε αυτή την περίπτωση μπορεί και πάλι να είναι υπερβολικά άκαμπτη αυτή η εξαίρεση. Νομίζω λοιπόν ότι η επιλογή των περιφερειών δεν είναι σωστή. Κατά δεύτερον, δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Ξέρω ότι βρισκόμαστε σε μια πρώτη φάση, αλλά θα ήθελα λίγο παραπάνω φιλοδοξία. Γιατί γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο πάντα παρεμβαίνει υπερβολικά σε αυτά τα θέματα. Γιατί η τοπική φορείς μεταφορών είναι αυτή που είναι στο επίκεντρο της προσοχής και όχι οι άνθρωποι, τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να μας οθήσει να είμαστε λίγο πιο αυστηροί τουλάχιστον στην πρώτη ανάγνωση, γιατί η δεν θα έχουμε καθόλου περιθώριο πραγματεύσεων. Τρίτον, για το barrier free, χωρίς ε, σύνορα, από τα γερμανικά μάλλον, πρόκειται για τη νέα επιλογή διατύπωσης των ε, ενώσεων ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα που δεν ε, αναφέρονται πλέον στο άτομο και στην αναπηρία του, στην ανικανότητά του εισαγωγικά, αλλά αναφέρονται στα εμπόδια που υπάρχουν στον δρόμο. Να πω στον συνάδελφο Σίμψον ότι φυσικά υπάρχουν ε, και σωματικές, σωματικά εμπόδια, αλλά υπάρχουν και πρακτικά εμπόδια. Για παράδειγμα, ότι δεν μπορεί κανείς να ταξιδέψει επειδή το καροτσάκι του ζυγίζει υπερβολικά πολύ. Δεν ε, είναι τα αγγλικά η μητρική μου γλώσσα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα οι Βρετανοί συνάδελφοι να μας προτείνουν την ιδανική διατύπωση. Δεν ξέρω τι έχουν να προτείνουν και οι σχετικέ ενώσει. οι σύνδεσμοι, να δούμε τι γίνεται με τον όρο reduced mobility. σω είναι προτιμητέο. Αλλά χαίρομαι και θα ήθελα να συζητηθεί αυτή η διατύπωση. Γιατί σημαίνει αλλαγή νοτροπίας, ότι εμείς θα αφαιρέσουμε τα εμπόδια για τα άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες, όχι ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάποιο πρόβλημα και θα πρέπει να τους δώσουμε κάτι. Νομίζω ότι σημαίνει κάτι σημαντικό αυτή η αλλαγή διατύπωσης. Και ξέρω ότι οι ενώσει των ε, αναπήρων θέλουν να τονίζεται αυτή η διάσταση, όχι μόνο των όσων δεν μπορούν να κάνουν, αλλά των όσων μπορούν να κάνουν κιόλας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο συγκείμενο αυτό. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Λιχτεμπέργκερ. Ο κύριο Δεγκράντε Πασκουάλ. Ευχαριστώ. Καταρχήν, ένα διαδικαστικό. Θα μιλήσω συντάκτη ε, τροπολογία, όχι εκ μέρου του ΕΛΚ. Δεν ξέρω αν ε, ο πρώτο γύρο ερωτήσεων ε, θα γίνει από εκπροσώπου των πολιτικών ομάδων. Γιατί ζητώ το λόγο συντάκτη τροπολογία και όχι ω εκπρόσωπο τη ομάδα μου. Αν μου δίνετε το λόγο τώρα, καλώ, αλλιώ θα περιμένω. Καλώ, καλώ. Πείτε μα τη γνώμη σα. Οποιοδήποτε ευρωβουλευτής μπορεί να εκφέρει την προσωπική του γνώμη. Ακόμη και αν έχετε εισηγητή σκιώδη στην ομάδα σας. Ακόμη και αν δεν είχατε συντάξει τροπολογής. έχετε κάθε δικαίωμα να υποστηρίξετε ορισμένε από αυτές. Το, το γνώριζα κύριε Πρόεδρε, αλλά επειδή διαπίστωσα ότι μίλησαν πρώτα εκπρόσωποι των ομάδων, ε, νόμιζα ότι πρώτα θα ακούσουμε όλου του εκπροσώπου των ομάδων. Εν πάση περιπτώσει, μου δίνετε το λόγο, πολύ ωραία. Θα είμαι σύντομο. Ο εισηγητή τη ομάδα μα είναι ο κύριο Αλμπερτίνη. Το συγχαίρω γιατί πραγματικά το έργο του είναι αξιέπαινο. Και το εύχομαι καλή επιτυχία. Ελπίζω να συγκεντρώσει την απαραίτητη συνένεση για να λάβει και το πράσινο φως από την Επιτροπή. Μιλώ προσωπικά. Εκφέρω την προσωπική μου γνώμη και δεν δεσμεύει κανέναν άλλον εκτός από μένα. Η προσωπική μου γνώμη σχετίζεται με τη δική μου αντίληψη και δεν έχει καμία σχέση με τη θέση της ομάδας. Έχω καταρχήν μια γενική παρατήρηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχική της πρόταση ξέχασε ότι διάφοροι τρόποι μεταφοράς δεν είναι συγκρίσιμοι μεταξύ τους, δεν είναι ισοδύναμοι. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις ε, μεγάλες ε, ε, αερομεταφορικές εταιρείες ή τις εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών με τις εταιρείες οδικών μεταφορών οι επιχειρήσει ελευθερίου και πουλμαν είναι πολύ πιο μικρές και πιο απλή διαχείρισης και οργάνωσης. το και το πεδίο δραστηριοτήτων τους είναι το ίδιο. Δεν είναι θέμα εδαφικό ή περιφερειακό, οπότε το να ισχύουν τα ίδια μέτρα και σταθμά και για αυτές τις επιχειρήσεις, κατά τη γνώμη μου, είναι επικίνδυνο και άδικο. Αυτό το σκοπό της ε, διόρθωσης έχουν οι τροπολογίες μου. Ορισμένες βέβαια μπορεί να τις διαπραγματευτώ, αλλά θα ήθελα να εκφέρω τη γνώμη μου. Καταρχήν, στο άρθρο 2, παράγραφος 1, το πεδίο εφαρμογής προτιμώ να περιοριστούμε στις ε, εθνικές μεταφορές, στις διακρατικές μεταφορές, γιατί συνήθως τα λεωφορεία περιορίζονται στις εθνικές επικράτειες και έχουν και ιδιαιτερότητες αυτές οι μεταφορές. Θα πρέπει να γίνει σεβαστή λοιπόν η αρχή της επικουρικότητας. Δεν μπορούμε να τα ρυθμίζουμε όλα κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε, οι οδικές μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν περιορίζονται περισσότερο σε εθνικές παραδόσεις, την Πορτογαλική, την Ισπανική, την Βρετανική, ενώ άλλες χώρες δεν ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό, ενώ εμείς ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα. Άλλο θέμα, άρθρο 2, παράγραφος 2 εξαιρέσεις. Οι εξαιρέσεις που προτείνονται, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να περιλάβουν και τις ε, διαπεριφερειακές υπηρεσίες μεταφορών, για να μην δημιουργήσουμε διαφορετικά συστήματα ευθυνών για τις επιχειρήσεις. Για το άρθρο 3 τώρα, σημείο 12, περιλαμβάνεται στον ορισμό της καθυστέρησης ε, για να επιρρύπτεται στον μεταφορέα θα πρέπει αυτό να είναι ο υπέτειος της καθυστέρησης. Όπως ξέρετε όμως, στην πραγματικότητα και με τις ιδιαιτερότητες οδικής μεταφοράς, συνήθως υπάρχει συγχρονισμός με άλλα είδη μεταφοράς και πολύ συχνά η, με, καθυστέρηση δεν οφείλεται σε ένα μόνο τρόπο μεταφοράς. Δεν μπορούμε λοιπόν να ενοχοποιούμε μόνο τον οδικό μεταφορέα που είναι ο τελευταίος κρίκος αλυσίδας γιατί μπορεί η καθυστέρηση να οφείλεται σε προηγούμενη φάση σε ένα άλλο μέσο μεταφοράς. Είναι άδικο λοιπόν αυτό. Στο άρθρο 4, παράγραφος 2α νέο, προτείνεται το εισιτήριο να έχει το ελάχιστο περιεχόμενο ενημέρωσης ευθυνών του μεταφορέα. Σίγουρα μιλούμε για δικαιώματα των επιβατών, αλλά χρειαζόμαστε και κάποια αμοιβαιότητα. Θα πρέπει σίγουρα να γνωρίζει ο καταναλωτής ε, ελάχιστες πληροφορίες για το ποια είναι τα δικαιώματά του, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, αλλά αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, θα πρέπει κάτι αντίστοιχο να ισχύσει όπως ισχύει και για τις άλλες μεταφορές. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 8 παράγραφος 1, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και εδώ έχω μια γενική παρατήρηση. Τώρα το να ε, επιρρύπτουμε αυτεπάκελτα, αυτόματα στον οδικό μεταφορέα της ε, αποζημιώσεις, νομίζω είναι παράλογο. Φυσικά θα πρέπει να δούμε και το θέμα της επανάληψης ε, ορισμένων δράσεων των ασφαλιστικών εταιριών. Εγώ όταν ήμουν ενεργεία δικηγόρος είχα εμπειρία με τροχαία ατυχήματα. Το να ορίζουμε υπεύθυνο αυτόματα τον ε, μεταφορέα, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις αυτές ε, συνήθως είναι μικρές επιχειρήσεις, ε, δεν έχουν μεγάλη επιφάνεια, με μια τέτοια διάταξη θα τους αυξήσουμε υπερβολικά το άχθος. Δεν λέω ότι θα πρέπει να απαλλάσσονται από τις ευθύνες τους, αλλά θα πρέπει να δούμε και το θέμα της επανάληψης. Άρθρο 8 τώρα παράγραφος 2. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Και εδώ θέλουμε να περιορίσουμε την ε, επίληψη της ευθύνης αυτόματα από τον, ε, στον ε, οδικό μεταφορέα. Αυτό δεν σημαίνει θα πρέπει να υπάρξει κάποια παρέλκυση της διαδικασίας ή καθυστέρηση της αποζημίωσης, αλλά δεν μπορούμε άμεσα να επιβαρύνουμε μία επιχείρηση που πολλές φορές δεν έχει τα μέσα να αντιμετωπίσει τέτοιες αποζημιώσεις. Γι' αυτό υπάρχουν και οι ασφαλιστικές εταιρείες, είναι υποχρεωτική ασφάλιση του οδικού μεταφορέα. Θα πρέπει λοιπόν να είναι άμεση η ευθύνη των ασφαλιστικών εταιριών να ανταποκριθούν και να καταβάλουν τι αποζημιώσει και να μην αναλαμβάνουν την ευθύνη αυτή που είναι ευθύνη των ασφαλιστικών οι μεταφορεί. Επίση, άρθρο 1, παράγραφο 1. Αναφέρεται ατέλεια μεταφορά ή αποσκευών για κάθε επιβάτη. Αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να περιληφθεί σε ένα παράρτημα. Γιατί υπάρχουν βέλτιστε πρακτικέ, θα πρέπει να τι μιμηθούμε. Άλλωστε, οι πρακτικές αυτές χρησιμεύουν για την καλύτερη άσκηση των δικαιωμάτων του καταναλωτή, αλλά και την διασάφηση των ευθυνών των μεταφορέων. Αυτά και επαφή φυσικά στην κρίση του εισηγητού. Ήθελα να παρουσιάσω τις τροπολογίες μου. Φυσικά όποιες προσκρούν ε, στη γνώμη του εισηγητού θα μπορούσαν και να τις αποσύρω. Ευχαριστώ κύριε Τεγκράντες Πασκουάλ. Ήθελα πρώτα να δώσω το λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων εφόσον τα είχα ζητήσει. Γι' αυτό το κάναμε και μετά λάβατε το λόγο και εσείς. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή Αλμπερτίνη για το πολύ αξιόλογο και σχολαστικό του έργο σε ένα τόσο σημαντικό θέμα που κλείνει κατά κάποιο τρόπο τον κύκλο αυτό των μέσων μεταφοράς. Και όπως είπε και ο κύριος Δεγκράντες Πασκουάλ, μιλούμε για επιχειρήσεις με συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Άλλωστε, πρόκειται για επιχειρήσεις που προσφέρουν όλο και περισσότερο ποιοτικές υπηρεσίες. Γι' αυτό και εγώ πρότεινα η εφαρμογή του κανονισμού να γίνει με φιλικό τρόπο από τις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά και τις ανάγκες των αναπήρων ή των ανθρώπων με περιορισμένη κινητικότητα. Θα πρέπει με διάλογο να καταλήξουμε στις καλύτερες λύσεις και στις πιο δόκιμες προτάσεις που θα έχουν και δεσμευτικό χαρακτήρα μια και πρόκειται για κανονισμό. Από αυτή την άποψη είναι χρήσιμος αυτός ο διάλογος για τους διάφορους εξοπλισμούς. Τώρα για τις ε, τροπολογίες που ίσως ε, δημιούργησαν προβλήματα. Στις ε, προθεσμίες, εγώ πρότεινα μείωση από 48 σε 24 ώρες για την προειδοποίηση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είχαμε ραγδαίες εξελίξεις ό,τι αφορά τις συνδυασμένες μεταφορές και γενικώ τη μεταφορά επιβατών. Και τα τελευταία χρόνια προσθέσαμε στις μεταφορές διάφορες ευκολίες και για τους ανθρώπους ε, με περιορισμένη κινητικότητα και για αναπήρους. Οπότε είναι δυνατό μόνο με 24 ώρες ε, προειδοποίηση να μπορούν να έχουν πρόσβαση στον εξοπλισμό που χρειάζονται οι επιβάτες. Δεν χρειάζεται να έχουμε το, τις 48 ώρες. Άλλωστε οι περιφερειακές γραμμές έχουν διάφορους σταθμούς και συλλογικούς και συνδυασμένο με το φορόν, οπότε είναι εύκολο μέσα σε 24 ώρες με την ε, σχετική προειδοποίηση να βρουν το κατάλληλο εξοπλισμό. Δεν χρειάζεται να πετούμε 48 ώρες ε, προθεσμία για να ενημερώνει για την αναπηρία του ο επιβάτης προκειμένου να εξασφαλιστεί ο εξοπλισμός. Αρκούν 24 ώρες. Πιστεύω ότι οι επιχειρήσεις ε, έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και μπορούν να αντιμετωπίσουν εύκολα αυτό το αίτημα του επιβάτη. Διαπιστώνω κύριε Σιγητά ότι έχουμε τις τροπολογίες 108, 109, 110 και 111 που φαίνονται ως σχεδόν ταυτόσιμες. Γιατί σχεδόν ταυτόσιμες, ε, εγώ βλέπω ότι είναι απολύτως πανομοιότυπες. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον από την ε, ισπανική μετάφραση. Από την ισπανική μετάφραση δεν βλέπω διαφορά μεταξύ των τεσσάρων τροπολογιών. Να το διευκρινίσουμε αυτό για να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Προτείνει αντικατάσταση του εξοπλισμού αν έχει χαθεί, μια τροπολογία και δεν ξέρω γιατί χαρακτηρίζονται ως ε, σχεδόν ιονή ταυτόσημες, ενώ κατά τη δική μου άποψη είναι ένα και το αυτό όλες αυτές οι τροπολογίες. Ευχαριστώ κυρία Γιάλα. Αν δεν υπάρχει άλλος που ζητά το λόγο, θα ζητήσω την κυρία Ούτμαν να πάρει το λόγο εν ονόμα της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα, καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για όλη τη δουλειά που επετελέστη τη θεωρούμε έξοχη. Εν γέννη, στόχος μας είναι να παραμείνει το πεδίο εφαρμογής που θα είναι το ευρύτερο δυνατό. Τι ούτω τρόπος εξασφαλίζουμε την ισότιμη αντιμετώπιση. Όχι μόνο όλων των επιβατών, στους διάφορους τρόπους μεταφορών, αλλά και όλων των μεταφορέων. Για μας είναι σημαντικότατο αυτό. Θεωρούμε ότι κάποιες τροπολογίες επιφέρουν διευκρινήσεις χρησιμότατες. Κυρίως οι τροπολογίες που θέλουν να διευκρινίσουν το συσχετισμό μεταξύ της προτάσεως και της οδηγίας περί ασφαλίσεων. Και κάποιες τροπολογίες επίσης που διευκρινίζουν το κείμενο. Είναι χρήσιμες όσον αφορά τις ε, παρεκκλήσεις, όσον αφορά την δομή που έχουν τα λεωφορεία και το θέμα της προσβασιμότητας στα διάφορα μεταφορικά μέσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ότμαν. Να ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Κύριε Αλμπερτίνη, ευχαριστώ τον πρόεδρο που μου δίδει το λόγο και τους συναδέλφους που ανέπτυξαν διάφορες σκέψεις που τις κατανοώ, ήταν λογικές. Αν και από από την έποψη εκείνου που θέλει να πετύχει συμβιβασμό μεταξύ αντικρουμένων συμφερόντων και οραμάτων, δεν είναι όλες οι προτάσεις αποδεκτές. Κύριε Σίμψον, αναφερθήκατε στην απόσταση περισσότερο από ότι στην αφηρημένη έννοια της περιφέρειας και της περιοχής. Διότι κειμενικά η διαφορά έγκυται σε αυτό. Θεωρώ όμως πολύ μεγάλη λεπτομέρεια να μπει αυτή η έννοια, η ποσοτική. Όποιος ήθελε να καλύψει όλες τις υποθέσεις, αστικές, τοπικές μεταφορές και ένας τέτοιος κανονισμός να τα καλύπτει όλα και απ' την άλλη είχαμε εκείνους που θέλουν να εξαιρέσουν αυτούς τους τομείς. Και νομίζω ότι η διατύπωση που επελέξαμε, αφήνοντας εκτός κανονισμού τις αστικές και τοπικές μεταφορές, που θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλη εργασία. Υπό τη διεύθυνση του Προέδρου Σαβαρή θα γίνει αυτή η προσπάθεια. Θα συνταχθούν οι κανόνες που αφορούν τις τοπικές μεταφορές και αστικές τέτοιες. Έλεγα ότι σε αυτό το πλαίσιο, στην επόμενη οδηγία θα αφήσουμε το θέμα αυτό. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις για τους φραγμούς άρθρο 32, τα barriers, του συναδέλφου Μπέργκερ και του κυρίου Σίμψον. Ίσως, σε μια τη σκέψη, θα μπορούσαμε να διευκρινίσουμε καλύτερα τι εννοούμε από τη διατύπωση φραγμή. Αν είναι φυσικός φραγμός που αναφερόμαστε ή νομικός φραγμός. Πιθανόν να βρούμε σωστή διατύπωση. Καλό τις αρμόνες υπηρεσίες και συναδέλφους να αναπτύξουν κάποιες σκέψεις πάνω σε αυτό και είμαι διαθέσιμος να εξετάσω προτάσεις, να τις αξιολογήσω. Ο συνάδελφος Τέρξ που απουσιάζει στιγμιαία έκανε κάποιες παρατηρήσεις. Τις κατανοώ και τις ημερίζομαι εν μέρη. Αφορούσαν παρατηρήσεις στην τροπολογία 45, την τροπολογία 47 και 3. Εκεί προσπαθήσαμε να συμφιλιώσουμε θέσεις. Προφανώς παραμένουν κάποιες απόψεις που δεν συμπίπτουν απολύτως με το κείμενο. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Γίνεται μια αντιπαράθεση και βρίσκουμε όπου είναι δυνατόν μια ισόρροπη διατύπωση και μετά εκφράζονται τοποθετήσεις. Και η πλειοψηφία έχει το νόμιμο προνόμιο να επικρατεί επί της μειοψηφίας. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και στην Επιτροπή των Μεταφορών. Ο συνάδελφος Ντεγκράντες έκανε παρατηρήσεις ακριβέστατες που προσωπικά θεωρώ ότι έχουν λογική και αντικειμενικότητα, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του συστήματος των μεταφορέων, των μικρών μεταφορέων, που έχουν σοβαρή οργάνωση και να λάβουμε υπόψη και τη γενική οικονομική κρίση που πλήττει όλους τους τομείς και το μεταφορικό τομέα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη. Οι παρατηρήσεις σας με βρίσκουν σύμφωνο. Τις εκτιμώ. Είναι λογικότατες. Επίκαιρες. Όπως πάντα. Όσον είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποιοι είναι οι γενικοί μας στόχοι. Από τη μία πλευρά είναι οι μεταφορείς και τα νόμιμα συμφέροντά τους, από την άλλη είναι οι επιβάτες και αν μέσα σε αυτούς του επιβάτες είναι αυτοί με μειωμένη κινητικότητα που και αυτοί έχουν κάποιες προσδοκίες και αυτός ο κανονισμός όπως λέει και ο τίτλος έχει σκοπό να διευρύνει και να ενοποιήσει τα δικαιώματα των επιβατών, να τα παγιώσει. Χρειάζεται σύμπτωση μεταξύ αντικρουμένων απόψεων. Δύσκολο να βρεθεί το σημείο ισορροπία. Επιφυλάσσομαι από αυτόν όμω, τον όσον είπε ο κ. Δεγκράντη, να το συζητήσω ενδελεχέστερα το θέμα μαζί του και ή δυνατόν να βρούμε μια διατύπωση που να γίνεται αποδεκτή έστω και εν μέρη από τον κύριο Δεσάντης. Την Γκράντες μας συγγνώμη. Η κυρία Γιάλα Σέντερ έκανε κάποιες παρατηρήσεις, κάποιες επικρίσεις άκουσα για κάποιες στοιχές και άφησε όμως να δοθεί κάποια απάντηση, περιμένει απάντηση εγώ δεν μπορώ να δώσω απάντηση, η γραμματεία θα τις δώσει, αλλά η τοποθέτηση της κυρίας είναι απόλυτα λογική. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αύριο θα ψηφίσουμε βάσει καταλόγου ψηφοφορίας που ήδη έχει καθοριστεί, αλλά επιφυλάσσομαι μέχρι την Ολομέλεια να συζητήσω μαζί σας και με τους κοιόδης συγητές και με όλους τους συναδέλφους για να εμβαθύνουμε σε διάφορα ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Αλμπερτίνη, για τις διευκρινήσεις που μας δώσατε. Να σας πω ότι όσον αφορά την, τις αστικές μεταφορές, θα προτείνουμε μια χάρτα κινητικότητα σε αστικές μεταφορές, αλλά πόρο απέχει από το να μετατραπεί σε μια νομοθετική πρωτοβουλία. Δεν προτείνω κάτι τέτοιο άμεσα στην έκθεσή μου δεν είναι του ίδιου νομικού επίπεδου το κείμενο που ετοιμάζω εγώ με αυτό που ετοιμάζετε εσείς, να το διευκρινίσω αυτό. Ακόμα και αν ελπίζουμε να εισακουστούμε στο μέλλον, υπάρχουν και αντιρρήσεις να υπάρχει χάρτα της αστικής κινητικότητας. Κυρίως στην ομάδα σας υπάρχει αυτή η αντίρρηση. Είμαστε σε διαφορετικό επίπεδο. Διότι εδώ μιλάμε για κανονισμό που θα εφαρμοστεί άμεσα και, και τώρα η, η άλλη δική μας είναι έκθεση Πρωτοβουλία που ρίχνει τον μπαλάκι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν θα μα πει εκείνη πότε θα περάσει μετά από αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή διευκρίνηση θέλω να κάνω. Αν θέλετε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συζήτηση. Να περάσουμε στην έκθεση του κυρίου Μισελ Τέσνη για τα δικαιώματα των επιβατών στι θαλάσσιε μεταφορέ. Να δώσω το λόγο λοιπόν στον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Δύο ήταν οι βασικές αρχές ε, που με καθοδήγησαν στην προσέγγιση μου για την έκθεση. Καταρχήν, η ισοτιμία των δικαιωμάτων των ε, επιβατών σε, όλους, σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Θαλάσσιες πλωτές και αερομεταφορές. Και ιδιαίτερα μέρημνα για τους ανθρώπους με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα. Επίσης προσπάθησα, ξεκινώντας από το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να λάβω υπόψη τις δυσκολίες αυτού του θέματος, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε μια γεωγραφική ανομοιομορφία, από τη Βαλτική μέχρι τη Μεσόγειο, έχουμε τα ελληνικά νησιά και μεγάλη ετερογένεια μεταξύ των ποτάμιων μεταφορών, πλωτών μεταφορών και των ναυτιλιακών θαλάσσιων μεταφορών. Όλες αυτές τις ανομοιομορφίες προσπάθησα να τις λάβω υπόψη. Έχουν κατατεθεί αρκετές τροπολογίες για την έκθεσή μου ιδιαίτερα για το θέμα της άρνησης επιβίβασης ε, και ε, διευκρίνηση ορισμένων θέμάτων της Επιτροπής όπως ε, τον ρόλο των λιμένων, των εθνικών οργανισμών, των κουραζιέρων και των επιβατών σε κουραζιέρες κτλ. Το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση σε γενικές γραμμές, δεν χρειάστηκε ρηξικέλευτες αλλαγές. Σε σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μου με τους σκιώδεις ηγητές. Καταρχήν ήταν πολύ αγαστή η συνεργασία μας και πολύ αποτελεσματική. του ευχαριστώ θερμά. Προσπαθήσαμε να διορθώσουμε ορισμένα σημεία, ιδιαίτερα αυτά που είχαμε επισημάνει στη συνεδρίαση της 17ης Φεβρουαρίου, για παράδειγμα. Την εξαίρεση ιδιαίτερα στις πλωτές μεταφορές, στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις και τι θαλάσσιες μεταφορές για τις αστικές ή υποστικές μεταφορές ένα θέμα προσφυλά στον κύριο Σίμψον. Ορισμένα από τα σημεία της έκθεσης ε, είναι τα πιο σημαντικά. Άρθρο 7. Το κίνητρο της άρνησης. Ο λόγος για την άρνηση επιβίβασης. Για το σημείο αυτό έχουν κατατεθεί αρκετές τροπολογίες. Εγώ θα προτιμούσα να εμείνουμε στην τροπολογία 8, δηλαδή ο, η αναπηρία να μην είναι ο λόγος για την άρνηση επιβίβασης. Παρόλο που εφαρμόζονται οι κλασικοί όροι, αλλά οι κλασικοί όροι για την άρνηση επιβίβαση είναι για όλους τους επιβάτες και δεν θα πρέπει να στιγματίζουμε συγκεκριμένα τους αναπήρους. Σε ό,τι αφορά τι τις για την παροχή συνδρομής, άρθρο 12 είναι, είναι επικίνδυνη η τροπολογία 92, γιατί εκεί μειώνει τη δυνατότητα πρόσβασης στη συνδρομή. Ο μεταφορέας προτείνει την ώρα που θα καταθάσουν οι ΠΕΜΕΡ, κάτι που δεν είναι σωστό. Η τροπολογία τώρα 102 και 106 του κυρίου Γιαρζεμπόφσκι. Του το επισήμανα και στη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών είναι έως και ανησυχητικέ θα έλεγα οι τροπολογίες του, γιατί στο 102 προτείνει ολοσχερή κατάργηση του άρθρου που μιλάει για την, κατάργηση, για την κατάρτιση του προσωπικού που έρχεται σε άμεση επαφή με ανθρώπους με μειωμένη κινητικότητα, γιατί εμείς πιστεύω ότι πρέπει να προηγείται κατάλληλη επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού που έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα και επίσης ε, ε, άρθρα που αφορούσαν την ε, αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας εξοπλισμού, αναπηρικής απολυθρώνας ε, κτλ. Και αυτό το άρθρο πρότεινε κατά, κατά, να καταργηθεί ο κ. Γερζεμπόφης και δεν το καταλαβαίνω. Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις ε, των άρθρων 18, 19 και 20, σε περίπτωση ακύρωσης. Εκεί καταλήξαμε στη συμβαστική τροπολογία για τις ε, εξαιρετικές περιστάσεις. Εκεί υπήρξε συμφωνία επί της αρχής προκειμένου να προσδιοριστούν αυτοί οι, οι όροι. Υπάρχουν φυσικά κάποιοι α, όροι σε ό,τι αφορά τους, με, τις μετεωρολογικές συνθήκες, την κατάσταση της θάλασσας. Σε αυτό συμφωνούσαμε, αλλά όχι ε, λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πλοίου ή του, για λόγους του μεταφορέα σε ό,τι αφορά για την μείωση των τρόπων αποζημίωσης δεδομένων των διατάξεων που έχουμε για τις σιδηροδρομικές και τις αεροπορικές μεταφορές και από τη στιγμή που θέλουμε ισοδύναμη προστασία, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εναρμόνιση για όλα τα είδη μεταφοράς. Κάτι που προβλημάτισε και τον εισηγητή Αλμπερτίνη. Αυτά σε γενικέ γραμμέ και περιμένω τα σχόλιά σα, επαναλαμβάνοντα ευχαριστίε μου προ του και εισηγητέ για τη συνεργασία του. Περιμένω τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και τις αντιρρήσεις ακόμη για ορισμένα σημεία για τα οποία δεν επετάχθη συμφωνία. Σας ευχαριστώ κύριε Λίχτεμπεργκερ. Yeah, σας ευχαριστώ. Εδώ έχουμε ακόμα πιο έντονες δυσκολίες στο θέμα αυτό, γιατί εδώ πέρα εμπλέκονται και τα λιμάνια και οι γραμμές μας δυσκολεύει λοιπόν η κατάσταση, όπως μας δυσκόλεψε αρχικά και η κατάσταση και με τις αερομεταφορές. Και αυτό φυσικά μας οδήγησε και στην κατάρτιση ιδιαίτερων διατυπώσεων. Τα καταφέραμε αρκετά καλά νομίζω. Φυσικά να αποκλειστούν οι θαλάσσιες μεταφορές όταν θεωρούνται αστικές μεταφορές. Καταρχάς θα σκεφτούμε σίγουρα όλη τη Βενετία, αλλά υπάρχουν και άλλες πόλεις που είναι πολύ σημαντικές ε, οι θαλάσσιες μεταφορές στις πόλεις και ελπίζω λοιπόν να καταφέρουμε να τα περάσουμε αυτά και νομίζω ότι οι ρυθμίσεις για τις καθυστερήσεις δεν μπορούν να ισχύσουν με τον ίδιο τρόπο φυσικά, αλλά η, η δυνατότητα πρόσβασης χωρίς εμπόδια για τους ε, ανάπηρους είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό γιατί θεωρώ ότι πρόκειται θέμα μέλλοντος, αν θέλετε, και εντομίας, πρωτοπορίας. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών υπάρχουν και ιδιαίτερες προσφορές, για παράδειγμα, για διάφορους ασθενείς. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Πολλά σημαντικά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται λοιπόν και χαίρομαι ιδιαίτερα που προβλέπονται παντού τα δικαιώματα των επιβατών. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο δεν θα πατήσει φρένο και πάλι. Και αν δεν γίνει αυτό, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Μπλόκλαντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πάρα πολύ η επικοδομητική συζήτηση για τις τροπολογίες. Έχω κάποια στοιχεία που θα ήθελα να αναφέρω. Καταρχάς για την τροπολογία 65 66 ε, και 67 στον κατάλογο ψηφοφορίας ε, συνοδεύονται από ένα πλήν εκ μέρους του εισηγητή. Ο σκοπός τους είναι ο ίδιος, η κυρία Βορτμαν και ο πρόεδρος Κώστα και εγώ αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να συμπεριληφθεί μια δυνατότητα όταν σε επιβάτης με περιορισμένη κινητικότητα δεν μπορεί να μεταφερθεί, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να βρεθεί μια άλλη λύση. Για παράδειγμα, κάποια μικρά πλοία σε τουριστικές διαδρομές που χρησιμοποιούνται μόνο για πεζούς και για ποδηλάτες. Μόνο οι ποδηλάτες και οι πεζοί μπορούν να ανέβουν στο πλοίο αυτό. Αλλά τα πλοία αυτά, για παράδειγμα, δεν ενδείκνυνται καθόλου για τη μεταφορά επιβατών με αναπηρία. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και νομίζω λοιπόν ότι στο σημείο αυτό θα έπρεπε να συμπεριληφθεί μια εξαίρεση. Και φυσικά αν η δομή του πλοίου δεν καθιστά δυνατή την ε, σωστή μεταφορά των επιβατών, θα πρέπει να το πούμε στους επιβάτες αυτούς, ότι δεν είναι δυνατόν να ταξιδέψετε με το συγκεκριμένο μέσο και θα πρέπει να αναζητήσουμε εναλλακτικέ ε, λύσεις, προκειμένου να μην υποστούν ε, ζημιά, αν θέλετε, και τα συμφέροντα των επιβατών. Άρα να κοιτάξουμε αυτές τις τροπολογίες 65 και 67. Δεν χρειάζεται να συμπεριληφθεί μόνο η δική μου. Α διαλέξουμε μία από όλες για να διατρεθεί η ιδέα, γιατί είναι σημαντική νομίζω. Κατά τα άλλα, συμφωνώ απόλυτα με τις προτάσεις του εισηγητή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Δεγκράντες Πασκουάλ. Sí, gracias, señor presidente. Eh, yo he Κύριε Πρόεδρε, έχω καταθέσει επτά τροπολογίες για την έκθεση αυτή. Η πρώτη νομίζω ότι είναι αξιοπρόσεκτη, γιατί αφορά ένα ευαίσθητο θέμα, το θέμα της προσοχής που δίνουμε στα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα. Σίγουρα είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος στα θέματα αυτά, αλλά θα πρέπει να δούμε και τις λύσεις που υιοθετήσαμε σε άλλα μέσα μεταφοράς. Δεν μπορούμε να κάνουμε τάμπουλα ράζα και μονίμως να ξεκινούμε εκ του μηδενός. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς σε σχέση με τις ηλιμένες μας αποφάσεις και θέσεις. Η πρότασή μου λοιπόν είναι απλούστατη κύριε Σιγητά. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να προβλέπετε ένα πρωτόκολλο ευθύνη σύμφωνα με, την, τον κανονισμό που καλύπτει την μετάβαση των τόμων από το, λιμάνι κατά την άφηξη και την αποχώρησή τους. Νομίζω ότι ο φορέας του λιμένα θα πρέπει να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Άλλωστε, στην πράξη ισχύει αυτό και έχουμε καταλήξει συνένεση. Δεν θα ήταν δύσκολο να καταλήξουμε σε μια αποδεκτή από όλους συμφωνία. Σε ό,τι φορά, το 14-3 και εδώ θέλουμε οι πληροφορίες προς τον ε, επιβάτη να είναι ακριβείς, να είναι αληθείς. Γιατί μερικές φορές ε, στα μικρά γράμματα των συμβάσεων ή των εισιτήριων κρύβονται πολλά επικίνδυνα σημεία. Αυτά θα πρέπει να καταργηθούν. Θα πρέπει με ευανάγνωστα μεγάλα γράμματα να περιλαμβάνονται οι βασικές πληροφορίες για τα δικαιώματα του επιβάτη. Άρθρο 18, παράγραφος 4α9. Εδώ θα πρέπει να έχουμε μια εξαίρεση από την εφαρμογή του προηγούμενου άρθρου ό,τι αφορά την διαταγή του δικαιώματος ε, συνδρομής. Σε περίπτωση που η συμπεριφορά του μεταφορέα είναι επιμελής και δεν οφείλεται αυτός για το ατύχημα. Υπάρχει επίσης ένα διεθνές σύστημα ευθυνών που είναι διαφυσβήτητο και δεν μπορούμε να λέμε ότι από τη στιγμή που πρόκειται για δικαιώματα του επιβάτη, την ευθύνη φέρει αυτόματα ο μεταφορέας. Όχι. Θα πρέπει να δούμε τι σύστημα κάλυψη υπάρχει εδώ. Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική. Θα πρέπει οι ασφαλιστικές εταιρείες να είναι άμεσα υπεύθυνες, να μην περιμένουν να, να τους ασκήσει κανεί αγωγή και να πάνε στα δικαστήρια. Γιατί αν ο καημένο ο μεταφορέας ήταν επιμελής και δεν αποδειχθεί το αντίθετο, δεν μπορεί να κατηγορείται για αμέλεια, γιατί έμεσα αν τον υποχρεώνουμε σε αποζημίωση τον κατηγορούμε για ευθύνη. Το είπα και προηγουμένως. Θα πρέπει να συσχετίσουμε αυτές τις ευθύνες με την κάλυψη από τις ασφαλιστικές εταιρείες αφού είναι ούτως ή άλλως υποχρεωτική ασφάλιση για τους μεταφορείς. Θα πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθούμε και με το θέμα αυτό, για να έχουμε μία σαφή γραμμή δικαίου και να γνωρίζουν όλοι ποια είναι τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. Σε ό,τι αφορά άρθρο 4, για το άρθρο 19 παράγραφος 2, το ίδιο ισχύει και εδώ. Δεν θέλουμε υπερβολικές ευθύνες για, την, για τις εναλλακτικές μεταφορές. Βέβαια, όταν υπάρχει έδειξη για άμεση ευθύνη, θα πρέπει να προσέξουμε για την ευθύνη του μεταφορέα. Άρθρο 24. Από τη στιγμή που έχει αποδειχθεί επιμέλεια του μεταφορέα, δεν μπορούμε να τον κατηγορούμε και να του επιρρύπτουμε ευθύνε. Άρθρο 20 νέο. Αλφα νέο. Και εδώ είναι εξαιρετική κατάσταση. Παρόμοιο χαρακτήρα έχουν όλε μου οι τροπολογίε. Και άρθρο και παράρτημα 2, παράγραφος 7. Και εδώ προσπαθώ να διορθώσω το κείμενο. για τα συνεργεία της κινητικότητας ή και τους εξοπλισμούς. Γιατί ορισμένες, ορισμένες, ορισμένοι τέτοιοι εξοπλισμοί που χρησιμοποιούνται από όλους μπορούν να, να εφαρμοστούν. Αυτά είναι πολύ καλό το έργο σας, πολύ καλή έκθεση. Αν θεωρείτε ότι με τις δικές μου τροπολογίες θα βελτιωθούν ορισμένα σημεία, είμαι απόλυτα πρόθυμος να συνεργαστούμε. Αν θεωρείτε ότι οι τροπολογίες μου διαστρεβλώνουν την έκθεσή σας, δεν πρόκειται να παραμείνω διάλεκτος, είμαι συνεργάσιμος. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν ανυπέρβλητα προβλήματα μεταξύ μας. Ο κύριος Στόκμαν. Κύριε Στόκμαν. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο συνάδελφος ε, εργάστηκε πολύ επίμελος και με μεγάλο πνεύμα συνεργασίας. Να τον ευχαριστήσω για το πνεύμα αυτό που επέδειξε. Με τις τροπολογίες μου, μάλλον συμφωνεί σχεδόν ε, με όλες, αλλά θα ήθελα δύο πράγματα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί δεν επιδεικνύει ευελεξία για τα θέματα αυτά. Το πρώτο είναι σε σχέση και με την αποζημίωση, του. τι μπορεί να αφορά την αποζημίωση από σε λογικής, είναι η, όρις, η ώρα άφηξη. Δεν με νοιάζει αν αργήσει, αν καθυστερήσει, να αναχωρήσει το μέσο μεταφοράς, τι ώρα θα φτάσει με ενδιαφέρει. <laughs> Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν ως επιβάτη, Εκτός και αν ορίσουμε την ώρα που παραμένει κανείς στο πλοίο ως ώρα διακοπών και μου στηρίζουν δηλαδή κάποια ώρα διακοπών. δάλος το μοναδικό λογικό είναι ότι θα πρέπει να μετράει η ώρα άφηξης, όχι και τα δύο. Εντάξει, αν με πείσετε όμως ότι το λογικό είναι το αντίθετο και αν καταφέρετε να ανατρέψετε το σύστημα αυτό, εντάξει, τι να κάνω, θα υποχωρήσω. Κάτι άλλο που έθιξε ο κύριος Πασκάλ. Για τις ενέργειες μεταφορές είπαμε ότι στην τελική ανάλυση οι θα έχουν την ευθύνη για το πώς θα λειτουργήσουν τα συστήματα αυτά. Άκουσα τα επιχειρήματα. Υπάρχουν λιμένες ε, στην Ελλάδα που δεν υπάρχει σχετική διοίκηση λιμένα και τα πράγματα δυσκολεύονται, δυσκολεύουν. Αλλά το θέμα αφορά τις υπηρεσίες στους λιμένες, κατά πόσον είναι εφικτό το θέμα αυτό, ή άλλως να παραμείνουμε στο τωρινό σύστημα. Κατά τα άλλα νομίζω ότι σωστά έχει διαμορφωθεί η έκθεση, με μεγάλο ζήλο, και ελπίζω να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια. Αν Σας ευχαριστώ. Ο κ. έχει το λόγο. Ναι, να αναφερθώ και εγώ στην ε, κατάσταση αυτή σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία. Έχουμε έρευνε στη Γερμανία από το Υπουργείο Μεταφορών ότι 30% των επιβατών αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικότητα. Όχι μόνο τα άτομα που μετακινούνται με καροτσάκι, αλλά οι ηλικιωμένοι, ή μητέρε ή πατέρε με μικρά παιδιά άτομα με προσωρινά προβλήματα που έχουν το πόδι του γύψο για παράδειγμα και ούτω καθεξής. Δεν είναι μικρός λοιπόν ο ρυθμός. Όταν μας λέει λοιπόν ο κύριος Δεγκράντας Πασκάλ ότι είναι ότι είσαστε ανοιχτό στο θέμα αυτό, εντάξει, αλλά αυτό το είχατε πει και για τις ενέργειες μεταφορές και εσείς ήσασταν πάντα εκείνος που πατούσε φρένο όταν παραπήγαινε. Γιατί είχαμε συζητήσει αν θα συμπεριληφθούν και ψυχικά ανάπηροι και είχαμε πει ότι θέλουμε να υπάρξει αυτή η ρύθμιση και δεν θέλουμε να εξαιρέσουμε κανέναν. Υπάρχει απαγόρευση κατά των διακρίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό ισχύει για όλους μεταξύ αυτών και, με τα άτομα, και για τα άτομα με αναπηρία. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε με σαφήνεια ότι αυτό αποτελεί το στόχο μας και φυσικά είναι η εφαρμογή δύσκολη, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να το θέσουμε ως φιλοδοξία. Και θυμάμαι όταν είχαμε ξεκινήσει στη Γερμανία τη δεκαετία του 70, οι Σκανδιναβοί ήταν 30 χρόνια μπροστά. Ήταν αυτονόητα αυτά τα πράγματα τα οποία προσπαθούσαμε να περάσουμε στην Γερμανία με τις κυλιόμενες σκάλες τότε για παράδειγμα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει επιτέλους να διορθωθεί αυτή η κατάσταση και να μην συνεχίσουμε να επινοούμε εμπόδια. Ευχαριστώ. Η κυρία Τικάου έχει το λόγο κύριε Αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών, πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά τα μικρά σκάφη, είναι σημαντικό να ισχύουν οι κατάλληλες συνθήκες για να έχουν οι επιβάτες πρόσβαση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εσωτερική ναυσιπλοεία. Δυστυχώς, πολύ λίγα μέτρα έχουν ληφθεί και τα μικρά πλοία δεν έχουν διευκολύνσεις για την πρόσβαση των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα. Ευχαριστώ κυρία Τικάου. Υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Η ε, κυρία Ότμαν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα επαναλάβω. Les autobus Για αυτό που είπα για τα λεωφορεία και τα πούλμαν. Συγχαρητήρια καταρχάς ε, στον εισηγητή για την έξοχη δουλειά που έκανε και πολλές τροπολογίες που προτείνει και άλλες τροπολογίες έχουν στόχο την ενίσχυση των δικαιωματών επιβατών, άρα είναι ευπρόσδεκτες τροπολογίες και εδώ μέρημνά μας είναι να εξασφαλίσουμε ένα πεδίο εφαρμογής ευρύ για ισότιμη αντιμετώπιση όμως θέλουμε και κάποια ευελιξία για να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στον τομέα. Και εδώ μεταξύ των τροπολογιών υπάρχουν πολλές που θεωρούμε ότι επιφέρουν χρησιμότατες διευκρινήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει ο συγητής να ολοκληρώσει. Κύριε συγητά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω εντάχει να αναφέρω κάποια σημεία, λέει ο κ. όσον αφορά την παρέμφαση Λίχτεμπεργκερ για τα λιμάνια, αυτά που έθιγα στην αρχή. Πράγματι έχουμε ένα κείμενο για τα δικαιώματα των επιβατών και όχι ένα κείμενο για τι υποδομέ. Θα ήθελα να επενθυμίσω ότι αν οι επιχειρήσει δεσμεύονται να δώσουν βοήθεια ε, στου επιβάτε υπάρχουν όμω και κάποια θέματα που εξεταστούν. Τα λιμάνια στην Ευρώπη είναι εμπορικά και μεταφοράς φορτίων. Υπάρχουν κάποια λιμάνια που είναι δικαιωμένα για επιβάτε, αλλά είναι πολύ περιορισμένα. Όπω χωρί ο κ. Στόκμαν μετά, υπάρχουν πολλέ αποβάθρε που δεν έχουν υποδομές, δεν έχουν προσωπικό και δεν μπορούν να υποδεχθούν κατάλληλα τους επιβάτε. Και τι ανακάλυψα ζητώντα με τι επιχειρήσει, ότι και ο πλευρά των επιχειρήσεων φέρει ή για κρουαζιέρε ε, εκφράστηκε η επιθυμία, βούληση στον ανταγωνισμό με άλλε εταιρείε που προσφέρουν τον ίδιο προορισμό ε, να δώσουν αυτή τις υπηρεσίε που πρέπει. Θέλουν να εσωτερικεύσουν αυτού του είδου τι υπηρεσίε. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, διότι είναι επιθυμία των επιχειρήσεων όσον αφορά τις κουραζιέρες. Αν πάρουμε τον ορισμό γενικά, αυτό που καλύπτεται τα 5-40% των πελατών που επιλέγουν αυτή τη διασκέδαση πρέπει να υποδέχονται αυτή την πελατεία και θα πρέπει να προσαρμοστούν στο τουριστικό προϊόν που υπάρχει, που προσφέρουν και αν μπορούν να βελτιώσουν ε, πρέπει να το βελτιώσουν σε σχέση με την πελατεία που θέλουν να προσελκύσουν να για να συμμορφωθούν με έναν κανονισμό. Όσον αφορά τον κύριο Μπλόκλαντ για το 76 και 77 είναι θέμα αρχής. Αν λέμε ότι παραμένει η καθιστική ατάξη, δηλαδή η δομή του σκάφους καθορίζει ποιος θα επιβαστεί ή όχι, θα μελήσουμε την επιλογή μας. Δηλαδή να υποστηρίξουν τα δικαιώματα των καταναλωτών, των επιβατών και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Κύριε Δεγκάντε Πασκάλ, όσον αφορά την κινητικότητα, θα ξεκινήσω διάλογο μαζί σα. Όσον αφορά τη 14.3 και τη 18, μπορούμε κάτι να κάνουμε και να προχωρήσουμε. Όσον αφορά το 4 και το 20α, ίσω να κάνουμε λιγότερα, αλλά θα γίνει ανταλλαγή απόψεων και εγώ μπορώ να συνεχίσω μαζί σα τη συζήτηση εν ώψη τη Ολομελία. Αυτά εντάχει κύριε Στόκμαν, το θέμα της αναχώρησης και της άφηξης είναι και το θέμα της διαδρομής. Μπορεί να καλύψει, παίζει ρόλο η άφηξη γιατί μπορεί να καλύψει καθυστέρηση το σκάφος. Αναφέρει ο Ράφη στο κείμενο. Αν διατηρήσουμε την ώρα αναχώρηση, είναι ότι αν δεν φύγει το σκάφο για διάφορα προβλήματα, θα πρέπει να υπάρχουν κάποια μέρη να εφαρμοστεί το κείμενο. δεν μπορούμε να έχουμε μόνο την ώρα άφηξη στο, στο κείμενο. Έχει σημασία όλη η διαδρομή. Αυτά. είμαστε στη διάθεσή σας. Ψηφίζουμε αύριο. Και είμαστε στην πρώτη ανάγνωση. Λοιπόν, υπάρχει ακόμα και ένα περιθώριο. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Τώρα περάσουμε στην έκθεση Στόκμαν όσον αφορά το πρόγραμμα Μάρκο Πόλο θα δώσω το λόγο στον κύριο Στόκμαν. Είναι ένα σχέδιο κανονισμού. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Στο Μάρκο Πόλο μιλάμε για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών φιλικών ε, μέσων μεταφοράς. Και συμφέρει λοιπόν όλους να καταλήξουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση προκειμένου να δοθούν τα κονδύλια αυτά γιατί μιλάμε για 50 εκατομμύρια μέχρι το 2013. Ο ανεπίσημος τριμερής διάλογος βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και καλέσαμε και τους κοιόδης εισηγητές. Τι καταφέραμε ως τώρα. Την αύξηση για παράδειγμα των επιπρόσθετων ποσοστών από 10 σε 20%. Αυτό απασχόλησε ιδιαίτερα την κυρία Λίχτενμπέργκερ σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες οι, οποία, οι οποίες παρατάθηκαν κατά μισό ε, χρόνο σε περιπτώσεις όπως η σημερινή κατάσταση ύφεσης. Ιδάλλως θα είναι δύσκολος, ε, δύσκολο να κατανεμηθούν σωστά οι πόροι συμπεριλάβαμε και τους λιμένες που ζήτησε η κυρία Σε Συνολικά καταφέραμε να περάσουμε πολλά από τα στοιχεία που πρότειναν οι συνάδελφοι. Γιατί οδεύουμε προς τον Μάρκο Πόλο 3. Καταφέραμε λοιπόν πολλά στοιχεία τέτοια να τα συμπεριλάβουμε και αναμένουμε μία ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να μας απαντήσει για τα θέματα αυτά τα οποία θέσαμε προτού περάσουμε στο Μάρκο 3 και να αξιολογηθούν φυσικά και όλα αυτά τα στοιχεία. Ποιο είναι ο αντίκτυπος, για παράδειγμα, του προγράμματος, πώς ε, λειτουργεί η υπηρεσία, η εκτελεστική που υπάρχει από το Μάρτιο του 2008. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, διαφοροποιήσεις αναπροϊόν. Πώς λειτουργεί η αποφυγή κίνησης. Θα πρέπει να υπάρξουν ξεχωριστά προγράμματα για τις πλωτές μεταφορές. Αυτό ήθελα να το βάλουμε κυρία Βόρτμαν Κόλου. Ύστερα ο κύριος Κώστα για το κατά πόσο μπορούν να επεκταθούν τα προγράμματα και σε γειτονικά κράτη. αν μπορούν ε, οι επιχειρήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συγχρηματοδοτήσουν και άλλα τέτοια θέματα τα οποία θέξαμε τα συμπεριλάβαμε και για τη σύνδεση με το πρόγραμμα δράσης για την επιμελητία και σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του TENS, παρόλο που το κόμμα δεν έχει γίνει, αυτό κατά επιθυμία της κυρίας Αγιά Σέντερ. Και άλλα θέματα. Νομίζω ότι θίγονται τα θέματα που μας ανέφεραν οι συνάδελφοι χωρίς να διακυβεύσουμε ενδεχόμενη συμφωνία. Κάποια θέματα δυστυχώς αναγκάστηκα να τα απορρίψω. Δεν τα ξεκινήσαμε καν να τα συζητάμε με το Συμβούλιο και επιμένω στη θέση αυτή. Για όλα αυτά τα οποία ανάφερε ο κύριος Δεγκράντος και ο κύριος Φερνάντες για την ειδική λειτουργία για τις περιφέρειες που προσπάθησαν να κατοχυρώσουν δεν είναι ότι δεν το λαμβάνω αυτό σοβαρά, αλλά δεν καταστρώνουμε εδώ πολιτική συνοχή. Εκεί θα πρέπει να κοιτάξουμε τα διευθυντικά ταμεία. Εδώ μιλάμε για τους ίδιους όρους πανευρωπαϊκά για τέτοια προγράμματα επιδότησης. Γι' αυτό και θεωρώ ότι δεν μπορούν να επιτρέπουν ιδιαίτερε συνθήκες, ιδιαίτεροι όροι για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, όπω ζητάει ο κύριο Μπλόκλαντ. Μειώσαμε τις ε, κατώτατες τιμές προκειμένου να μπορούν και οι μικρές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν και να ενισχυθούν και αυτές. Και την επανεισαγωγή στην διαδικασία της επιτροπολογίας που ζήτησε η κυρία Τικάου και αυτή ε, την απορρίπτουμε. Χαιρόμαστε που επιτέλους έχουμε μία υπηρεσία που λειτουργεί για το σκοπό αυτό. Δεν έχει νόημα λοιπόν αυτό που προτείνεται. Κυρία Τσικάου επίσης. Και οι υπόλοιπε παρατηρήσεις σας πραγματικά δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Θα αναφερθώ στις οριακές τιμές για την αύξηση των τιμών αυτών από 35% σε 80%. Ε, δεν μου φαίνεται πραγματικά σκόπιμο αυτό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η υπηρεσία, επιτελεί το έργο της σωστά και καλά πιστεύω και συζητήσαμε μήπως την τεχνική αρρωγή θα μπορούσαμε να επιδείξουμε μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου στα κράτη-μέλη όπου ενδεχομένως δεν υπάρχει τέτοια έντονη παρουσία να μπορούν να ενισχυθούν πιο έντονα για τη μείωση του ελάχιστου χρόνου, νομίζω προς την ε, αντίθετη κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε στην ε, παράταση αυτής της προθεσμίας. Υπάρχουν δύο θετικά στοιχεία τα οποία θα ήθελα να αναφέρω για τις διαπραγματεύσεις ε, στο Συμβούλιο για τη μείωση των οριακών τιμών, οι οποίες θα επιτρέψουν να εισέλθουν στο πρόγραμμα ακόμα πιο πολλά έργα Γι' αυτό λοιπόν η μείωση των οριακών τιμών αυτών είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα θυμάστε ότι στο Μάρκο Πόλο 52 είχε αρχικά προτείνει, είχαμε αρχικά προτείνει 52 τόνους χιλιόμετρα ένα έτος, μετά προτάθηκαν 80 και τελικά καταλήξαμε στα 60. και για τους ε, θαλάσσιους ε, διαδρόμους θα αλλάξει η κατάσταση. Έχουμε καταλήξει πλέον στο 200 χιλιόμετρα ένα έτος. Νομίζω ότι όποιος ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό θα μπορέσει με χαρά να διαπιστώσει ότι περιορίζονται αυτές οι οριακές τιμές και είναι θετικό αυτό το μήνυμα. Και θα χαιρόμουν αν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε στην πρώτη ανάγνωση, προκειμένου το πρόγραμμα να διατηρηθεί, αν θέλετε, γιατί τρέχει μια χαρά, ίσως όχι τόσο καλά όσο θα θέλαμε, αλλά είναι σημαντικό το πρόγραμμα αυτό και γι' αυτό είναι απαραίτητες και οι βελτιώσεις και οι διορθώσεις αυτές που θα κάνουμε. Ευχαριστώ κύριε Στόκμαν. Ο κύριος Νταγκάντες Πασκουάλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα είμαι λακωνικός. Είχα υποβάλει έξι τροπολογίες με την συνυπογραφή του κυρίου Φερνάντες που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε θέματα υπεραπόμακρων περιοχών Υπέβαλα λοιπόν τις τροπολογίες μου προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα των υπεραπόμακρων περιοχών. Νομίζω ότι αυτό είναι πια αναγνωρισμένο από όλους. Αν θέλουμε να είμαστε δίκοι θα πρέπει να εξαιρέσουμε τις υπεραπόμακρες περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους. Ο κύριο Στόκμαν σε μια πολύ φιλική επιστολή που μου έστειλε μου είπε ότι κατά τη γνώμη του ο υπεραπόμακρος χαρακτήρας δεν είναι αξιοκαταφρόνητος, αντίθετα βρίσκει τη θέση του στην έκθεση. Αλλά δεν είναι λόγος για εξαίρεση από τις διατάξεις. Ενώ η συζήτηση ή η έγκριση αυτών των τροπολογιών ίσως δημιουργήσει προβλήματα Στι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και δεχομένως η έγκριση αυτών των τροπολογιών οδηγεί σε απόρριψη της πρώτης από το Συμβούλιο. Σημειώνω τι ανησυχίε του, αλλά επιμένω στι τροπολογίε μου, στην ουσία τους, παρόλα αυτά μπορώ να τις αποσύρω, αλλά ελπίζω να δείξουμε την ευαισθησία προς υπεραπόμακρες περιοχές για να μην αισθανθούν ακόμη ε, πιο απομονωμένες. Γιατί δεν είναι από καπρίτσιο η που ζητούν ιδιαίτερη μεταχείριση αυτές οι υπεραπόμακρες περιοχές, αλλά επειδή ακριβώς έχουν ε, ιδιαίτερες ε, ευαισθησίες και εξέχοντα χαρακτηριστικά και που είναι δίκιο να τύχουν διακριτικής μεταχείρισης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την προσπάθεια που κατέβαλα να επιταχύνει τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ που συμπεριλάβατε και τα θέματα που σας ε, ζήτησα. Ένα πρόβλημα έχω στην τροπολογία υπαριθμών 17, όπου γίνεται λόγος για να μην αναφέρονται υπεραβολητικέ επιπτώσεις, αλλά μόνο το εξωτερικό κόστος. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι επαρκές. Δεν μπορούμε μόνο να περιορίσουμε δηλαδή το περιβάλλον σε θέματα κόστους και τα έργα αυτά δεν εκφράζονται πάντα σε τιμές εξωτερικού κόστους. Δεν μπορούμε να τα θέσουμε όλα υπό νομισματικούς, αν θέλετε, όρους. Γι' αυτό θα ήθελα να συμπεριληφθούν και τα δύο στοιχεία αυτά. Αν δεν το θέλει αυτό το συμβούλιο, ε, τι να κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι καλύτερο είναι να καταρτήσουμε μια σωστότερη έκθεση, γιατί υπό κάποιους όρους θα αποκλείονταν πάρα πολλά έργα. Και αυτό θεωρώ ότι δεν θα ήταν σωστό. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να το συμπεριλάβουμε αυτό το θέμα. Γιατί πραγματικά αυτό αφορά το πόσα έργα τελικά θα συμπεριληφθούν. Ευχαριστώ. Κύριος Μπλόκλαντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον εισηγητή Στόκμαν για την έκθεσή του και θεωρώ ότι είναι εξαιρετική η έκθεση. Γιατί ο περιορισμός των οριακών τιμών θα καταστήσει το πρόγραμμα πιο προσιτό. Στις τροπολογίες μου 1235 και 36 σκοπός μου ήταν να δώσουμε στις μικροεπιχειρήσεις την ευκαιρία να θεωρηθούν επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Ξέρω ε, φυσικά ότι θα ήταν δυνατόν να σχηματίσουν όμιλο κάποιες μικρές επιχειρήσεις, αλλά αυτό συχνά παρουσιάζει περιπλοκές και δυσκολίες. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι με τις τροπολογίε αυτές νομίζω ότι μπορεί να συμφωνήσει το Συμβούλιο με τις τροπολογίες αυτές και θα έδιναν πραγματικά μια ευκαιρία για αυτές τις μικροεπιχειρήσεις. Δεν ε, ήθελα δηλαδή να δημιουργήσω προβλήματα, απλά θεωρούσα ότι δεν ε, θα παρουσίαζε πρόβλημα αυτή η λύση και να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν πραγματικά υπάρχει κάποιο εμπόδιο για αυτές τις μικροεπιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ και Μπλοκλάντη, κυρία Τικάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις προσπάθειες που κατέβαλε όσον αφορά την τροπολογία 7 περί επιτροπολογίας θα ήθελα να την αποσύρω. Για την 23 και 26 τις υπέβαλα, τις τροπολογίες αυτές, διότι θεωρούσα ότι η κοινοτική οικονομική ενίσχυση για το διατροπικές μεταφορές και για την εκμάθηση επίσης για την μαθητεία θα πρέπει να αυξηθεί ε, μέχρι το 80%. Το λέω αυτό διότι δυστυχώς το Μάρκο Πόλο 1 και 2 έχουν καθυστερήσει πολύ, δυστυχώς. Τα κονδύλια που δόθηκαν σε αυτά τα προγράμματα δεν χρησιμοποιήθηκαν με επαρκή τρόπο από τα κράτη-μέλη. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ουσιαστικό να βελτιωθεί η κατάσταση, να βελτιωθούν οι δυνατότητες, η προσβασιμότητα αυτών των προγραμμάτων. Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, πρότεινα να μικρύνει η περίοδος να πάει στους 24 μήνες για την υποβολή της αίτησης όσον αφορά τον εύξηνο πόντο και όλη την περιοχή αυτή το πρόγραμμα Μάρκο Πόλο έχει πολύ μεγάλο δυναμικό κυρίως για τα νέα κράτη-μέλη το, το Μάρκο Πόλο 2 είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη βελτίωση της ναυσιπλοείας και για την ανάπτυξη ειδικών συγκεκριμένων προγραμμάτων. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ έχει το λόγο. Συγχαρητήρια κύριε Στόκμαν, γιατί εσείς ήσταν ο πρωτεργάτης αυτού του προγράμματος, του κοινοβουλευτικού προγράμματος Μάρκο Πόλο και το παρακολουθήσατε με ιδιαίτερη προσοχή και με πολύ στοργή και φροντίδα και τον ευχαριστώ θερμά για την ευαισθησία που έδειξε προς τις ε, τροπολογίες μου, τις δύο πρώτες τροπολογίες που στόχο είχαν ε, την ε, βελτίωση και τη συμπλήρωση των κινήτρων για το πρόγραμμα αυτό, προκειμένου να προωθηθεί ακόμη περισσότερο. Παρόλο που λυπούμαστε που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχει εφαρμοστεί με την απαραίτητη επιτυχία, την αναμενόμενη επιτυχία. Και το θέμα της πλατφόρμας με τα dry ports είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι από τα πιο ενδιαφέροντα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να δούμε πώς θα διαρθρώσουμε τις διάφορες περιοχές εσωτερικά και να μην τους δημιουργήσουμε το αίσθημα της απομόνωσης. Επίσης, μην ξεχνάμε και τη συζήτηση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τη διαδικασία αναθεώρησης που έχει ξεκινήσει. Όταν ανοίξουν τα δίκτυα προς όλο το σύστημα των λιμανιών και όλες τις εξωτερικές ροές, το Μάρκο Πόλο θα εμπλουτίσει αυτή τη συζήτηση αναθεώρησης των ε, δικτύων. Γι' αυτό και ευελπιστώ ότι θα διεκπαιρεωθεί γρήγορα το θέμα του Μαρκοπόλου για να έχουμε ένα επιπλέον στοιχείο στις επόμενες μας συζητήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σέλε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ευχαριστήσει τον κύριο Στόκμαν. Έξοχη δουλειά που έκανε, έξοχη έκθεση. και ήταν αποτελεσματικότατος ο τρόπος διεξαγωγής του τριμερούς διαλόγου. Προσβλέπουμε στην επόμενη συνεδρίαση αυτού και ελπίζουμε ότι εκεί θα καταλήξουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά σε ένα αποτέλεσμα. Πρώτη ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Καλωσορίζω επίσης την προθυμία πολλών μερών πολλών μελών μάλλον αποσύρουν τροπολογίες και θα ήταν σημαντικό αυτή η αναθόρηση του κανονισμού να εστιαστεί σε αποτελεσματικότερη εφαρμογή κατά την υπόλοιπη περίοδο. Και καλωσορίζουμε αυτές τις αναφορές που περιέχονται για την προπαρασκευαστική έκθεση που θα μας οδηγήσει στο Μάρκο Πόλο 3. Εκεί θα αναφέρονται διάφορα ζητήματα που είναι σημαντικότατα. Η την 17 σημειώνω τα σχόλια της κυρίας Λίχτεμπεργκερ. Θέμα λογικής είναι το εξωτερικό κόστος και η συμπερίληψη των περιβαλλοντικών δαπανών. Μάλλον να εξαιρούνται οι δαπάνες για το περιβάλλον, τα ωφέλη για το περιβάλλον εντάξει. Θα το σκεφτούμε θετικά στοιχεία όσον αφορά το περιβάλλον. Θα το δούμε αυτό, το συζητήσουμε στον άτυπο τριμερή διάλογο. Τώρα για τις μικροεπιχειρήσεις. Θα θέλαμε αυτές να εφαρμόζουν το πρόγραμμα και να συμπεριλαμβάνονται. Ταυτόχρονα όμως φοβούμε ότι δεν αποτελεί αυτό αποτελεσματική χρήση των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δηλαδή, το κόστος διαχείρισης σταθμιζόμενο προς τα ωφέλη που θέλουμε να πετύχουμε στο του προγράμματος, αν αυτός ο λόγος είναι πολύ υψηλό, δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό έχουμε τα όρια. Αν μειωθούν τα όρια πολύ, τότε το κόστος όφελος μειώνεται ακόμα. Μειώνεται το όφελος. Συναρτήσει του κόστους διαχειρίσεως των προγραμμάτων. Όμως είμαστε στα όρια του εφικτού. Και η αρμόδια υπηρεσία είναι βασικός παράγων να δίνει βοήθεια μέσω ενημέρωσης, μέσω άμεσης βοήθειας, μέσω υπολογιστού online προς τους ετούντες και αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος τις μικρές επιχειρήσεις και τις μικροεπιχειρήσεις. για τις τροπολογίες 23 και 27 της κυρίας Τικάου. και το συσχετισμό με τις συνολικές δαπάνες. Διπλασιάζουμε από ένα ευρώ σε δύο ευρώ, σε 500 τόνους ανά χιλιόμετρο. Το να πάμε στο 80% κυρίας Τικάου είναι κάτι μη ρεαλιστικό. Αν πάμε στο 80% ακόμα και στα περιορισμένα προγράμματα που χρηματοδοτήσαμε υπό το παρόν καθεστώς, θα ξεπερνούσαμε κατά πολύ τη διαθέσιμη χρηματοδότηση. Υποτίθεται ότι χρηματοδοτούμε προγράμματα που είναι βιώσιμα υποτίθεται μακροπρόθεσμα. Εάν το 80% των δαπανών χρηματοδοτούνται για μια περίοδο πολιετή, πώς μετά τη λήξη της χρηματοδοτήσεως τα προγράμματα θα εξακολουθούν να Εμείς δεν θέλουμε να δημιουργούμε βραχυπρόθεσμα προγράμματα που ξεψυχάνε άμα σταματήσει η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θέλουμε να υποστηρίζουμε τα συμπροματικές δαπάνες και να καλύπτουμε τις αβεβαιότητες όταν εκινούν τα προγράμματα, αλλά θέλουμε να εφαρμόζονται μακροπρόθεσμα τα προγράμματα. Παρομοίως για τη μείωση του ελάχιστου χρόνου για τα προγράμματα στου 24 μήνες. Θεωρούμε ότι 24 μήνες είναι πάρα πολύ μικρή περίοδος για να είναι βιώσιμο ένα πρόγραμμα και να πετύχει πραγματικά τη βιωσιμότητα που απαιτείται. Αν μειώσουμε λοιπόν το ελάχιστο χρονικό διάστημα σε 24 μήνες, θα χρηματοδοτούμε προγράμματα που θα κινδυνεύουν να εξαφανιστούν στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σέλε. Ο κύριος Στόκμαν έχει το λόγο για να κάνει τα τελικά του σχόλια στην ανακτησή του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Θα δω τι θα μπορέσω να συνεχίσω να διαπραγματεύομαι σήμερα στον πριμερή διάλογο. άλλος. χαίρομαι που θα γίνει και μια γενική συζήτηση όταν θα παρουσιάσουμε την έκθεση. Θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους για όλα αυτά τα θέματα και θα προσπαθήσουμε να το ολοκληρώσουμε στην πρώτη ανάγνωση, γιατί πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο σε ό,τι αφορά την ε, μετακίνηση με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. Αυτό θα αποτελέσει λοιπόν το στοιχείο προσανατολισμού τους. Ευχαριστώ λοιπόν τους συναδέλφους για την καλή συνεργασία και ελπίζω αύριο να μπορέσουμε να ψηφίσουμε με τρόπο που θα μας επιτρέψει τελικά να ολοκληρώσουμε την έκθεση αυτή στην πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αν δεν έχετε αντίρρηση, θα περάσουμε στην επόμενη έκθεση που είναι της κυρίας Γένσεν. Με το χρόνο είμαστε άψογοι. Θα ακούσουμε λοιπόν την έκθεση Γένσεν για τα ευφυή συστήματα μεταφορών. Έχετε το λόγο κυρία Συγγετρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε επιτάπητος και το σχέδιο δράσης και την πρόταση οδηγίας και συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Τσεχική Προεδρία για να διαπιστώσουμε κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα πρώιμης συμφωνίας. Δεν είναι απίθανο, αλλά δεν είναι και εύκολο. Για το θέμα της οδηγίας, πολλές χώρες φοβούνται ότι οι προτάσεις αυτές ε, επεμβαίνουν υπερβολικά στον εθνικό τρόπο λήψης αποφάσεων. Πληθώρα ήταν οι προθεσμίες που κατατέθηκαν και για το σχέδιο δράσης, αλλά κυρίως για την πρόταση οδηγίας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους βουλευτές που συνέβαλαν στη διαδικασία, είτε με την υποβολή τροπολογιών, είτε με τη συμμετοχή τους στη συζήτηση. Για Η γραμμή που ακολούθησε και στις δύο εκθέσεις μου είναι ότι τα συστήματα, τα ευφύ συστήματα μεταφορών καλύπτουν κυρίως τις οδικές μεταφορές, όπως φαίνεται και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε βέβαια συστήματα για το σιδηρόδρομο, για άλλα μέσα μεταφοράς, για άλλους τρόπους μεταφοράς και βλέπουμε ιδέες όπως τα παιχνίδια για τα παιδιά όπως λέμε και διάφορες προτάσεις για τις οδικές μεταφορές. Πάντως η όλη ιδέα και του σχεδίου δράσης και της πρώτης οδηγίας είναι να έχουμε περισσότερη προτυποποίηση και πιο εκτεταμένη εφαρμογή των εφιών συστημάτων μεταφοράς. Πολλές τροπολογίες προσπάθησαν να αλλοιώσουν αυτή τη γενική τάση του προγράμματος, διευρύνοντας το υπερβολικά. Βέβαια, τα FEE συστήματα μεταφορών, το σχέδιο δράσης για τα ITS, αλλά και η οδηγία, θα πρέπει φυσικά να λάβουν υπόψη το θέμα της ε, διαπαφής μεταξύ των τρόπων μεταφοράς. Αλλά το επίκεντρο των δύο προτάσεων είναι οι οδικές μεταφορές. Δεν θα πρέπει να παρεκτραπούμε από αυτό το κεντρικό μας στόχο που είναι οι οδικές μεταφορές. Αυτή ήταν η αρχική πρόταση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και η πρόταση για τα e συστήματα μεταφορών αφορά κυρίως τις οδικές μεταφορές, φυσικά με εξασφάλιση διαλειτουργικότητας και διαπαφής, αλλά χωρίς αλλαγή του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου δράσης και της οδηγίας. Γι' αυτό λοιπόν θα σας προτείνω καταψήφιση της πρώτης τροπολογίας ε, που επιχειρεί να τροποποιήσει τον τίτλο, την ονομασία της οδηγίας. Είμαι κατά και αυτής της τροπολογίας αλλά και πολλών άλλων τροπολογιών που στόχο έχουν την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογή της οδηγίας. Επίσης, για μένα ήταν πολύ σημαντική η διευκρίνηση της οδηγίας, γιατί στόχος της οδηγίας είναι η σύσταση μιας επιτροπής προκειμένου να βελτιωθεί η προτυποποίηση. Και φυσικά θέλουμε να εξασφαλίσουμε την αποφυγή επικάλυψης. Δεν θα πρέπει να επανεφευρίσκει τον τροχό αυτή η Επιτροπή, δεν θα επαναλάβει προηγούμενο έργο ή θα κάνει επικάλυψη, γιατί ήδη ένας βαθμός προτυποποίησης έχει επιτευχθεί. Οπότε η νέα αυτή η Επιτροπή θα κανει επικαλυψη γιατι ηδη ενας βαθμος προτυποποιησης εχει επιτευχθει οποτε η νεα αυτη επιτροπη θα συμπληρώνει το προηγούμενο έργο αξιοποιώντας το και δεν θα το επαναλαμβάνει. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε στενή σύνδεση μεταξύ του σχεδίου δράσης και του έργου αυτής της Επιτροπής. Και αυτό για να διευκρινιστεί περισσότερο η οδηγία και για να εξασφαλίσουμε και ακριβή κάλυψη των τομέων της οδηγίας, ώστε να μην χαθεί η νέα αυτή επιτροπή σε δραστηριότητες επιπαντός επιστητού, αλλά να περιορίζεται στους βασικούς τομείς που καλύπτονται από την οδηγία και το σχέδιο δράσης. Η στάση μου αυτή αντικατοπτρίζεται και στον κατάλογο ψηφοφορίας που έστειλα σε όλες τις ομάδες. και για το σχέδιο δράσης και για την Επιτροπή και για την οδηγία της Επιτροπής. Θέλω να υπάρχει η σαφής αυτή σύνδεση. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με τις τροπολογίες της κυρίας Μπάρση Πατάκη. Επίσης συμφωνώ με ορισμένες από τις τροπολογίες της κυρίας Τσικάου όχι όμως με όλες. Δέχθηκε και κάποιες τροπολογίες του κυρίου Σαβαρή. Για παράδειγμα το συνδυασμό με τις αστικές μεταφορές. Τη διασύνδεση με τις αστικές μεταφορές. Αλλά με άλλες τροπολογίες ε, του κυρίου Σαβαρή διαφωνώ. Ο κύριος ε, Κωστάτσο είπε αλλά ζητούν, ζητά όχι μόνο ευφιέστερες τεχνολογίες και συστήματα, αλλά και καλύτερη ενημέρωση του μεταφορέα και του οδηγού. Το μήνυμα ελήφθη και έβαλα και εγώ σχετική τροπολογία. Κατέθεσα και μία σειρά συμβαστικών τροπολογιών, τέσσερις στον αριθμό, που ομαδοποιούν πολλές τροπολογίες διαπίστωσα ότι το ΕΛΚ ζήτησε ξεχωριστή ψηφοφορία για δύο συμβαστικές λύσεις. Εγώ θα λάβω υπόψη τη μία για τις αστικές μεταφορές, προκειμένου να υπάρχει αυτή η ιδέα της διασύνδεσης, της διαπαφής στα ευφύ συστήματα μεταφορών, γιατί θέλουμε τα ευφύ συστήματα μεταφορών να παρέχουν στον ε, καταναλωτή τις πληροφορίες για τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να μεταβεί από το σημείο Α στο σημείο Β. Γι' αυτό και είναι καλό να εξασφαλιστεί μια διαπαφή μεταξύ των τρόπων μεταφοράς. Το ΕΛΚ ζήτησε ξεχωριστή ψηφοφορία και για τα εισιτήρια που θα πρέπει να είναι συνδυασμένα και να καλύπτουν πολλά μέσα μεταφοράς. Η κυρία Σικάου στην τροπολογία 50 μιλά για την οικονομική ευθύνη. Δεν είναι και πολύ σαφής όμως αυτή η τροπολογία. Τι εννοεί με την ευθύνη αυτή η κυρία Τσικάου. Θα ήθελα να μου το εξηγήσει. Μήπως αντί για το liabilities ε, μπορέσουμε να πούμε responsibilities για να είμαστε σαφείς ως προς το τι καλύπτει ο όρος αυτός. Τροπολογία 52. Μιλάει για κάποια μορφολογικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Νομίζω ότι καλύπτεται αυτή η τροπολογία, αλλά έχω βάλει ερωτηματικό στον κατάλογο ψηφοφορίας, αν και μάλλον το πρόσημο το κατάλληλο θα ήταν να πλήν, γιατί νομίζω ότι καλύπτεται από άλλη τροπολογία, την υπαριθμόν 8. Η τροπολογία 79 της κυρίας Τσικάου μίλα για τη συμβατότητα ε, με τα συστήματα τηλεματικής για τους επιβάτες ε, και τα συστήματα ναύλων και μεταφορών εμπορευμάτων. Και εδώ θα ήθελα διευκρινήσεις πριν κατασταλάξω τι πρόσημα να βάλω στον κατάλογο ψηφοφορίας. Αυτά κύριε Πρόεδρε και περιμένω τις απόψεις των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ κυρία Γέντσεν. Ε, κυρία Τσικά, όχι το λόγο. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την κυρία Γέντσεν, διότι υπήρξε άριστη συνεργασία μεταξύ μας. Έγιναν συναντήσεις με τους κοιόδης εισηγητές και μπορώ να σας πω ότι διεξήχθησαν άκρως επικοδομητικές συζητήσεις. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω για τις συμβαστικές τροπολογίες. Διαπίστωσα ότι συμπεριλήφθηκαν πολλές από τις ιδέες που είχα εκφράσει. Θα ήθελα και θα μου άρεσε να διευρυνθεί αυτή η οδηγία και να καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφορών. Θα ήταν καλό, θα ήταν καλή ιδέα κατά την άποψή μου. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες είναι τροπολογίες που ακολουθούν την κατεύθυνση εκείνου που προτείναμε. Η μόνη επιφύλαξη είναι ότι εξακολουθούμε να περιορίζουμε στις οδικές μεταφορές το πεδίο εφαρμογής και κατά την άποψή μας καλό θα ήταν να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας. Διότι δεν θα έχουμε την ευκαιρία να θεσπίσουμε νομοθεσία για τους έξυπνους τρόπους μεταφορών στο εγγύς Και θεωρήσαμε ότι ήταν καλή ευκαιρία αυτή για να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής τα έξυπνα μεταφορικά συστήματα θα έπρεπε να καλύπτουν όλους τους τρόπους μεταφοράς. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των διαφόρων εφαρμογών και των διαφόρων υπηρεσιών. Νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικό να ασχοληθούμε και με τις αστικές μεταφορές για όλους τους τρόπους μεταφορών. Αυτό ήταν σημαντικό να γίνει. Αλλά ειδικά για τις αστικές μεταφορές το έξυπνο σύστημα μεταφορών θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, διδραματή σημαντικό το, ρόλο. Κατέθεσα ε, τροπολογίε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία αυτά που συλλέγονται και ε, αποτελούν την κύμα εξεργασία στα τέτοια συστήματα μεταφορών θα πρέπει να ε, υπόκειται σε κατεργασία που σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία προσωπικά δεδομένα Επίσης ε, θα πρέπει να επικρατεί και ανωνυμία όσον αφορά τα συλλεγόμενα στοιχεία, όσον αφορά την οικονομική ευθύνη των μεταφορέων και την ευθύνη των μεταφορέων γενικά διαφορετικά θέματα. Όταν μιλάμε για έξυπνα συστήματα μεταφορών, ε, αναφερόμαστε σε αποφάσεις που λαμβάνονται, αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει στοιχείων, στοιχείων που παρέχονται, βάσει πληροφοριών και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ευθύνε των μεταφορέων. Είτε μιλάμε για τα οχήματα, είτε μιλάμε για τις υποδομές. Όσον αφορά την οικονομική πτυχή, είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη που υπέχουν υποχρεώσεις να διαθέτουν επίσης επαρκείς πόρους. Νομίζω ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να δει τι οικονομικούς πόρους διαθέτει και πώς προτίθεται να υποστηρίξει την ε, εφαρμογή και χρήση αυτών των έξυπνων συστημάτων μεταφορών. Δεν θα πρέπει να παραμείνουμε σε διακηρύξεις, θα πρέπει κάθε κράτος μέλος να βρει τα κατάλληλα χρήματα για να υποστηρίξει ε, την σωστή υλοποίηση αυτής της οδηγίας. Όσον αφορά τη συμβατότητα με τις διάφορες τηλεματικές εφαρμογές, ε, πρότεινα σχετικά μια τροπολογία διότι θέλαμε ακριβώς να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και να καλύπτει και άλλους τρόπους μεταφορών. Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι θα δούμε πώς θα πάει η αυριανή ψηφοφορία. Ελπίζω αυτή η έκθεση να εγκριθεί. Είναι σημαντικότατο έγγραφο. Θέλουμε ακόμα μια φορά να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής και να καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφορών και υπογραμμίζω για μία ακόμη φορά που σημαντικό ήταν να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα, η πολυτροπική όλων των εφαρμογών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυριατικά, Ο κύριος Κωνστάτσο για τους ε, πρασίνους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ να επενέσω την κυρία Γένσον, η οποία επέδειξε ιδιαίτερα πνεύμα συνεργασίας και φυσικά τη συνηθισμένη της ε, φιλική διάθεση. Μας ε, κάλεσε σε πολλές περιπτώσεις να διαπραγματευτούμε. Ωστόσο, κοιτώντα ε, τον κατάλογο ψηφοφορία, δεν μου φαίνεται εξίσου φιλικό το γεγονό ότι συμπεριλαμβάνονται τόσα πλήν. Στην πρώτη ανάγνωση, στην πρώτη συζήτηση, είχα ήδη πει ότι τα FEE e οχήματα, τα FEE e αυτοκίνητα είναι κάτι το οποίο δεν μας έβρισκε σύμφωνος. Το είχε πει και ο Μαρινέσκο. Είχα πει ότι από γλωσσική άποψη προκαλεί σύγχυση αυτή η διατύπωση και αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, θέτουμε την τεχνική διάσταση στο επίκεντρο της έκθεσης και αυτό είναι προβληματικό. Δεν έχω καμία αντίρρηση για την τεχνολογία για να πετύχουμε μεγαλύτερη εξοικονόμηση, να προστατεύσουμε το περιβάλλον αλλά να μην καταστεί και αυτός σκοπός της βιομηχανίας. Να κατασκευάζουμε δηλαδή ακριβά αυτοκίνητα για όσους θέλουν να αλλάζουν αυτοκίνητο κάθε 2-3 χρόνια. Και να τα πληρώνουμε δηλαδή όλα αυτά δημοσία το πάνη. Κάτι που είπε η κυρία Τικάτου θα πρέπει να διαβριθεί, να μην περιοριζόμαστε στους δρόμους. Συμφωνώ απόλυτα με αυτή την πρόταση της κυρίας Τικάου. Και ξέρω ότι θα συμφωνήσει και η φιλική κυρία Γένσεν. Εμείς θα θέλαμε κυρίως να μιλάμε για συστήματα πληροφόρηση οθούν. Για παράδειγμα, τα άτομα που δεν χρησιμοποιούν τέτοια συστήματα, τα οποία βρίσκονται σε κάποια άλλη χώρα. Να μην ε, αντιμετωπίζουν τελικά εμπόδια σε ό,τι αφορά την χρήση των δημόσιων μέσων επικοινωνία, συγκοινωνία, συγγνώμη, επειδή πολύ απλά είναι τόσο, δύσκολη, τόσο δύσκολος ο χειρισμός των συστημάτων αυτών. Για την ανωνυμία να πω και δύο λόγια. Χαίρομαι που συμφωνηθηκε που φαίνεται να επικρατεί μάλλον αυτή η, η άποψη για την ανωνυμία, αλλά σε πολλά συστήματα χάνεται η ανωνυμία. Για παράδειγμα, αναφέρεται σε γερμανική εφημερίδα ότι η, η ασφάλεια θα μπορεί να παρακολουθεί τους πελάτες της με το σύστημα αυτό. Για να ελέγχει, για παράδειγμα, την ταχύτητα του κάθε οδηγού κατά πόσο προσπερνάει με τη σωστή ταχύτητα. Και αυτό ανάλογα θα αυξάνει τα ασφάλιστρα. Άρα, πού βλέπετε εσείς την ανωνυμία και το σύστημα e-call. Πρόκειται να είναι ένα σύστημα το οποίο θα το χρησιμοποιούν όχι μόνο φυσικά η αστυνομία, αλλά και οι ασφαλιστικές και οποιοδήποτε. Άρα για ποια ανωνυμία μιλάμε. Θα δούμε τι θα ψηφίσουμε κι εμείς, θα εξαρτηθεί και από την ψηφοφορία. Αλλά αν παραμείνει έτσι η έκθεση κυρία Γέντσαν, πραγματικά θα δυσκολευτώ να την υποστηρίξω. Ευχαριστούμε κύριε Κουστατσέρ. Θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω την έκθεση αυτή να εκφέρω την προσωπική μου γνώμη. Κατέθεσα πολλέ τροπολογίε γιατί πιστεύω ότι ευφύες στι μεταφορέ δεν είναι μόνο ευφύα των οχημάτων και δεν παραβλέπω το σημαντικό οικονομικό διακύβευμα του θέματος αυτού γιατί υπάρχουν και τα ψηλή κονδύλια για το σημείο αυτό. Βέβαια η αυτοκινητοβιομηχανία ε, φαίνεται ότι συμφωνεί. Και έχουμε κάποια προγράμματα στο 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο για την ανάπτυξη της αυτοκίνησης, επίσης ε, κάποια προγράμματα για τους σιδηροδρόμους. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά θέματα που θα καταστήσουν πιο ευφύς τις μεταφορές, χωρίς ταυτόχρονα να κάνουν άκαμπτες τις τεχνολογίες ε, οδήγησης είτε είναι παθητικές, δηλαδή στην ακραία λωρίδα ή ε, ενεργητικές μέσα στα οχήματα. Και επίσης και το θέμα της εμπιστευτικότητας των δεδομένων. Δεν θα πρέπει να θυσιάσουμε την ανωνυμία. Και είναι πολύ εύλογες οι αντιρρήσεις του κ. Κούστατσερ. εκτός ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα οργουλιανό σύστημα με τις προτάσεις αυτές, ε, σαν αυτό που παρουσιάζει ο Όργολος στο βιβλίο του 1984, και στα πλήρη συστήματα, όπως είναι τα συστήματα οδικών μεταφορών, γιατί περί αυτού πρόκειται, η περιορίζεται σε αυτά, το θέμα της ε, μη ολοσχερούς κατάργησης ε, της προσοχής του οδηγού δεν είναι αμεληταίο. Γι' αυτό και κατέθεσα πολλές τροπολογίες διεκδικώντα ένα τμήμα των κονδυλίων, δεν το λέω ακριβώ έτσι βέβαια, ένα τμήμα των κονδυλίων να προσανατολίζεται σε συστήματα που εξασφαλίζουν καλύτερη διασύνδεση των ε, τρόπων μεταφοράς, της ε, υποδοχή των ε, ατόμων μειωμένης κινητικότητας. Αυτό είναι ξυπνάδα. Επίσης, κονδύλια να αφιερωθούν σε συστήματα που θα καθοδηγούν τμήματα του πληθυσμού που έχουν δυσκολίες, τους τυφλούς για παράδειγμα, Υπάρχει ένα αντίστοιχο σύστημα στο μετρό. Τέτοιου είδου ε, συστήματα επίση μα ενδιαφέρουν ή συστήματα που θα ενημερώνουν, θα ενημερώνουν καλύτερα για τις κυκλοφοριακέ συμφορήσει ή για τα προβλήματα που υπάρχουν στην κυκλοφορία. Και αυτοί είναι τρόποι για να γίνουν πιο ευφύ οι, διαφορές, οι μεταφορές και όχι μόνο η τοποθέτηση κάμερας και ραντάρ σε όλα τα οχήματα ή σε όλα τα σταυροδρόμια και τους δρόμους. Για όλα αυτά λοιπόν τα θέματα υπέβαλα τροπολογίες κυρία Γέννησεν, άλλες τις δεχτήκατε, άλλες απορρίψτε, δικαίωμά σας, αλλά προσοχή. Δεν θα πρέπει να ενδώσουμε στις εύλογες ίσως ενησυχίες ή ορέξεις μίας ε, ομάδας πίεσης που είναι αυτή των μεταφορών, γιατί οι μεταφορές είναι ένα πιο πολυσύνθετο και περίπλοκο φαινόμενο και καλό θα ήταν να επικεντρωθούμε στην διατροπικότητα, γιατί εκεί είναι που δεν είμαστε ιδιαίτερα ευφύ. Γιατί ευφύα έχουμε για τις αερομεταφορές, για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, αλλά δυστυχώς η διατροπικότητα έχει περάσει και παραμείνει ανεκμετάλλευτη μέχρι στιγμής. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη για το πώς θα καταστήσουμε πιο ευφυή τα συστήματα μεταφορών στις οδικές μεταφορές. Και το λόγο δίνω στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Τιέλμαν. Would... Καλησπέρα. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, την εισηγητρία για την εξαιρετική εργασία της και τις εκτενέστατες ε, τροπολογίες που λάβαμε για την έκθεση. Εξετάσαμε τις τροπολογίες και θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποιες εξ αυτών. Να ξεκινήσω καταρχάς με τα χρήματα τα οποία ανέφερε μόλις ο κύριος Σαβαρή. Τα χρήματα προέρχονται από το πρόγραμμα TNT κατ' ουσίαν. Και ένα μεγάλο τμήμα του προγράμματος αυτός θα πρέπει να κινηθεί προς τις ευφύς μεταφορές για να τις καταστήσει ακόμα ευφιέστερες. Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται λιγότερο στην πλευρά του δρόμου, γιατί δεν προηγείται οι οδικές μεταφορές. Καταρτήσαμε σημαντικά προγράμματα βασιζόμενοι στο ΤΕΝΤΗ για να προωθήσουμε τις αερομεταφορές και τις ε, πλωτές μεταφορές. Αυτή τη φορά όμως ε, εστιαστήκαμε στις οτικές μεταφορές αλλά και στις διασυνδέσεις με τους άλλους τρόπους μεταφορών. Δεν περιοριζόμαστε δηλαδή μόνο στις οτικές μεταφορές. Υπάρχει πρόσθετη αξία και σε ό,τι αφορά το συνδυασμό με τα άλλα μέσα. Τώρα από την πλευρά την αστική θα χαρούμε να συμπεριληφθούν οι αστικές περιοχές στο πρόγραμμα μεταφορών. Γιατί θεωρούμε ότι αντιμετωπίζουμε όλο και μεγαλύτερα προβλήματα για τη σύνδεση των αστικών περιοχών με τα ευρωπαϊκά δίκτυα και για τη λειτουργία των ε, διαστικών, αν θέλετε, των υπεραστικών μεταφορών. Να θέσω το θέμα της προσωπικής σφαίρας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό για μας. Τόσο σημαντικό που έχουμε αφιερώσει ξεχωριστό τμήμα και στην οδηγία. αναφερόμαστε στην πλήρη εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων οδηγιών για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας προειδοποιήσω ότι αν ε, βάλουμε οτιδήποτε για την ιδιωτική σφαίρα στην οδηγία αυτή, όταν θα τεθεί σε εφαρμογή θα έχουμε προβλήματα σε περίπτωση που η, η οδηγία για την ιδιωτική σφαίρα θα εξελιχθεί. Προσοχή λοιπόν να σεβαστούμε τα θέματα αυτά της ανωνυμίας, τα οποία σέβομαι απόλυτα σε ό,τι αφορά το ITS, γιατί μιλάμε για δεδομένα, για πληροφορίες. Αλλά θεωρούμε ότι δεν πρόκειται για ένα ιδιαίτερο θέμα που αφορά ιδιαίτερα το ITS. Αποτελεί πάντα ένα θέμα σε ό,τι αφορά τα δεδομένα, αλλά τα δεδομένα τα χρησιμοποιούμε και σε άλλα συγκείμενα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ισχυρή πολιτική, μια ισχυρή οδηγία για την προστασία των δεδομένων. Να πω δύο λόγια μετά για την συμβουλευτική ομάδα την οποία καταρτήσαμε. Προτείναμε η Επιτροπή να συνοδευτεί από μια συμβουλευτική ομάδα που θα περιλαμβάνει εκπροσώπους της βιομηχανίας, των τοπικών φορέων, των αστικών περιοχών και το καθεξής. Θεωρούμε ότι το έργο της συμβουλευτικής αυτής επιτροπής θα βοηθήσει την Επιτροπή να λάβει καλύτερες αποφάσεις βάσει των πραγματικών ρεαλιστικών στοιχείων. Αλλά να σας ε, ζητήσω να αφήσετε την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το έργο αυτό θα είναι το καλύτερο δυνατό και όσο πιο διαφανές γίνεται. Τέλος, να πω δύο λόγια για την τροπολογία για τις ειδικέ τεχνολογίες. Υπάρχουν δύο τροπολογίες που αναφέρονται στο SRC, η 51 και η 80. Δεν πρόκειται για κάτι καινοτομικό, πρόκειται για μια τεχνολογία η οποία υπάρχει εδώ και καιρό. Νομίζω λοιπόν ότι την έκθεση αυτή δεν θα πρέπει να αναφέρουμε τις υφιστάμενες τεχνολογίες, αλλά να προεριστούμε στις καινοτομικές τεχνολογίες ή παρόμοια, παρόμοιες τεχνολογίες. Σας ευχαριστώ κύριε Κέλμαν. Να δώσω το λόγο εν κατακλείδη στην κυρία Γένσεν, την εισηγήτρια. Έχετε το λόγο κυρία Γένσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για τα όσα είπαν. Λυπούμε που ο κ. Κούστατσερ αισθάνθηκε κάπως αποκλεισμένο στο τέλος. Δεν είναι ότι δεν θέλω να τον ακούω. Αλλά πάνω σε μερικά ζητήματα απλώς δεν συμφωνούμε. Ας συμφωνήσουμε σε αυτό. Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Προσπάθησα να εστιαστώ στα ζητήματα που ακούστηκαν στην ακρόαση όπου, όπου οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Προστασίας των Δεδομένων είπαν ότι είναι σημαντικό η προστασία των δεδομένων λαμβάνεται υπόψη και μάλιστα στην αρχική φάση αυτή, δηλαδή του καθορισμού των τυποποιημένων ε, λύσεων. Και αληθεύει ότι έχουμε νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θα κάλυπτε το θέμα, έχουμε σχετικό κανονισμό και το ανέφερα αυτό στις σχετικές μου τροπολογίες. Φαντάζομαι ότι πρέπει να δημιουργεί συστήματα που απομονωμένα μεταξύ τους, με συνικά τείχη ούτως όπως για την ίσπραξη διοδίων. Πρέπει να ξέρεις όνομα του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου που είναι υπεύθυνο για την οδήγηση σε κάποιες περιοχές. Για άλλους σκοπούς συλλέγει πληροφορίες παραδείγματος χάρη για κυκλοφοριακή συμφόρηση συλλέγει πληροφορίες για να στέλνει πληροφορίες στους άλλους οδηγούς για να ξέρουν που υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τα στοιχεία λοιπόν μπαίνουν σε διαφορετικά κουτιά για διαφορετικούς σκοπούς. Και έτσι είμαστε σίγουροι ότι πράγματι προστατεύονται τα δεδομένα όσον αφορά την πολυτροπικότητα, τα διάφορα είδη μεταφορών. Πράγματι πρέπει να υπάρχει αυτή η πολυτροπικότητα στο σχέδιο δράσης. Πόσο βάρος έχει αυτό το ζήτημα, αυτό έχει σημασία, πόσο σημαντική είναι αυτή η επιτυχία για τις οδικές μεταφορές. Έχουμε μείνει πίσω, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι έχουμε πάρα πολλούς εμπλεκομένους και κάποιος πρέπει να λάβει πρωτοβουλία. Το θέμα είναι πώς ταθμίζεις τα διάφορα ζητήματα, πού έγκυται η ισορροπία. Διαφωνώ με τη λογική των πρασίνων και των σοσιαλιστών στο συγκεκριμένο θέμα. Για τα χρήματα. Η χρηματοδότηση είναι σημαντικότατο θέμα. Όμως θα πρέπει να δούμε ότι όταν τα κράτη-μέλη ασχοληθούν με το θέμα, όταν ασχολούνται με το θέμα ανησυχούν, διότι πρέπει να δώσουν πολλά χρήματα για τα έξυπνα αυτά συστήματα μεταφορών. Θέλουν ελευθερία επιλογής. Και πρέπει να δεχτούμε σε κάποιο βαθμό ότι θέλουμε μια τυποποίηση, όμως θέλουμε και ανταγωνιστικά συστήματα και έτσι τα κράτη-μέλη να μπορούν να επιλέγουν, να διαλέγουν ποια τεχνολογία επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν. Θα δούμε πώς θα πάει η ψηφοφορία αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία. Σας ευχαριστώ κυρία Γέντσεν, συγχαρητήρια για τη σοβαρότητα της εργασίας σας. Σύνηθες αυτό, ε, εξαιρετικά έχω μια ανακοίνωση. Να κάνει κάποια ανακοίνωση η κυρία Τικάου. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, όσον αφορά τα συστήματα μεταφορών, να σας καλέσω αύριο στο 10.30 να, να κάνουμε τα εγγένεια της εκθέσεως για το Δούναβι που είναι στην ε, βασική Πασαρέλα. Σχετίζεται άμεσα με την Επιτροπή μας και ελπίζω αυτό το ποτάμι να αποκτήσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στον όλο προβληματισμό στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ήταν διαφημιστικό διάλειμμα, λέει ο Πρόεδρος χαριτολογώντας. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ας περάσουμε στην επόμενη έκθεση, αν θέλετε. Οπότε να φορέσω, είναι η δική μου, να φορέσω λοιπόν το καπελάκι μου του συγητή για να θέσω το πλαίσιο της έκθεσης πρώτα απ' όλα. Να υπενθυμίσω στο παρόν κοινό ότι πρόκειται περί εκθέσεως πρωτοβουλίας της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελήψη πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι αρκετά σπάνιο αυτό. Ήταν αρκετά περίπλοκο το να γνωμοδοτήσουμε επί ανακοινωθήσεις πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσπαθήσαμε να καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε λόγω παρετήσεως από το θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κ. Μπαρό, αφού κ. Λογιόλα Παλάσιο, πιο επίμονα, ετοίμασε έκθεση εξουσιμίωτη για την κινητι... βιώσιμη κινητικότητα το 2001. Και εκεί αναφερόταν ότι θα ενδιαφερόμαστε για την αστική κινητικότητα, διότι έχει ιδιαίτερη θέση στην κινητικότητα εν γέννη. 60% των συμπατριωτών μας, των Ευρωπαίων, ζουν σε αστικές περιοχές. Θεωρούμε ότι το 2020 80% παγκόσμιο φαινόμενο αυτό δεν μπορούμε να ενδιαφερόμαστε στις μεταφορές χωρίς να ενδιαφερθούμε για την περιπλοκότητα των αστικών, των μεταφορών σε αστικές περιοχές. Ο Ζακ Μπαγού αποφάσισε ούτως και βάσει των συνθήκων που μας δίνουν κοινή αρμοδιότητα τα κάτι μέλη ανακοίνωσε μια, ένα σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα που δεν μπορεί να καταλήξει κάπου λόγω καθυστερήσεων δεν μπορούσαμε να τηρήσουμε τις διάφορες χρονικές προδιαγραφές που προβλέπει η νομοθεσία πριν τη νέα θητεία που θα ξεκινήσει μετά τις εκλογές του Ιουνίου. Όλες λοιπόν οι ομάδες στο Προεδρείο αποφασίσαμε να τοποθετηθούμε επί της αστικής κινητικότητας διότι πιστεύουμε ότι είναι τόσο σημαντικό το θέμα και θέλουμε πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιληφθεί του θέματος πλήρως και να μας κάνει πρόταση δράση στην επόμενη θητεία. Πρόκειται περί αρκετά παράδοξης εκθέσεως, εκθέσεως πρωτοβουλίας, που δεν έχει καμία νομική εμβέλεια, αλλά έχει πολιτική εμβέλεια μεγάλη και θα είναι πιο σημαντική, διότι θα γίνουν πολύ σημαντικές, αν έχουμε πολύ, ε, πολλές ψήφους να στηρίξουν αυτή την έκθεση. Δεν μπορούμε να διαφορούμε. Θέλουμε τεράστια υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα, το θεωρούμε ευαίσθητο και θεωρούμε ότι είναι και μελλοντικό. Αν όλες οι πολιτικές ομάδες και κυρίως οι συντονιστές. Έτσι αποφασίστηκε στο Προεδρείο. Και έτσι διαβιβάστη στην Επιτροπή αποφασίσαμε να δώσουμε συνέχεια στο Δεκέμβριο σε μια πρωτοβουλία που δεν υπήρχε. Έγινε αυτό, διότι το Δεκέμβριο το Συμβούλιο ανέλαβε υποχρέωση στα σχέδια για το κλίμα να ακολουθήσει πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, το 3 φορές 20%. Συμφωνία του Συμβουλίου για ένα σχέδιο για το κλίμα και ένα πακέτο για το κλίμα και θεωρούμε λοιπόν ότι ήταν αντιφατικό και παράδοξο εάν δεν λαμβάναμε υπόψη τις αστικές μεταφορές στα πλαίσια των μεταφορών εν γέννη. Ξέρουμε πλευράς κλιματολογικής ότι η παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου προέρχεται κυρίως από τις μεταφορές και τη στέγαση, τις κατοικίες και η βιομηχανία έχει το βάρος της, αλλά έχει εξηγιανθεί πολύ η βιομηχανία Είναι και το θέμα τώρα της ρύθμισης μέσω των δικαιωμάτων εκπομπών, αλλά τα προβλήματα είναι πιο δύσκολα για τις μεταφορές. Και η παραγωγή αερίων θερμοκηπίου και διαφόρων μορφών ε, ε τα προβλήματα αυτά είναι στις ζώνες που συγκεντρώνει το πληθυσμό περισσότερο, σε αστικές περιοχές και έχουν επιπτώσει όλα αυτά για την υγεία. Γι' αυτό αποφασίσαμε ότι δεν μπορούσαμε αένα να δείχνουμε ότι δεν κάνουμε κάτι για τις αστικές μεταφορές. Πολύ γρήγορα αυτή η πρωτοβουλία όμως έπεσε πάνω σε αντιρρήσεις, συστηματικές αντιρρήσεις, αλίμονο, ε, που στηριζόταν στην επικουρικότητα. Λοιπόν, εγώ είμαι τοπικός ε, ερετός εκπρόσωπος, πριν γίνω ευρωβουλευτής, ήμουν εκπρόσωπος αυτοδίκησης και ξέρω ποια είναι τα πλεονεκτήματα το να είναι κανείς κοντά στον κόσμο, σε τοπικό επίπεδο. Και πόσο καλή είναι η τοπική δημοκρατία, υπάρχουν τοπικές συνελεύσεις, υπάρχουν άμεσες εκλογές λοιπόν, και καλύτερος έλεγχος διεξάγει σε τοπικό επίπεδο από τον πληθυσμό από στο δικό μας θεσμικό όργανο. Και αν βέβαια η τοπική αυτοδιοίκηση δεν ικανοποιεί τον ε, εκλογέα, ε, είναι πολύ πιο πιθανό να είναι πανεκληγή. Η αρχή της επικουρικότητας θα πρέπει λοιπόν απόλυτα να γίνεται σεβαστή. Αυτό διαπνέει την έκθεσή μου. Δεν είναι πλέον δική μου αυτή η έκθεση άλλωστε. Διότι λόγω του ετερόδοξου χαρακτήρα της διαδικασίας της τολμηρής διαδικασίας της κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας που αναλάβαμε λήψη πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη και τις καθυστερήσεις που είχαμε της πολιτικής φύσεως και που λύγει η θητεία μας τον επόμενο Ιούνιο, λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, ετοιμάσαμε αυτή την έκθεση πολύ μαζί και κάναμε πάρα πολλές διαβουλεύσεις με στους συντονιστές πριν κατατεθεί η έκθεση και ακούσαμε τι απόψει διαφόρων των πολιτικών ομάδων. Δεν λέμε ότι είναι ομόφωνη άποψη επί τη έκθεση. Έχουμε 70 τροπολογίε. Αλλά εργάστηκα σκληρά. Συνεργάστηκα με τον κύριο Ρακ και με τον κύριο Κράμερ και τον κύριο Μπλοκλάντ. Συνεργάστηκα με όλου εκείνου που θα συνεργαστούν εκ των προτέρων πριν καταθέσω την έκθεση. Δημιουργήσαμε αυτή την έκθεση λοιπόν. Έχει το δικό μου όνομα μεν, αλλά έπρεπε να έχει το όνομα όλων των συναδέλφων που είναι παρόντε και φέρουν ευθύνη σε αυτό το χώρο, διότι αποφασίσαμε από κοινού να δώσουμε συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια εντάχει. Να σκιαγραφίσω τους βασικούς άξονες. Ήδη συζητήσαμε τα θέματα εδώ. Πρώτος άξον είναι η βελτίωση της αμοιβέ ενημέρωσης όσον αφορά τις αστικές μεταφορές, στατιστικά στοιχεία κυρίως, να δημιουργηθούν όμως και βήματα συζητήσεων, φόρα, στα οποία κάθε χρόνο να ανταλλάσσονται απόψεις, οι βέλτιστες πρακτικές, να ανοίξουν διάφορες πύλες του στο διαδίκτυο, να δημιουργηθεί ένα μικρό ελαφρύ παρατηρητήριο για τα στοιχεία που αφορούν το θέμα, να φροντίσουμε το ώστε οι οργανωτικές αρχές των μεταφορών στο τοπικό περιφερειακό επίπεδο να συναντώνται τακτικά στις Βρυξέλλες και να εμπλουτίζουν αυτές τον προβληματισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και να γίνει και την αλλαγή των βελτίστων πρακτικών. Αυτό σημαντικότατο. Δεύτερο σημείο. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις αστικές περιοχές να σκεφτούν το θέμα, να το δουν σφαιρικά, να δουν τι γίνεται με τη μετακίνηση. Δεν αφορά μόνο τον τρόπο μεταφορών, αλλά τα συστήματα μεταφορών γενικά, μετακίνησης. Τα συστήματα μετακίνησης δεν μοιάζουν, διαφέρουν από πόλη σε πόλη. Η Βενετία δεν είναι Βερολίνο. Η Βενετία δεν είναι Βερολίνο. Και δεν έχουμε τον ίδιο τρόπο μετακίνησης στη Βενετία όπως το Βερολίνο. Α, όχι απόλυτα τους ίδιους τρόπους μετακίνησης. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό κάθε πόλη, κάθε αστική περιοχή να σκεφτεί τις ιδιαιτερότητες της, να δει τι θέλει να κάνει με το σύστημα μετακινήσεως που έχει, ρόλο του αυτοκινήτου, ρόλου των μαζικών τρόπων μεταφοράς, τι γίνεται με τους πεζούς, τι γίνεται με τα εμπορεύματα, τι γίνεται με τους ποδηλάτες. Πώς όλα αυτά εντάσσονται, πλαισιώνονται, συντονίζονται και πώς όλα αυτά συσχετίζονται με το χρήστη και πώς ενημερώνεται ο χρήστης. Γι' αυτό εδώ προτείνουμε μία προσέγγιση που δίνει κίνητρα, δεν επιβάλλει πράγματα. Κάποιοι συνάδελφοι θα θεωρήσουν ότι είμαι πολύ μετριοπαθή όσον αφορά του στόχου. Διότι έχω κάποιε τροπολογίε που λένε «Ε, χρειαζόμαστε λιγότερα αυτοκίνητα. Ναι, πιθανότατα, αλλά, αλλά δεν συμφωνώ με την κατάσταση των τροπολογιών. Διότι αν λέμε χρειάζεται να χρησιμοποιούμε λιγότερα αυτοκίνητα στη Βενετία, δεν υπάρχουν αυτοκίνητα στη Βενετία. Αυτό θέλω να πω. Δεν θα πρέπει να, να επισέλθουμε σε επιβολή μέτρων. Θα πρέπει να εμπιστευτούμε την ε, τοπική ευφυΐα, την προσαρμογή σε τοπικό επίπεδο. Μπορεί κάπου να θέλουν περισσότερο σιδηρόδρομο. Και εγώ είμαι για περισσότερο σιδηρόδρομο. Αλλά δεν έχουν όλε οι ευρωπαϊκέ πόλει ή πρόσβαση σιδηροδρόμου με τον ίδιο τρόπο. Η ιδέα είναι να υπάρχει ένα πρόγραμμα μετακινήσεω αστικό επίπεδο και όλε οι πόλει να σκεφτούν τι συστήματα μετακίνηση αστική θέλουν και να λάβουν υπόψη και τα ήπια συστήματα. Τρίτο, Θέλαμε να δώσουμε κάποια κίνητρα. Δεν, θα δεν θέλουμε και άλλα, κίνητρα, ε, και άλλα χρήματα ευρωπαϊκά. Δεν θα δοθούν άλλα χρήματα όπως μέσω του Φεντέρα αν δεν γίνει ο δέον προβληματισμός. Δεν θέλουμε να προδώσουμε την επικουρικότητα. Όπως οι άλλες πάλιες βάσεις της Ευρώπης δίνουμε πιστώσεις για να δώσουμε κίνητρα εφαρμογής μιας πολιτικής. Αν αυτή η πολιτική δεν είναι η πολιτική της τοπικής αυτοδιοίκησης τότε δεν δίνονται επιστώσει. Αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ελεύθερη. Να μην ακολουθήσει αυτή την προσέγγιση. Το κάνουμε αυτό και στα πλαίσια του ΦΕΝΤΕΡ. Υπάρχουν κανόνε για το ΦΕΝΤΕΡ. Τα κάνουμε και αλλού. Το κάνουμε και για τα ολοκληρωμένα κοινοτικά προγράμματα. Προτείνω λοιπόν να υπάρξει ένα οικονομικό μέσο για τη χρηματοδότηση τουλάχιστον των μελετών, ίσω και ένα τμήμα των επενδύσεων, χωρί να είναι πολύ επακριβή η όρη, Διότι αυτό εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το σχέδιο δράση τα προτείνει. Από το 2013 μέχρι το 2020. Το 2020, υπενθυμίζω, θα πρέπει να πετύχουμε τους στόχους για το κλίμα. Οπότε ήρθε η ώρα να σκεφτούμε και τι γίνεται στις πόλεις και στις αστικές περιοχές. Τέλος, για να ολοκληρώσω. Προτείνω, προτείνουμε κάποιες διατάξεις σχετικά με την ενεργοποίηση της έρευνας, την ενίσχυση της έρευνας και η κυρία Γέντσεν έφυγε αλλά θέλαμε να εξοικονομήσουμε κάποια, να τις πάρουμε λίγα χρήματα, θέλαμε να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα για τα έξυπνα συστήματα μεταφορών. Θεωρούσαμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι εξαστικό επίπεδο. Θέλουμε να βελτιωθεί η άνεση για το χρήστη. Πρέπει να σκεφτούμε τον χρήστη. Εδώ βρισκόμαστε. Όσον αφορά τι τροπολογίε, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πολλών ειδών τροπολογίες. Υπάρχουν εκείνες κάποιων συναδέλφων της κυρίας Ζόμερ, του κυρίου Φέρμπερ. Αυτές είναι τροπολογίες, πώς να το πω, λίγο ανοιχτές όσον αφορά αυτή την πρόταση. Και λόγω της επικουρικότητας που δεν προδίδεται βέβαια στην πρότασή μας, αρνούνται την προσέγγισή μας. Δεν θέλουν να ασχοληθούμε με την αστική κινητικότητα παρόλο που η πρόταση είναι του Ζακ Μπαρό ουσιαστικά και η κυρία Λογιόλα Παλάσιο έχει ξεκινήσει την όλη προσπάθεια. Υπάρχουν τροπολογίες Φέρμπερ και Ζόμερ που αυτές δεν μπορώ να αποδεχθώ. Επίσης υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες που θα μπορούσα να αποδεχθώ, όπως του κυρίου Χίγκινς για το ITS, για τα ευφυή e συστήματα μεταφορών και διάφορες άλλες τροπολογίες του κυρίου Κρέμερ που ε, είναι πιο περιοριστικές τροπολογίες που φιλοσοφικώς θα μπορούσα να τις υποστηρίξω όσον αφορά την προώθηση διαφόρων άλλων τρόπων μεταφοράς. Δεν λέω ότι πρέπει να υπερψηφίσουμε αυτές τις τροπολογίες, γιατί περνάμε την κόκκινη γραμμή της επικουρικότητας αν το κάνουμε αυτό και αν τις δεχτώ. Τέλος, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες της κυρίας Αγιάλα Σέντερ για την επιμελητία και για τα εμπορεύματα, χρησιμότατες τροπολογίες. Συμπεριλαμβάνω κάποιες τροπολογίες, τις απορρίπτω άλλες, διότι εν μέρη έχουμε καλύψει αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες της Κέτσι όσον αφορά την χρήση των διαθροτικών ταμείων. και όχι αποκλειστικά για τα διεθνωτικά ταμεία, αφορούν και την χρήση τοπικών πιστώσεων και θεωρώ ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πιο πέρα και να αντικαταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την θέσπιση κανόνων για τα μέσα που χρησιμοποιούν τα διεθνωτικά ταμεία. Δεν εξαρτάται από εμά αυτό. Δεν μπορούμε να επισέλθουμε στη λεπτομέρεια των ε, διατάξεων και των κανόνων. Τέλος, θα δείτε ότι υπάρχουν κάποιες τροπολογίες Σαβαρή, ρακτικό και Κράμερ και Μπλόκλαντ. Είναι προσαρμογές του, που αφορούν το πρώτερο κείμενο και έχουμε τρεις προφορικές τροπολογίες που θα ήθελα να αποδεχθείτε που στην πραγματικότητα αποκαθιστούν σφάλματα του εισηγητού μια προφορική τροπολογία ιδιαίτερα που αφορά την παράγραφο 5 όπου εκεί αναφερόμουν στο ΣΥΒΙΤΑΣ 3 εξηγώντα ότι θα πρέπει να διευρυνθεί το πρόγραμμα Σιβητάς που πάει ήδη πολύ καλά και ήδη υπάρχει μια πρωτοβουλία να δώσουν περισσότερα μέσα και να ανοίξουμε λίγο περισσότερο το πεδίο όσον αφορά την καινοτομία. Αλλά εφόσον υπάρχει ήδη το Σιβητάς 3, ο, ο εισηγητής διορθώνει και ζητά να δεχτείτε αυτή την προφορική τροπολογία που θα αναφέρεται, μια νέα, θα αναφέρεται σε μια νέα γενιά Σιβητάς, το Σιβητάς 4, μετά στην παράγραφο 7 Εδάφιο 3. Είναι βάση τροπολογίας του κ. Μπλόκλαντ. Είναι προφορική τροπολογία. Έχει σαν στόχο να κάνει αντιληπτή την τροπολογία του κ. Μπλόκλαντ. Στα γαλλικά είχα μια εκδοχή που ήταν ε, δυσνόητη. Είναι μια τροπολογία που αφορά το λεξιλόγιο και το εύληπτον του κειμένου. Και μετά υπάρχει και μια τελευταία προφορική τροπολογία. Αυτή θέλει να λύσει ένα πρόβλημα που δημιούργησα. Μίλησα για ευρωπαϊκέ κρατικές, ευρωπαϊκές κρατικές ενισχύσεις, είναι κρατικές ενισχύσεις και η Ευρώπη δεν είναι κράτος. Δεν μπορούν να είναι ευρωπαϊκή κρατική ενίσχυση. Μιλάω για ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, είτε πρόκειται για επιδοτήσεις, φεντέρ κλπ. Και, και εκεί παρακαλώ να το διορθώσετε, δεν αλλάζει η ουσία του κειμένου. Αυτά αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά μπορώ να σας πω. Ε, ζητώ συγγνώμη μακρηγόρησα, περιμένω να ακούσω σχόλιά σας και μπορώ να σας απαντήσω επισκεκριμένων τροπολογιών μετά αυτή τη συζήτηση. κυρία Ζόμερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είπατε μόλις ότι οι τροπολογίες ε, Φέρμπερ, ε, Γκέγκλερ και δικές μου δεν ε, επιτρέπουν πιο ανοιχτό χαρακτήρα σε σχέση με τις δικές σας. Αντιθέτως, ε, κύριε Σαβαρή, εσείς δεν επιτυκνύετε ανοιχτό πνεύμα για τις τροπολογίες μας. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Με εκνευρίζει αυτό που συμφωνήθηκε για την τοποθέτηση μεταξύ του σχεδίου, για το σχέδιο αυτό, μεταξύ του εισηγητή και του σκιώδου εισηγητή. Δεν είναι εφικτό αυτό. Μας είπατε ότι αυτά είναι και δεν το συζητάμε. Ένα θέμα μόνο μπορούμε να προσθέσουμε, δεν δεχόμαστε τροπολογίες κτλ. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά μη δημοκρατικός αυτός ο τρόπος εργασίας. Και φυσικά θα συνεχίσω να διακηρύττω την απόψή μου και να υποστηρίζω και τις τροπολογίες μου και σίγουρα θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με το θέμα αυτό στην επόμενη θητεία. Αρκετά θέματα δεν με βρίσκουν σύμφωνοι στην έκθεση αυτή για ενδεχόμενο σχέδιο δράσης. Αυτό που ασφαλώς είναι θετικό είναι ότι όλοι πλέον ε, αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να λεφθεί υπόψη η αρχή της επικουρικότητας. Δεν είμαστε φυσικά αρμόδιοι ως Ευρωπαίος νομοθέτης για τη ρύθμιση των ε, εσωτερικών ζητημάτων παρά το γεγονός ότι ο Επίτροπος Μπαρό το έπλασε αυτό. Αλλά στη τελική ανάλυση ο 80% του κόσμου ζει σε πόλεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται και η όλη συζήτηση για το κλίμα και οι άνθρωποι α, στις πόλεις ε, οδηγούν αυτοκίνητα, άρα θα αναλάβουμε και εμείς αυτή την αρμοδιότητα. Αυτή ήταν η επιχειρηματολογία. Δεν ισχύει φυσικά κάτι τέτοιο αλλά φυσικά και μπορούμε να υποστηρίξουμε την συλλογή βέλτιστων πρακτικών για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό που με ανησυχεί παρόλα αυτά είναι η ίδρυση ενδεχομένω επιπλέον κονδυλίου για τη χρηματοδότηση πιο φωλικών μεταφορών προς το περιβάλλον στις πόλεις. Φυσικά χρειαζόμαστε φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές σε άλλες πόλεις και καταλαβαίνω ότι Υπάρχουν και μεγάλα ελλείμματα σε πολλές ε, πόλεις, αλλά δεν είναι δυνατόν ασφαλώς να δημιουργούνται νέα χρηματοδοτικά όργανα και τα κράτη-μήλη εκείνα τα οποία επέδειξαν επιμέλεια και επί δεκαετίες επένδυσαν σε φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές, θα πρέπει τώρα δηλαδή, να πληρώσουν για τα άλλα κράτη-μέλη. Αγαπητοί φίλοι, με όλο το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης και ενότητας που θέλω να επιδείξω. Αν θέλουμε να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία. Και με τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να τεθούν οι ανάλογες προτεραιότητες από τα κράτη-μέλη τα οποία είναι πιο πίσω γιατί άλλωστε τα διευθυντικά ταμεία προς τα νέα κρατημέλη κυρίως ε, αφιερώνονται. Και νομίζω ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές. Αυτό που δεν κατάλαβα καν είναι η κάρτα χρήστη για την αστική μεταφορά, για τις αστικές μεταφορές. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και το βρίσκω και ανόητο. γιατί και εγώ από την ε, δημοτική πολιτική προέρχομαι και ασχολήθηκα πολύ καιρό σε αυτό το επίπεδο. Αλλά πραγματικά αυτή η κάρτα χρήστη δεν καταλαβαίνω τι σκοπό εξυπηρετεί. Κάτι άλλο παρατήρηση για τις ε, αστικές μεταφορές αγαπητοί φίλοι. Αυτό πραγματικά παραπάει γιατί συνεπάγεται τεράστιο γραφειοκρατικό άχθος και τεράστιο κόστος στις Βρυξέλλες. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι κάτι το οποίο το επιθυμούμε. Πρόκειται για έργο το οποίο θα πρέπει να επιτελέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί δηλαδή να δημιουργηθεί ξεχωριστό παρατηρητήριο. Και δεν καταλαβαίνω γιατί ο εισηγητής δεν υποστηρίζει την τροπολογία μου για την ενίσχυση της έρευνας σε ό,τι αφορά την κατανομή των αγαθών στις πόλεις. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις και ιδέες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις αστικές περιοχές με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού, σε ό,τι αφορά τη λιανική κατανομή των προϊόντων. Γιατί να μην συνεχίσουμε και να μην ενισχύσουμε, να μην υποστηρίξουμε τις έρευνες προς την κατεύθυνση αυτή και θεωρώ γενικά ότι οι πόλεις είναι σημαντικές ε, οικονομικές αιστείες και θα πρέπει να παραμείνουν σημαντικές οικονομικές αιστείες. Άρα θα πρέπει να επιτρέπει ένα ποσοστό των μετακινήσεων και σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των ιδιωτών, σε ό,τι αφορά τη μηχανική μεταφορά των ιδιωτών, ούτε αυτό το δέχεστε οι Γιατί? Είμαι κατά της ε, πλήρους κατάργησης των γεωταχή στις πόλεις. Γιατί αυτό δεν θα βελτίωνε, δεν θα ανταποκρινόταν στις δημογραφικές κανονάγκες στις σημερινές. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή τη, δημογραφική, τη δημογραφική αυτή αλλαγή και σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις στις πόλεις, γιατί οι πιο ηλικιωμένοι συνήθως έχουν προβλήματα κινητικότητας και άρα συχνά ε, επιλέγουν να μένουν στις πόλεις όπου έχουν καλή πρόσβαση στις μεταφορές, στα ψώνια, αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζονται και το αυτοκίνητό τους. Γιατί να μην το αναφέρουμε λοιπόν αυτό σε ό,τι αφορά θέματα κινητικότητας της πόλης. Η δημογραφική λοιπόν αλλαγή είναι κάτι το οποίο σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να αναφερθεί. Νομίζω ότι αρκετά μίλησα. Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά από τα σχόλιά μου. Ευχαριστούμε κύριε Σόμερ. Το λόγο έχει ο κύριος Κράμερ. Πρόεδρε. Ω εισηγητή συνήθω λέει κανείς, ε, θέλει κανεί ε, να μιλήσει πιο πολύ, αλλά συνήθως τον διακόπτει ο πρόεδρο, αλλά αυτό το πρόβλημα το έχετε εσεί άλλωστε, γιατί είσαστε και πρόεδρο και εισηγητής ο ανοιχτός χαρακτήρας στον οποίο επικρίνεται ότι λείπει. Φυσικά έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε κάθε τροπολογία, αλλά ξέρουμε ότι μεταξύ πρασίνων και συντηρητικών σε ό,τι αφορά θέματα μεταφορών και αστικής πολιτικής υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Τι είπα, τι είπα λέτε? Εκτός μικροφώνου τα σχόλια. Α, πώς το λέμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λέμε και χριστιανό ναι, συγχωρέστε με, συγχωρέστε με. Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό, για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ε, υπάρχει μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά τέτοια θέματα από τους πράσινους. Και μιλήσατε και για την ε, μηχανική μεταφορά των ιδιωτών και για τη δημογραφική αλλαγή. Αν ε, σας απασχολεί η δημογραφική αλλαγή, θα πρέπει να υποστηρίξετε πολύ την έκθεση αυτή, γιατί διαπιστώνουμε ότι στη Γερμανία το 20% των οικοκυριών δεν διαθέτει αυτοκίνητο, αλλά το 80% των οικοκυριών πάνω από τα 65 ετών δεν έχει αυτοκίνητο. Δηλαδή, εξετάζοντας το πώς εξελίσσεται δημογραφικά η κοινωνία, προκύπτει ότι οι ηλικιωμένοι χρησιμοποιούν τα δημόσια μέσα συγκοινωνιών. Και Να σα αναφέρω και το παράδειγμα τη Ολλανδέζα γιαγιά, η οποία επισκέπτεται την κόρη τη με το ποδήλατο και τη λέει ευτυχώ γιατί δεν θα μπορούσε να έρθει με τα πόδια. Αυτή λοιπόν είναι η γενικότερη τάση και θα πρέπει να την υποστηρίξετε. Το δεύτερο το οποίο θέλω να υποστηρίξω σε ό,τι αφορά το ότι είπε ο Πρόεδρος, φυσικά και η Βενετία διαφέρει από τη Βερολίνο. Όντως, ναι, ναι, ναι. Στο Βερολίνο όμως, ακόμη και αν το πιστεύετε, έχουμε πιο πολλέ γέφυρε από τη Βενετία. Είπατε ότι δεν θέλετε να περιορίσετε, να... Σας πω όμως κυρία Ζόμερ ότι υποστηρίξετε περιπαθώς την επικουρικότητα. Δηλαδή όλα όσα αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ισχύουν και στις πόλεις, όπως για παράδειγμα χώρο χώρος ανάπαυσης ή η Ευρωπαϊκή Άδεια Οδήγηση. Όλα αυτά ισχύουν και για τις πόλεις. Ε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι, κοιτάξτε, στι διάφορες πόλεις αυτά δεν ισχύουν. Και να σας αναφέρω και ένα γερμανικό παράδειγμα. Οι δήμοι, για παράδειγμα, θα πρέπει να υποστηριχθούν όταν δημιουργούνται νέα τραμ, αλλά μόνο εφόσον έχουν μία τροχιά. Άρα στο Στρασβούργο, για παράδειγμα, δεν μπορούν ε, να υποστηριχθούν το 80% των τραμ. Τι έγινε τελικά? Βάλαν το τραμ κάτω από το έδαφος προκειμένου να έχουν πιο πολύ χώρο τα αυτοκίνητα και ανακοίνωσαν ότι πρόκειται για ένα μέτρο φιλικό προς το περιβάλλον. Όχι, όχι, στο διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Αν αυτή είναι η δικαιολογία σας, και η επιχειρηματολογία σας να συνεχίσετε. Αλλά εγώ έχω κι άλλα και καλύτερα μάλιστα μέτρα να προτείνω για τον εισηγητή τώρα. Είπατε ότι θέλετε να προκάνετε οποιαδήποτε προδιαγραφές, ότι ισχύει το tempo 30, μάλλον συγγνώμη ταχύτητα, τώρα ταχύτητα των 30 χιλιόμετρων και ότι επαφείτε στην, αρμο... στην επικουρικότητα. Νομίζω ότι πρέπει για κλασικό παράδειγμα επικουρικότητα, γιατί σε τελική ανάλυση οι πόλει αποφασίζουν που σε ποιου δρόμου μπορεί κανείς να οδηγήσει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Στο Βερολίνο το 75% των δρόμων ε, έχει όριο ταχύτητας τα 30 χιλιόμετρα. Αλλά και όλοι που διαμαρτύρονται και λένε ότι πράγματα πρέπει να παραπονηθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υποβάλουμε ενστάσεις. Όχι όμως όλα μπορούν να αλλάξουν, να εφαρμόσουμε αυτόν τον κανόνα. Τον κανόνα. Και γι' αυτό, κύριε Σιγητά, είπατε ότι από πλευράς φιλοσοφικής είσαστε υπέρ. Αλλά ωστόσο να μπορείτε να συμφωνήσετε σε πρακτικό επίπεδο με την τροπολογία αυτή. Να σας πω ότι και εγώ από, φιλοσοφικό, από φιλοσοφικής άποψης συμφωνώ, ίσως πρακτικά θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Και στη τελική ανάλυση, γιατί είναι τόσο σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί με τις αστικές μεταφορές. Είπατε ότι 80% των ε, ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν στις πόλεις και 70% των ε, ουσιών που ρηπαίνουν την ατμόσφαιρα προέρχονται από τις μεταφορές. Αλλά και εσείς ε, αποφασίσατε αυτό το τριπλό 20 μέχρι το 2020 20% ε, περιορισμό των αέριων λοιπόν, ρήπων και το καθεξής στα πλαίσια της γερμανικής προεδρίας. Η κυρία Μέρκελ τα αποφάσισε. Ωστόσο το εξής είναι σαφές. Αν θέλουμε να αλλάξουμε και να αντιστρέψουμε την αλλαγή του κλίματος, θα πρέπει να επέμβουμε στις πόλεις, γιατί από εκεί προέρχεται το 70% της ρήπανσης. Γι' αυτό υποστηρίζω τη γενικότερη κατεύθυνση και θα ήθελα να υποστηρίξω και τις τροπολογίες μου. Και θα χαιρόμουν αν δεχόσασταν αυτήν την τροπολογία για το όριο ταχύτητα των 30 χιλιόμετρων και την επικουρικότητα των ναι. πόλεων στο τομέα αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Κράμερ. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία σας. Το λόγο έχει ο κύριος Μπλόκλαντ. Ευχαριστώ πρόεδρα. Θα είμαι σε ό,τι αφορά την εκθέσή σας. Ε, με ικανοποιεί το αποτέλεσμα και η συνεργασία που είχαμε αναδρομικά θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε προσθέσει πιο πολλά στοιχεία για τις ιστορικές πλωτές μεταφορές, γιατί ο εισηγητής τώρα αναφέρει ένα πλήν ο εισηγητής στην τροπολογία υπαριθμών 30. Αλλά νομίζω ότι στην Ολομέλεια θα πρέπει να κάνουμε μια παρατήρηση ότι προτείνουμε να γίνει έρευνα για την υπεραξία των μεταφορών μέσα των πλωτών οδών για τον εξοπλισμό των πόλεων. Την προηγούμενη εβδομάδα διάβασα σε ένα περιοδικό στην Ολλανδία για τον εξοπλισμό της ε, πιο πυκνά κατοικημένης περιοχής της ε, Ολλανδίας σε ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής ε, πλωτής μεταφοράς. Νομίζω ότι είναι πολύ πετυχημένο το άρθρο αυτό και ελπίζω ο εισηγητής να συμφωνίζει μαζί μου για την συμπερίληψη αυτού του στοιχείου πριν από την Ολομέλη. Η έκθεση είναι εξαιρετική, αλλά την κάνουμε τέλεια με την προσθήκη αυτού του στοιχείου. Euh, Ευχαριστώ κύριο Σεράκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη που κατέθεσα καθυστερημένος για τη συζήτηση αυτή, αλλά η πολιτική για τις μεταφορές δεν μας βοηθά να τηρούμε τα χρονικά όρια και τις προθεσμίες μας. Λυπάμαι. Επί της ουσίας ε, είμαστε υπέρ της έκθεσης, όπως την παρουσίασε και ο εισηγητής και όπως προσπάθησε να τη διαμορφώσει. Είμαι βέβαιος ότι θα υποστηριχθεί από την ε, συντριπτική πλειοψηφία του Κοινοβουλίου και δικαίως, γιατί συνεργάστηκαν πάρα πολλές πλευρές για την κατάκτηση της έκθεσης. Να ευχαριστήσω τον Σκιώδη εισηγητή και τον εισηγητή. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό αποτέλεσμα μιας πολύ καλής συνεργασίας. Το γεγονός ότι υπήρξε μια έντονη συζήτηση είναι κάτι που με χαροποιεί. Το γεγονός ότι η συζήτηση αυτή ίσως επικεντρώθηκε υπερβολικά στη γερμανική κατάσταση, θεωρώ ότι οφείλεται στο γεγονός ότι στη Γερμανία περιμένουμε εκλογές... όχι μόνο ευρωεκλογές... αλλά και εθνικές εκλογές. Και αυτό φαίνεται ότι επισέρχεται ως στοιχείο και στη συζήτηση. Τρία θέματα ήθελα να αναφέρω μόνο. Επειδή η συνάδελφος Ζόμερ αναφέρθηκε και στον εξοπλισμό με προϊόντα. Είπε ο εισηγητής ότι όλοι συμφωνούμε και όλοι φροντίσαμε συνειδητά σε ό,τι αφορά τις εμπορευματικές μεταφορές και τον εξοπλισμό των πόλεων να θέσουμε υψηλά πρότυπα. Θεωρούμε ότι τα σούπερ μάρκετ, οι αγορές δεν πρέπει να περιοριστούν στο εξωτερικό των πόλεων, θα πρέπει να παραμείνουν ζωντανές οι πόλεις. Άκουσα και τον ε, διάλογο μεταξύ των συναδέλφων σε ό,τι αφορά τις μεταφορές των ιδιωτών. Δεν θέλουμε να καταργήσουμε ασφαλώς τις μεταφορές των ιδιωτών στις πόλεις, απλά θα πρέπει να φροντίσουμε να διαμορφωθεί με το σωστό τρόπο. Θα πρέπει να αναζητήσουμε ολοκληρωμένες λύσεις και να τις βρούμε, ελπίζουμε. Και χρειαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή κοινέ προσπάθειες. Τέθηκε και το θέμα της έρευνας για το παρατηρητήριο επικρατεί η ανησυχία. Το θίγει άλλωστε και ο εισηγητής στο κείμενό του ότι δεν θέλουμε να προσθέσουμε γραφειοκρατία, απλά θέλουμε να φροντίσουμε να ασχοληθούν οι αρμόδιοι φορείς επαρκώς με τους ε, όρους που προκύπτουν από την έρευνα για το θέμα αυτό. Εκ μέρους λοιπόν του ΕΛΚ πρέπει να σας πω ότι και μας μας απασχολεί να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει επιπρόσθετη γραφειοκρατία στο θέμα αυτό. Τελευταίο στοιχείο. Επειδή επί δεκαετίες δεν ήταν δούριος ύπος, αλλά τέλος πάντων πρόκειται για ένα άλλο μέσο μεταφοράς που απασχολεί τον κύριο Κράμερ. Όχι, όχι, για το, τα 30 χιλιόμετρα. Το θέμα εδώ είναι, και αυτό το υπογραμμίζω επειδή είναι πολύ σημαντικό, τα παρουσιάζονται τα πράγματα, λες και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λες και θα ήταν ελάφρυνση για τους δήμους, για τις πόλεις και σε καμία περίπτωση παρέμβαση σε ό,τι αφορά τον κανονισμό της επικουρικότητας αν επιβληθεί ευρωπαϊκά όρια ταχύτητας. Ε, θεωρητικά έχει δίκιο. Φυσικά κάθε δήμος μπορεί να πει ότι θέλω στον τάδε ή να να υπάρχει πιο υψηλό όριο ταχύτητας. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει το πρόβλημα. Ότι οι πόλεις θα θεωρήσουν ότι έχουν καπελωθεί από την Ευρώπη. Γιατί αυτέ οι ρυθμίσεις, κύριε Κράμαρ, έχουν προκύψει από κάτω προς τα πάνω και θα πρέπει, θεωρώ, να αφήσουμε την κατάσταση όσο έχει. Χαίρομαι που έγινε τόσο ζωηρή συζήτηση και έτσι ακούστηκαν όλες οι πλευρές στη συζήτηση αυτή. Είναι ωραίο να συζητούμε και θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι υπάρχουν διαφορές απόψεων και ότι τελικά θα επικρατήσει η πλειοψηφία. Εσείς θέλετε να αποφασίσετε εσείς ο ίδιος και καλά κάνετε και προασπίζετε την θέση αυτή σε τοπικό επίπεδο. Ελπίζω όμως η έκθεση αυτή να τύχει της υποστήριξης της πλειοψηφίας προκειμένου να αποστείλουμε και ένα καλό μήνυμα υπέρ μιας διαδικασίας η οποία έχει πάει αρκετά καλά και θα είχε πάει ακόμα καλύτερα αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πραγματοποιήσει την αρχική της πρόθεση και είχε αποφασίσει εγκαίρως, είχε υποβάλει εγκαίρως την πρότασή της. Θα αποτελούσε αυτό ένα πολύ καλύτερο μήνυμα από αυτό που προσπαθούμε τώρα να διαμορφώσουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ράκ και για την ομιλία σας, αλλά και για την αποφασιστική σας υποστήριξη, γιατί εσείς με τη δική σας έκθεση για την Πράσινη Βίβλο είχατε ανοίξει το δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Και ακριβώ επειδή δόθηκε συνέχεια με ένα σχέδιο δράσης αποφασίσαμε κάπως να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκριθεί και ελπίζω να το κάνει. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας συγχαρώ κύριε Πρόεδρε για την ε, τόλμη σας και την αποφασιστικότητά σας ε, στη μάχη αυτή που δίνετε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αστική κινητικότητα. Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αθέτησε την υπόσχεση που είχε κάνει στο ίδιο το πρόγραμμα εργασιών της. Γι' αυτό και σας συγχαίρω, κύριε Πρόεδρε, για την Ανδρία που δείξατε και για την ε, πρόταση αυτή προκειμένου να αποκρισταλώσει γνώμη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αστική κινητικότητα πριν τις ευρωεκλογέ. Θα ήθελα να επιμείνω σε τρία σημεία, ελπίζοντας ότι θα σας πείσω να τα λάβετε υπόψη. Σε ό,τι αφορά τα αστικά διόδια. Είναι σημαντικό αυτό το σημείο και όσοι μίλησαν για αυτό το θέμα τάχθηκαν υπέρ. Τάχθηκαν όχι μόνο υπέρ της μελέτης, αλλά και υπέρ των τροπολογιών που καλύπτουν αυτά τα σημεία. Εγώ δεν είμαι κατά των διοδίων στις πόλεις, αλλά πιστεύω ότι από άποψη διαφοράς της αστικής ανάπτυξης, αλλά και της κοινωνικής ανάπτυξης στις διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις και μητροπόλεις, γιατί πρόσφατα εγκρίναμε και μία έκθεση για την ε, αστιφιλία και την αστική ανάπτυξη στην Ισπανία. Υπάρχουν όμως κάποιες οικονομικές επιπτώσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και που καλύπτονται στη μελέτη. Γι' αυτό θα μπορούσατε να προσθέσετε στο κείμενό σας την τροπολογία 56, τη δική μου, γιατί ζητώ στη μελέτη αυτή για τα διόδια στις πόλεις να υπάρχει ειδικό εδάφιο για τον κοινωνικο-οικονομικό τους αντίκτυπο, δεδομένης της ε, ποικιλομορφίας του βαθμού αστικής ανάπτυξης στις διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Έχω πει πολλές φορές ότι στην ε, Ισπανία η αστιφιλή αυτή έχει εκδιώξει από το κέντρο της Ισπανίας ε, τους νέους, τις ε, πιο χαμηλά εισοδηματικές οικογένειες που Σπρώχνονται όλο προς τα έξω, προς τα προάστια, ενώ αναγκάζονται να επανέλθουν στο κέντρο για να εργαστούν. Σκεφτείτε τέτοιοι άνθρωποι που ούτως ή άλλως έχουν οικονομικά προβλήματα θα πρέπει να πληρώνουν και διόδια. Λοιπόν, σε αυτή τη μελέτη θα ήθελα να περιλάβουμε και τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο αυτών των διοδίων σε ομάδες ανθρώπων που εκδιώχθηκαν ουσιαστικά, αναγκάστηκαν να, να εγκαταλείψουν το κέντρο της πόλης. Επίσης, Συμφωνώ με την πρότασή σας για το κατευθυντήριο σχέδιο σε ό,τι αφορά τον προβληματισμό για τα αστικά κέντρα. Επίσης, ό,τι αφορά τα σχέδια αστικής ε, μετατόπισης. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συμπεριληφθούν ε, στο σχέδιο για τις αστικές συγκοινωνίες. Και επίσης, εντός των σχεδίων αυτών, να συμπεριλάβουμε και πολλά άλλα στοιχεία. Στην τροπολογία μου 47 ουσιαστικά σας υπενθυμίζω ότι αυτά τα σχέδια αστικής μετατόπισης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τη μετακίνηση και των εμπορευμάτων αλλά και των υπηρεσιών. Γιατί πολλές φορές μιλήσαμε για τη διανομή του ταχυδρομείου ή την παράδοση διαφόρων πακέτων δεν είναι κατά ανάγκη μεταφορά ή μετακίνηση εμπορευμάτων, αλλά μετακίνηση συγκεκριμένων υπηρεσιών. Σας παρακαλώ, λοιπόν να συμπεριλάβετε και την τροπολογία 47 στο κείμενο. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 14 για το Civitas Mundo, διμερώς είχαμε συζητήσει, μια και είναι πενιχρό το κονδύλιο της νέας γενιάς των Civitas, να προσπαθήσουμε να διευρύνουμε τις αρμοδιότητες ε, και τις εξουσίες του ΣΥΒΙΤΑΣ χωρίς ε, αύξηση της χρηματοδότησης. Αλλά ξαναδείτε την τροπολογία μου 14, γιατί εκεί προτείνω να συμπεριληφθεί το ΣΥΒΙΤΑΣ σε άλλες δημοσιονομικές γραμμές χρηματοδότησης, όπως είναι η συνεργασία της, για την ανάπτυξη ή η πολιτική γειτονία. Και αυτό είχαμε προτείνει στη συνεδρίαση της ε, του για την εκπνοή του υφισταμένου ΣΥΒΙΤΑΣ γιατί σε τέτοιου είδους αναπτυξιακές ε, πολιτικές και πολιτικές γειτονίας εφαρμόζονται κάποια σχέδια, αδιαφορώντας όμως ή χωρίς να γίνεται δέους εκμετάλλευση του κεκτημένου του Σύβητας και των πολλών θετικών του σημείων. Το λόγο έχει εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Νουκ Μαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι προβληματισμοί που διεξάγονται και ανταλλαγές απόψει που έλαβαν χώρα προετοιμάζοντα το εγγραφό μα για το μέλλον των μεταφορών καταδεικνύουν άριστα ότι οι στόχοι τη ε, πολιτική μεταφορών δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρί να διαφερθούμε για την αστική κινητικότητα. Η πράσινη βίβλος που δημοσίευσαμε το Φεβρουάριο δείχνει ότι θεωρούμε ότι αστικέ μεταφορέ αποτελούν το πρόσφατο τμήμα του Ευρωπαϊκού Σύστηματο Μεταφορών και Μάλιστα, η περισσότερη κυκλοφορία στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών ξεκινά και καταλήγει σε αστική ζώνη. Euh, δεν θα σχολιάσω τι τροπολογίε, διότι δεν υπάρχει πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα επαναλάβω τη δέσμευση που έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρο Ταγιάννη να αναπτυχθούν δραστηριότητε στον τομέα τη αστική κινητικότητα στο σεβασμό βέβαια της αρχής επικουρικότητας και να ένα σχέδιο δράσεως πλήρες σχετικά με την αστική κινητικότητα τους επόμενους μήνες. Αυτό το σχέδιο δράσεως θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο σε όλες τις δραστηριότητε που ήδη έχουμε δρομολογήσει και που θα συνεχίσουμε στον τομέα. Το σχέδιο εκθέσεώς σας είναι χρησιμότατο και είναι άλλη μια συνεισφορά στον προβληματισμό μας και καταδεικνύει τον πολύ ενεργό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σχετικό αυτό τομέα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Χότμαν. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή για να ολοκληρώσουμε και για να απαντήσει σε κάθε σημείο ξεχωριστά. Εγώ μου ο εισηγητής βέβαια. Λοιπόν που η κυρία Ζόμερ. Θα ήθελα να της απαντήσω παρόλα αυτά. Θα ήθελα να της πω ότι δέχομαι τις τροπολογίες 25, 6 και 10. Δεν απερίφθησαν όλες αυτές. Και δεύτερον, την καλώ στην Σύνοδο του Στρασβούργου σε μια συζήτηση ε, που εκπροσωπήθηκε μάλλον σε αυτή τη συνεδρία από την βοηθό Δεν μπορούσα να μην συζητήσω μαζί της, το έκανα και με την κυρία Γέγκλε και συνεργαστήκαμε στενά και με τον κύριο Ρακ θα με συγχωρήσει που κάλεσα την κυρία Ζόμερ σε μια συζήτηση που όμως δεν μπόρεσε να λάβει χώρα την περασμένη εβδομάδα. Όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό μέσο, το συμπληρωματικό, καταλαβαίνω ότι ίσως σχετικά με αυτό να υπάρχουν κάποιες, ε, κάποιοι δισταγμοί. Εγώ δεν είπα να δίνονται πίσω τα χρήματα από τον Ευρωπαϊκό προπολογισμό, εγώ έλεγα ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε το 2013-2020 τις προτεραιότητες του προπολογισμού. Δεν θα πρέπει να παραμείνουμε σε προπολογισμού τη δεκαετία του 80 και του 90, όταν έχουμε έσω προτεραιότητε όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα θέλω να προτείνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τον δεχόμενο υπάρξεω χρηματοδοτικού μέσου για τι αστικέ μεταφορέ, που θα είναι πάρα πολύ ευέλικτο μέσο. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θα μπορούσε να είναι, ένα νέο μεγάλο πρόγραμμα προτεραιότητα ή κάτι άλλο αυτό που συστήνει το Κοινοβούλιο είναι να δώσουμε κάποια κίνητρα στον τομέα των μεταφορών ε, να γίνουν κάποιες προτάσεις που είναι στατικής σημασίας. Ε, στο Μάρκο Πόλο, σε άλλου τομεί τη μεταφορέ κάνουμε κάτι. Θα πρέπει και εδώ συγκεκριμένο πλαίσιο να κάνουμε κάτι, σεβόμενοι πάντα την επικουρικότητα, αλλά ακολουθώντα μια προσέγγιση που δίνει κίνητρα. Ναι, τα διεθντικά ταμεία θα μπορούσαν να καλύψουν τι ανάγκε, αλλά χωρί τι σεζόνε όπω ξέρουν όλοι άρα δεν μπορούν να ικανοποιήσουν ισότιμα τις ανάγκες όλων των ευρωπαϊκών περιοχών και θεωρώ ότι το θέμα αυτό είναι ένα θέμα που ξεπερνά κάποια συγκεκριμένη περιοχή της Ευρώπης και είναι σχεδόν γενικό θέμα, καθολικό θέμα και χρειάζεται το ενδεδειγμένο εργαλείο στον τομέα αυτό. Ε, τώρα η χάρτα του Χρήστου δεν ξέρω τι είναι, δεν ξέρω τι ενόχλησε η κάρτα χρήστη στην έκθεσή μου. Εγώ δεν έχω εφεύρει κάτι τέτοιο, ευρωπαϊκή κάρτα χρήστη. Θα ήταν περίπλοκο, πάρα πολύ περίπλοκο κάτι τέτοιο. δεν ξέρω σε τι αναφέρεται όσον αφορά το παρατηρητήριο των αστικών μεταφορών, νομίζω ότι χρειάζεται, τουλάχιστον αυτό μου λένε όλοι οι επαγγελματίε του κλάδου, να υπάρχουν εναρμονισμένα και συγκρίσιμα στοιχεία σε έναν τομέα που είναι και τα λιγότερα στοιχεία και τα πιο αδύναμα ποιοτικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ε, συμπληρωματικός μηχανισμός, επιπρόσθετος. Μπορεί να ταθεί αυτό στη Eurostat ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, στη διατύπωσή μας ε, αποκλείουμε μια, ε, έναν φορέα που είναι ξεχωριστό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ μπορώ να ικανοποιήσω την κυρία Ζόμερ. Αν υπάρξει παρατηρητήριο θα πρέπει να υλοποιηθεί αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι από αλλοφορέ όσον αφορά την επιμελητία. Εγώ υποστηρίζω την τροπολογία 20 ε, και έχω βάλει και πρόσημο θετικό σαν εισηγητή στον κατάλογο ψηφοφορία. Και αντίθετα από αυτά που μα είπε, και Σόμερ, νομίζω ότι ε, ικανοποιούμε το αίτημά τη και αυτό διασκεδάζει και τι ανησυχίε τη κυρία Αγιάλα Σέντερ. Όσον αφορά τα αυτοκίνητα τη πόλη, δεν είμαι ότι υπέρ ούτε κατά. Δεν θέλω να φέρω συγκεκριμένου τρόπου μεταφορών μεγάλη απογοήτευση του Κράμερ, εγώ δεν θα πάρω πλευρές. Απλώς αρνήθηκα την τροπολογία 11 της κυρία Ζόμερ που λέει ότι θα πρέπει να παραμείνουν τα οχήματα στην πόλη διότι θεωρώ ότι αυτό είναι θέμα επικουρικότητας, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στον κύριο Παύλο Κώστα να ξαναβάλει στη Βενετία τα αυτοκίνητα όταν δεν υπάρχουν πλέον. Όσον αφορά τον κύριο Κράμερ, κύριε Κράμερ, εγώ τι να σας πω. Το έλεγε ο Ζρακ. Ε, επικίνδυνε και εκλογέ στη Γερμανία, οπότε αρχίζουν και ζεσταίνονται τα πράγματα. Γίνεται η προθέρμανση, έτσι κάνουν οι αθλητέ. Εγώ δεν είμαι υπέρμαχος του θέματος αυτού. Ήθελα να διευκρινίσω ότι η κυρία Λογιόλα Ντεπαλάθιο είχε αναφερθεί πρώτη σε αυτό. Ο κύριος Μπαρό ανακοίνωσε ένα σχέδιο δράσης όσον αφορά την αστική κινητικότητα. Ο κύριος Ρακ εδώ άνοιξε το δρόμο μέσω της εκθέσεώς του στην πρώτη ανάγνωση. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε πολύ πιο μεγαλύτερη υποστήριξη για το θέμα αυτό, διότι στα πλαίσια του κλίματος αυτό το θέμα που συζητούμε είναι κάτι που ξεπερνά τις πολιτικές διαιρέσεις. Όσον αφορά την περιοχή, τη ζώνη των 30 χιλιόμετρων την ώρα, θα σημειώσατε ότι στην τροπολογία μας υπαριθμών 54 είναι συλλογική τροπολογία αυτή. Ζητάμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση όσον αφορά τις ρυθιζόμενες ζώνες πρόσβασης αν αλλάξαμε την ορολογία, μιλούσαμε για αστικά διόδια. Δεν μιλάμε πλέον για αστικά διόδια, μιλάμε για ρυθμιζόμενη πρόσβαση σε κάποιες ζώνες. Αυτό μου προτάθηκε. Μου είπαν ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να μειώσουμε και να ελέγξουμε τη χρήση του αυτοκίνητου στο κέντρο της πόλης. Είναι οι ζώνες με 30 χιλιόμετρα την ώρα, οι απαγορεύσει, τα, τα διόδια, τα τέλη, Οπότε θα πρέπει να δούμε τι, δια... τι πολιτικές μπορούμε να εφαρμοστούν, τι συνέπειες έχουν διάφορες πολιτικές και συμφωνώ με την κυρία Γιάλα Σέντερ, είναι η ίδια απάντηση. Και νομίζω ότι καλύπτει πολύ ευέλικτη τροπολογία 54 όλες τις ανησυχίες. Ζητά έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βάζει τις εκθέσεις αυτής το επόμενο Κοινοβούλιο και η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσουν αν μπορούν να δρομολογηθούν κάποιες πρωτοβουλίες νομοθετικού περιεχομένου για να θες θεσπίζουν, να πλαισιώσουν αυτού αυτά τα τέλη κλπ. Να δούμε τι είναι η απαγορεύσει, οι ζώνε με 30 χιλιόμετρα την ώρα, ποια εργαλεία είναι τα πιο αποτελεσματικά. Υπάρχει ολόκληρη φαρέτρα μέτρων. Όσον αφορά τον κύριο Μπλόκλαντ, να το δω για την Ολομέλεια. Αναφερθήκατε στι ποτάμιε μεταφορέ. Θα πρέπει το κείμενο να έχει κάποια εμβέλεια ευρωπαϊκή, κύριε Μπλόκλαντ, βλέπετε. Θα έχουμε κάποια προβλήματα να αναφέρουμε τι ποτάμιε μεταφορέ τι γίνεται για διάφορε περιοχέ της Ευρώπης που δεν υπάρχει. Ε, διαφέρει κάθε περιοχή. Ιδού, αυτά μπορώ να σα πω για την κυρία Γιάλα Σέντερ, να τη επιβεβαιώσω ότι η 56 τροπολογία τη θεωρώ ότι είναι συμβατή πλήρω, συνάδει με τι τροπολογίε μα, θα γίνει αποδεκτή. Όσον αφορά την επιμελητία, την οργάνωση, στο σχέδιο με, έχουμε ε, τέτοιο, αναφερόμαστε ε, στις υπηρεσίες, τα εμπορεύματα κλπ. Μπορεί να ενταχθεί εκεί, μπορούμε να το εξετάσουμε το θέμα δεν αντελήφθη τι θέλετε να πείτε με τι υπηρεσίε, αλλά επειδή μιλώ για επιμελητία και υπηρεσίε, θεωρείτε ότι είναι στα πέσει επιμελητία και τα ταχυδρομεία, νομίζω ότι καλύπτεται. Όσον αφορά το Civitas Μούντο, εγώ δεν κατάλαβα την τροπολογία σα, αλλά είμαι έτοιμο να δεχτώ τυχόν προφορική τροπολογία, να με εξηγήσετε όμω, να μας πείτε ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια χρηματοδότηση και τι είδου εν ονόματι της πολιτικής ανάπτυξης και όχι εν ονόματι της πολιτικής των μεταφορών. Χρειαζόμαστε, ε, ζητάμε πολλά για, την, ε, για τις μεταφορές. Λοιπόν, απλά κάνω αυτή τη διευκρίνηση για αυτό που ζητάτε. Αυτά μπορώ να σας απαντήσω. Ευχαριστώ την κυρία Χότμαν που απέτησε φόρο τιμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απ' την άλλη θα της πω ότι περιμένουμε πολλά, θα περιμένουμε πολλά μετά από τις ψηφοφορίες στο Κοινοβούλιο, θα περιμένουμε μια πρωτοβουλία ορατή, ενθαρρυντική από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να σας πω εξάλλου ότι από τότε που αναλάβαμε αυτή την πρωτοβουλία, το κέντρο βάρους των επαγγελματιών του τομέα μετακινήθηκε προς εμάς, έρχονται σε επαφή μαζί μας, μας ζητάνε πράγματα. Και το λέω στους συναδέλφους, στους Γερμανούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, συνάντησα οργανισμούς, οργανώσεις των, της τοπικής Γερμανία, Γερμανίας, την Eurocities, ε, πόλεις κλπ. Όλοι είναι υπέρ και έχουν προσδοκίες. Και ο κύριος Ράκ το υπερασπίστηκε αυτό. Είναι καλύτερα τέτοιε πρωτοβουλίες κάπως ξεχωριστές να ξεκινάνε ξεχωριστά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι καλό να ξεκινάνε γιατί είναι πολλά τα διακυβευόμενα και στέλνω και ένα μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα απαντήσετε τώρα, διότι είναι πολιτικό το επίπεδο πριν δοθεί απάντηση. Εάν κάνει, ανοίξει δρόμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δείξει το δρόμο, θα πρέπει να αρπάξει την ευκαιρία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι ο στόχο μα. Να στρέψετε την πολιτική μας βούληση σε σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά θέλω να πω όσον αφορά αυτά τα θέματα και σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή τη νέα μέθοδο επεξεργασίας ενός κοινοβουλευτικού κειμένου. Θα ήθελα κλείνοντας, κλείνοντας να δώσω το λόγο στον κύριο Ντίσον για την έκθεσή του για τους διαδρόμους των εμπορευμάτων που είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα... να ζητήσω κι εγώ συγγνώμη γιατί έφτασα καθυστερημένα στη συνεδρίαση. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις ηγητές για την ε, αγαστή συνεργασία που είχαμε και επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που με βοήθησαν να τροποποιήσω χάρη στις τροπολογίες του στην έκθεσή μου. Κατατέθηκαν πάνω από 230 τροπολογίες στην ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάτι που δείχνει το πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα και πόσο τεράστιος είναι ο αντικτυπός του. Οι σκιώδεις ηγητές σε μία απόπειρα ανέβρεση συμβιβαστικής λύσης καθοδηγήθηκαν από τις ακόλουθες αρχές οι οποίες διατυπώθηκαν ήδη στην αρχή των διαπραγματεύσεων. Καταρχήν προσπαθήσαμε να ελαχιστοποιήσουμε κάθε πιθανή σύγκρουση μεταξύ σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων. Δεύτερον, Προσπαθήσαμε να πλουστεύσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να μειώσουμε και τη γραφειοκρατία που θα συνεπέφερε η εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Επίσης προσπαθήσαμε να διαφυλάξουμε την ισορροπία μεταξύ των κοινοτικών συμφερόντων αφενός και των εθνικών συμφερόντων αφετέρου. Ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να διαφυλάξουμε την ισορροπία μεταξύ των εκπροσώπων των υποδομών, των ε, διαχειριστών των υποδομών και των φορέων ε, και επιχειρήσεων σιδηροδρομικών μεταφορών. Ε, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε και κάποιο περιθώριο ελαστικότητας για την αντιμετώπιση περιπτώσεων κρίσης στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από τα άρθρα 11, 12 και 13 κυρίως. Και καταλήξαμε σε τρεις συμβαστικές τροπολογίες για τα προαναφερθέντα άρθρα. Οι τροπολογίες αυτές καλύπτουν μια, ένα μεγάλο αριθμό από τις υπόλοιπες τροπολογίες. Σε ό,τι αφορά τη συμβαστική τροπολογία για το άρθρο 11. προτείνουμε μια νέα διατύπωση με τον όρο των σιδηροδρομικών ε, χρόνων εφαρμογής των σλότς αντί για κατηγορίες προϊόντων. Έτσι, αποφεύγουμε να ορίσουμε ποια είναι τα εμπορεύματα που έχουν ευαισθησία ως προς το χρόνο μεταφοράς. Επίσης και για το σημείο 12 υποβάλαμε νέα διατύπωση για την κατανομή αυτών των ε, χρονικών περίοδων, των σλότ. Η πρόταση αυτή προβλέπει τη δυνατότητα κράτησης κάποιας ε, πρόσθετης δυνατότητας και τη αξιολόγηση της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων. Επίσης, με την πρόταση αυτή μειώνεται η αρχική προθεσμία των τριών μηνών σε ένα μήνα, προβλέποντας και εδώ κάποια ελαστικότητα. Η τελευταία τροπολογία αφορά το άρθρο 14. Συμβαστική τροπολογία. Χάρη στην συμβαστική αυτή τροπολογία θεσπίζουμε κάποιους, κάποιους κανόνες για την κατα, κατά προτεραιότητα κατακύρωση σλότ. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε δύο ακόμη τροπολογίες Ελάχιστη συζήτηση έγινε για την ε, θέση των επιχειρήσεων ε, σιδηροδρομικών μεταφορών στα, στους διοικητικούς φορείς. Τελικά καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι φορείς αυτοί θα πρέπει να εκπροσωπούνται στα διοικητικά σώματα, αλλά δεν θα πρέπει ταυτόχρονα να έχουν δικαίωμα συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Ο ρόλος τους θα είναι συμβουλευτικός. Θα δίνονται δηλαδή να παρακολουθούν τις ε, συνεδριάσεις των διοικητικών οργάνων. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία της κυρίας Γιάκοψ. Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει ότι οι υπάρχουσες υποδομές για τη μεταφορά των εμπορευμάτων διατηρούνται. Πρόκειται για τις τροπολογίες 1, ε, 2 και 3. Σε αυτά τα συμπεράσματα καταλήξαμε μετά από συζήτηση με τους σκιώδεις ηγητές, ε, τους οποίους ευχαριστώ και πάλι θερμά για τη συνεργασία. Merci beaucoup, pardon. ευχαριστούμε κυρία Ντουχόν. Το λόγο έχει η κυρία Τζάκοψ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή συνεργασία που ε, είχαμε. Ήταν ανοιχτός και για τις προτάσεις μας και για διαπραγματεύσεις. Υποστηρίζουμε τελικά τις ε, συμβαστικές προτάσεις οι οποίες προέκυψαν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και είναι σημαντικό να ενισχυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το πρόγραμμα αυτό. Και θα πρέπει σκληρά να εργαστούμε για τις καλές συνδέσεις, την διαλειτουργικότητα, την διαφάνεια, την ανταγωνιστικότητα, την φιλικότητα προς τον πελάτη των συστημάτων και σε πολλά άλλα θέματα. Αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους για το 2020, θα πρέπει να ενισχύσουμε τις ε, μεταφορές μέσω συνδροδρόμων. Είναι απαραίτητο αυτό. για να αναφέρουμε τα ποια είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία στην πρόταση αυτή. Καταρχάς, στον προτινόμενο κανονισμό θεωρούμε ότι θα δοθεί προτεραιότητα στην ε, μεταφορά των προϊόντων. Δεν θέλουμε όμως να επιβάλλουμε σκληρούς κανονισμούς και να περιορίσουμε την μεταφορά των επιβατών. Θέλουμε να επιδείξουμε αναδιάδρομο ευελιξία για να διαπιστώνουμε ποια κατηγορία θα πρέπει να λαμβάνει προτεραιότητα και πότε σε περίπτωση καθυστερήσεων και αυτό θα πρέπει να κρίνεται αναπερίπτωση. Αυτό αποτελεί μια ρεαλιστική προσέγγιση που θα ωφελήσει και τη μεταφορά εμπορευμάτων αλλά και τη μεταφορά των επιβατών. Επίσης, δεν θα πρέπει να ορίσουμε δεσμευτικέ ε, ε, κατανομές των ικανοτήτων. Αυτό θα πρέπει να καθορίζεται αναδιάδρομο και πάλι. Γιατί το να ορίσουμε κάποια δεσμευτικά όρια ε, είναι πολύ περιοριστικό και θα οδηγήσει και σε ένσταση από τον κλάδο. Είμαστε υπέρ ε, του One Stop Shop, το οποίο καθιστά τις μεταφορές πιο διαφανείς. Θέλουμε επίσης κάποιες ε, τροπολογίες ανά διάδρομο. ό,τι αφορά το εκτελεστικό συμβούλιο, πρόκειται για μια ε, βέλτιστη πρακτική η οποία απέδειξε την αξία της ε, στη διαδρομή Γένοβα-Άμστερνταμ. Συμφωνούμε όμως με την προφορική τροπολογία του εισηγητή ότι προκειμένου να μην υπάρξει περιττή γραφειοκρατία θα πρέπει να εξεταστεί κατά περίπτωση αυτό. Και κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνο με τον εισηγητή. Προκειμένου να έχουμε εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα παρέχουν συμβουλές σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των διαδρόμων. Υπάρχουν πάρα πολλά λόμπι που δραστηριοποιούνται προς την κατεύθυνση αυτή για να επηρεάσουν την έκθεση αυτή, αλλά εμείς δεν πρέπει να τους αφήσουμε να επικρατήσουν. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε την πράσινη οδό προς το μέλλον γιατί το παρελθόν μας διδάσκει ότι διαφορετικά δεν έχουμε καμία ελπίδα. Αν θέλουμε να πάρουμε στα σοβαρά την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να προασπίσουμε αυτή την πράσινη οδό σε ό,τι αφορά τις μεταφορές σας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κυρία Γιάκοψ. Κύριε Κράμερ, έχετε το λόγο. Ναι, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την καλή συνεργασία. Mm. Και καταλήξαμε σε δύσκολα θέματα, σε συμβαστικές προτάσεις, σε δύσκολα θέματα όπου δεν συμφωνούσαμε. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι το βασικό θέμα της έκθεσης αυτής είναι ότι στο Ευρωπαϊκό Συνδρομικό Δίκτυο δεν πέρασε αυτός ο διαχωρισμός του διεκδοσιακού καθεστώτος ε, που ήθελαν αρχικά το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Και γι' αυτό υπάρχουν καταχρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να αποφευθούν. Είναι παράλογο όμως να ορίζουν οι επιχειρήσεις ότι θα κλείνουν για παράδειγμα κάποιες τροχές τις οποίες δεν χρησιμοποιούν και μάλιστα χωρίς κόστος. Και αυτό για λόγους ε, πολύ απλά παρεμπόδισης του ανταγωνισμού. Θέλουμε λοιπόν πλέον να χρησιμοποιήσουμε με τον βέλτιστο τρόπο τα δίκτυα. Θέλουμε τα δίκτυα αυτά να αξιοποιούνται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και επειδή δεν υπάρχει με συνεπιτρόπο αυτός ο διοκτησιακός διαχωρισμός και φυσικά θέλουμε τον βέλτιστο, τη βέλτιστη χρήση, γι' αυτό λοιπόν αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο και προσπαθήσαμε να επιλύσουμε το έθιξα και στην προηγούμενη, στην τελευταία συνάντησή μας στην ε, Γαλλία, για παράδειγμα, το SNCF καθορίζει πλήρως τις τροχές και τα slots και έχει κλείσει πολλά slots, πολλές τροχές ε, η SNCF, τα οποία δεν χρησιμοποιεί και δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και άλλοι. Αυτό τι σημαίνει στη Γαλλία ότι χάθηκε το 28% των εμπορευματικών μεταφορών και αυτό ίσως, ε, ενώ σε άλλες περιοχές μάλιστα αυξήθηκε η εμπορευματική μεταφορά κατά 40%. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα από άλλες χώρες, όχι μόνο στη Γαλλία, αυτά ισχύουν και στη Γερμανία και στην Ολλανδία και ούτε καθεξής. και εφόσον δεν υπάρχει διεκτησιακός ε, διαχωρισμός, γιατί να μπορούν οι γερμανικοί συνδρόμοι να κάνουν μεταφορές και για παράδειγμα και στην Ολλανδία. Ασφαλώς θέλουμε να συμμετέχουν και οι συνδρομικές εταιρείες να συμμετέχουν με την εμπειρία τους. Αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται από τις εταιρείε υποδομής. Αν υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός λοιπόν, δεν θα αντιμετωπίζαμε το πρόβλημα αυτό, γιατί φυσικά με τα slots ε, με τις χρονοφυρίτες αυτές, ε, αυτές αυτά τα slots κοστίζουν χρήματα. Δεν θα αντιμετωπίσαμε λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα και προς αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να κινηθούμε. Θα μπορούσαμε να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό αν γίνονταν κράτηση για παράδειγμα κάποιου σλότ και τελικά δεν χρησιμοποιούνταν να το έχανε η εταιρεία όπως γίνεται στις αερομεταφορές. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να επεκταθούν οι μεταφορές και για τα εμπορεύματα. Καταψηφίσαμε καταψηφίστηκε η έκθεση επειδή ε, ζητούσαμε προτεραιότητα για τα εμπορεύματα. Γι' αυτό τελικά προέκυψε αυτό, σε αυτή η ρύθμιση που είναι ευέλικτη και χρειαζόμαστε σίγουρα και αυτό το one-stop shop. Και εδώ σταματάω λοιπόν. Ευχαριστώ, λυπούμε αγαπητοί συνάδελφοι. Αλλά η διερμηνία σταματάει στις 18.30. Έχουμε ελάχιστο χρόνο. Παρακαλώ να είστε πολύ σύντομοι. Ο κύριος Σίμψον έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή και τους σκιώδη εισηγητή, τους για τη δουλειά που έκαναν. Εγώ ειλικρινά θα ήθελα αυτή η πρόταση να είναι λίγο πιο ριζοσπαστική, με περισσότερη επιρροή όσον αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων μέσω σιδηροδρόμου. Αλλά είμαι στη μειοψηφία, το αναγνωρίζω και η σιδηροδρομικός τομέα εν γέννη δεν είναι έτοιμος να αλλάξει την παλιά πρακτική, δίνοντας προτεραιότητα στα εμπορεύματα. Επιδιώκοντα συμβιβασμό, ενθαρρύνομαι διότι κάποιε εταιρείε των σιδηροδρόμων πιστεύουν ότι προχωρήσαν πολύ μακριά, άλλοι όχι αρκετά μακριά και άλλοι ότι θα έπρεπε να κάνουμε το ένα, το τάδε, το δίνα και το άλλο. σω αφού εξετάσουμε το συμβιβασμό, ίσω τελικά να έχουμε πετύχει τελικά τη σωστή ισορροπία. Τι απέρευσε. Σαφή διαφωνία εντό του τομέα των σιδηροδρόμων. Και αυτό δεν μα βοηθάει καθόλου. Και διονύζει την αντίληψη ότι οι σιδηρόδρομοι είναι πάρα πολύ συντηρητικοί, πολύ εθνικιστικοί και πολύ προστατευτικοί. Ναι, απ' τη μια είμαι δυσαρεστημένο, απογοητευμένο που δεν αρπάξαμε την ευκαιρία που μα δόθηκε να είμαστε πιο ρεσβαστικοί. Από την άλλη, εγώ πιστεύω ότι το 1% του κάτι είναι περισσότερο από 100% του 0 και το να πέφτει κανεί ε, ηρωικά μαχώμε στην πολιτική δεν είναι πάντα υποφέλε. Οπότε υποστηρίζω αυτά που είπε η συνάδελφος κυρία Γιάκοψ. Είναι ένα βήμα σωστή κατεύθυνση. Ελπίζω ότι θα είμαστε αρκετά ειλικρινεί να μην θεωρήσουμε ζωσπαστικό το αποτέλεσμα. Διότι τι είναι, είναι το status quo με λίγο μεγαλύτερη ευελιξία, μερικά ψυχουλάκια για τα εμπορεύματα που έπεσαν το τραπέζι και έδειξε τι δύναμη έχουν κάποιες εταιρείες επιβατικές σε εθνικό επίπεδο τελικά, οι ομάδες πίεσης. Ο κ. Κρέιμερ ξέρει ποιους εννοώ. Δεν θα τους κατονομάσω. Διάλογος εκτός μικροφώνου και θόρυβος. Λοιπόν, δεν έχουμε προ... διόδους προτεραιότητας για τα εμπορεύματα, έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά δεν βοηθά τη συνεννόηση των εταιριών σε δυσυνορικό επίπεδο. Και συμφωνώ με τον κύριο Κρέμερ είναι ότι εδώ έχουμε τα θεμελιώδη προβλήματα της συνδρόμων. Έλλειψη συνεργασίας. Έλλειψη επικοινωνίας. Οι σιδηροδρομικές εταιρείε δεν συνεννούνται μεταξύ τους. Κάτι πρέπει να γίνει, συμφωνώ. Συμφωνώ λοιπόν με τους συμβασμούς πρόεδρε, θα περιμένω για μερικά χρόνια από τώρα, από τούδε και στο εξή, για να δω τελικά τις βαστικές ιδέες για τους σιδηροδρόμους εφαρμόζονται, κυρίως για τα εμπορεύματα σιδηροδρόμους, αλλά ευχαριστώ τον εισηγητή και τους κοιόδης για τη δουλειά που έκαναν. Τουλάχιστον φτάσαμε σε μια θέση όπου οι περισσότεροι μπορούν να την υποστηρίξουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σίμψον. Ο κύριο Στόκμαν και η κυρία Γιάλα για βραχύτατες παρεμβάσεις. Also, Σας ευχαριστώ. Ευτυχώς ε, που οι σκιώτες, οι συγητές και οι καταφρά καταφέραν να καταλήξουν σε, σε σωστό συμβιβασμό. Για το One Stop Shop είναι γνωστή η απόψή μου. Είναι καλό το γεγονός ότι εδώ πέρα ε, προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία και όχι αυστηροί άκαμπτοι κανόνες και σε ό,τι αφορά το εκτελεστικό αυτό όργανο. Ωστόσο είναι κρίμα που δεν μπορούν να συναποφασίζουν και αυτοί και να συμμετέχουν. Να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν όντω οι διάδρομοι η Γερμανία, για παράδειγμα, έχει τρεις ε, διαδρόμους, δεν θα αρκούσαν και δύο. Και κατά δεύτερο, προέκυψε και ανέκυψε το θέμα των μεικτών μεταφορών. Για παράδειγμα, όταν η διαδρομή θα μπορούσε να ακολουθεί μια όχι τόσο πυκνά κατοικημένη περιοχή γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις ε, χαίρονται και οι περιφέρειες, γιατί αποτελεί και δυνατότητα ανάπτυξης. Μπορεί να οριστεί λοιπόν μια τέτοια διαδρομή σε εθνικό επίπεδο και χρειάζονται για παράδειγμα τρεις διάδρομοι, μήπως αρκούν δύο. Κατά τα άλλα υποστηρίζω την έκθεση και θεωρώ ότι θα πρέπει να περάσει για να πετύχουμε κάτι όντως. Ευχαριστώ, Ινιές Αγιάλα Εντάχει κύριε Πρόεδρε γιατί τα θέματα της ουσίας δεν καλύφθηκαν. Ουσιαστικά δεχόμαστε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα ως προς τα ουσιαστικά θέματα. Αλλά στην τροπολογία 94, τη δική μου κυρία Σιγητά, υπάρχουν δύο τμήματα. Το πρώτο αφορά το θέμα του δυναμικού. Ξέρω, έχουμε διαφορετικές απόψεις, τι να σας πω γι' αυτό αλλά σε ό,τι αφορά την ε, σύσταση ή την τροποποίηση του διαδρόμου εμπορευμάτων, πρότεινα μετά από διαβούλευση των χρηστών και πελατών ε, των εμπορευματικών μεταφορών ε, μέσω σιδηροδρόμων. Γιατί όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη δική σας πρόταση, δεν φαίνεται να γίνεται καμία μνήα των χρηστών, των πελατών. Αναφέρονται μόνο οι διαχειριστές. Κύριε Ντούχον, παρακαλώ, λάβετε υπόψη και τη διαβούλευση με τους χρήστες και τους πελάτες, γιατί οι σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων δεν περιορίζονται μόνο στους διαχειριστές των υποδομών. Σας ευχαριστώ κυρία Γιάλα. Το λόγο έχει ο κύριος Πασκουαρέλη, εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, εκλυπαρώντας το να είναι εξαιρετικά λακωνικό ε, και ζητώ μια μικρή χρονική παράταση και από του ε, διερμηνεί. Μια και μόνο μια γλώσσα μπορώ να μιλάω κάθε φορά. Θα συμπυκνώσω την παρέμβασή μου για να τελειώσουμε γρήγορα. Συμφωνώ με το στόχο της πρότασης που είναι η θέσπιση νομικών και διοικητικών μέτρων ώστε η διάδραμη εμπορευμάτων που ζητάει ο κλάδος των σιδηροδρόμων να γίνει επιτέλους πραγματικότητα και όχι να παραμείνει στα χαρτιά και να είχαμε το ERTMS, το Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας και πολλά χρήσιμα συστήματα που όμως ήταν ανεπαρκή. Με βάση αυτές τις βάσεις όμως θέλουμε μία ανταγωνιστική προσφορά υπηρεσιών σε σχέση με τις υπόλοιπες μεταφορές. Κύριε Στόκμαν, με βάση την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια χώρα σαν τη Γερμανία, δεδομένου του όγκου εμπορευματικών μεταφορών που ε, διακινούνται ετησίως από, τα σιδηροδρομικά, από τις σιδηροδρομικές μεταφορές, θα χρειάζονταν τρεις διάδρομοι, κάτι που θα είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί, δεδομένο και των διαδρόμων του συστήματο διαχείρισης σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο Μεταφορών, εκεί έγινε πολύ σφοδρή συζήτηση για την οδηγία περί Ευρωβινιέτα. γιατί υπάρχει πρόοδο, αλλά είναι πολύ αργή και επίπονη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετάχθηκε υπέρ μια ισορροπημένη και υγιούς ε, ανταγωνιστικότητας διατροπική, που προποθέτει όχι μόνο μια πολιτική χρέωση των υποδομών με βάση την το πραγματικό κόστος των μεταφορών, αλλά χρειάζεται και μία ουσιαστική βελτίωση της προσφοράς των υπηρεσιών σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα απορρόφηση των αποδομών, όσο και την ποιότητα, δηλαδή ακρίβεια, αξιοπιστία, ταχύτητα και ούτω καθεξής. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκάλεσε εκτεταμένες συζητήσεις και ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή τον κύριο Ντούχον για το εμπεριστατωμένο του έργο. Η έκθεση είναι αρκετά κριτική, επικριτική. Οι συμβαστικές όμως τροπολογίες που συντάχθηκαν προτείνουν αρκετά παρα παραδεκτές λύσεις ε, και πιστεύω ότι ελπίζω μάλλον θα τύχουν υποστήριξης στην Επιτροπή Μεταφορών. Ομαδοποίησα τις τροπολογίες αυτές σε τέσσερις κατηγορίες. Καταρχήν διαχείριση των διαδρόμων. Αυτό είναι κέριο σημείο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί αυτό έλειπε μέχρι στιγμής από την πραγματοποίηση των διαδρόμων. Δυνατότητα συντονισμού μεταξύ των φορέων διαχείρισης, προκειμένου να επιτελεστεί κοινό έργο. Θα πρέπει λοιπόν να δοθούν κίνητρα για συνεργασία μεταξύ των διαφόρων διαχειριστών υποδομών. Επίσης, πέραν του θεσμικού ρόλου, θα πρέπει στο έργο αυτό να συμμετέχουν οι συνδεδομικές επιχειρήσεις, οι χρήστες δηλαδή του δικτύου. Με συστηματικό τρόπο μάλιστα, ε, φυσικά διασφαλίζοντας οι διαχειριστές των υποδομών την ανεξαρτησία της λήψης αποφάσεων. Προσπαθήσαμε λοιπόν να αναγνωρίσουμε τον αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων με την ανάγκη ευρεία συμμετοχής στην προετοιμασία των αποφάσεων. Και σίγουρα μετά την απελευθέρωση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οργανισμό διαχείρισης δεν μπορεί να δίνει προνόμια στον α ή β φορέα. Όλοι οι φορεί καλούνται να χρησιμοποιήσουν τους προκαθορισμένου διαδρόμους. Δεύτερη κατηγορία τροπολογιών αφορά την ε, κατακύρωση του δυναμικού των σλότ κατά την έναρξη της περίοδου για τα ετήσια ή εποχιακά ωράρια. Αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με το στόχο αναβάθμιση ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών, θα πρέπει να δώσουμε περισσότερα χέγγια στι μεταφορέ αυτέ, εξασφαλίζοντα όμω και την κατάλληλη ελαστικότητα προς τον διαχειριστή των υποδομών που θα προσαρμόσει αυτή την επικύρωση, κατακύρωση των, των δυνατοτήτων στις, ιδιαίτερες, ή στις ιδιαιτερότητες κάθε μεταφοράς εμπορευμάτων. Και εκεί υπάρχουν διαφορετικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τους διαδρόμους και για τις ε, υποδομές. Και εδώ νομίζω ότι η συμβαστική τροπολογία είναι πολύ καλή και μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Τρίτο θέμα αφορά τις προτεραιότητες σε περίπτωση διαταραχών. Και εκεί η συμβαστική τροπολογία του εισηγητού και των σχεδόν εισηγητών είναι πολύ χρήσιμη. Θα πρέπει όμως να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι δεν πρόκειται για κανονισμό του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου που θα θεσπίσει τις προτεραιότητες. Χρειαζόμαστε ένα κανονισμό ώστε οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι να καθορίζουν αυτές τις προτεραιότητες. Χρειαζόμαστε ένα νομικό πλαίσιο που προβλέπει την υποχρέωση θέσπισης προτεραιοτήτων προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Αλλά δεν είναι ο ίδιος ο κανονισμός που θεσπίζει αυτές τις προτεραιότητες. Και τελευταίο σχόλιο για τροπολογίες που δεν είναι συμβαστικές μεν, υποβλήθηκαν από κάποια μέλη της Επιτροπής Μεταφορών. Μιλούν για την ε, ηχορύπανση από τις σιδηροδρομικές μεταφορές, για το άνοιγμα της αγοράς στον ανταγωνισμό των ε, εθνικών ε, υπηρεσιών μεταφορών επιβατών. Αξιέπαινει αυτή η στόχη, αλλά κατά τη γνώμη μου εκτός θέματος σε σχέση με την πρόταση. Γιατί αλλοιώνουν κάπως διαβρύνουν το περιεχόμενό τους. Προτιμώ να επικεντρωθούμε στις συμβαστικές προτάσεις που στόχο έχουν την προώθηση των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών. Ο Πρόεδρος. Συγγνώμη που σας πίεσα, αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε. Κύριε Ντούχιον, παρακαλώ ένα πολύ σύντομο συμπέρασμα και συγχαρητήρια για το έργο σας. Ευχαριστώ. Απλώς αναφερθώ σε τρία συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα. Θα ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει να υποκύψουμε στον πειρασμό ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε τα πάντα και τους πάντες. Τέτοιος πειρασμού υφίσταται, ξέρετε. Και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επίγνωση αυτού. Και γι' αυτό έδωσε στο χώρο αρκετά στον αρμόδιο φορέα και στο Διοικητικό Συμβούλιο και για να ληφθεί υπόψη και έκανε τα πάντα για να ληφθεί υπόψη και άποψη των κρατών μελών. Και υπάρχουν και οι δυνάμεις της αγοράς που επηρεάζουν τους σιδηροδρόμους. Και από εκεί δίνονται διάφορα κίνητρα μακροπρόθεσμα και επηρεάζουν τα τεκτενόμενα. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό η πρότασή μας να σέβεται το ότι θέλουμε όλοι οι τρόποι μεταφοράς να υπόκεινται στις δυνάμεις αγοράς. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι, και αυτό είναι το τελευταίο μου σχόλιο, ότι όλη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εδώ, ούτω ώστε τελικά κάτι θα μπορέσουμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τη μεταφορά εμπορευμάτων μέσω σιδηροδρόμων, αλλά όχι εις βάρος, δεν θέλουμε να γίνει αυτό, εις βάρος της μεταφοράς των επιβατών. Νομίζω ότι το καταφέραμε αυτό και πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών αυτών και όλου του συνδρομικού δικτύου είναι ο κοινό μα στόχο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, για την συνοπτική σα παρουσίαση. Να ευχαριστήσω καταρχά του διερμηνεί και να του πω ότι είναι ελεύθεροι. Και ευχαριστώ όλου εσά, αγαπητοί συνάδελφοι. Και αύριο το πρωί στι 9 να είστε εδώ, σα παρακαλώ, για μακρά και μακρά και δύσκολη ψηφοφορία για όλη αυτή την έκθεση, αυτέ τι εκθέσει που θα περάσουν τον Απρίλιο από την Ολαομέλεια και θα είναι το τελευταίο μπουκέτο της θητείας αυτής της Επιτροπής Μεταφορών. Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.